Chers collègues, la séance est ouverte. Je vous demande d'abord de noter que le point 14, facilité pour les réfugiés en Turquie, initialement prévu comme. Καλημέρα συνάδελφοι. Το σημείο 14 της ημερήσιας διάταξης θα το εξετάσουμε σήμερα το πρωί προκειμένου η Γενική ε, και Νίρνα μπορέσουν να είναι παρούσες. Το σημείο 4 θα εξεταστεί πρώτο. Σήμερα το απόγευμα θα τελειώσουμε μισή ώρα νωρίτερα. Αμέσως μετά θα γίνει η συνάντηση των συντονιστών και αύριο το πρωί θα έχουμε και πάλι τη ε, συνεδρίαση. Αν δεν υπάρχουν ε, ε, αντιθέσεις θεωρούνται ότι έχουμε ε, εγκρίνει την ημερήσια διάταξη. αν δεν υπάρχουν ε, επίσης αντίθετες απόψεις, θεωρείται ότι έχουν, ε, έχει εγκριθεί η ημερήσια διάταξη της 22 Φεβρουαρίου. Θα ακούσουμε μια παρουσίαση για τη διαχείριση και την εποπτεία των καταπιστευματικών ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα ταμεία αυτά είναι πολύ ε, σημαντικά, ε, παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στον ε, προϋπολογισμό. Έχουν, ε, έχουμε καλέσει για να μας παρουσιάσουν τον κύριο Μουρισάν και την κυρία Κάρδια Ζαμπάλ, η οποία θα λάβει το, ρόλο, το λόγο εξ ονόματος κύριο Γκεγέρ και είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση της υλοποίησης των καταπιστευματικών ταμείων αυτών εξ ονόματος της Επιτροπής Προϋπολογισμών και ο κύριος Καρέρε και ο κύριος Γερεσφερέρ θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους και τις συστάσεις που θεώρησαν απαραίτητες. Ο κύριος Μουρεσάν. Μόλις έφτασα, Πρόεδρε. Δεν, είναι περίεργο που δεν με είδατε. Μόλις σήμερα το πρωί έφτασα. Είναι ένα σημαντικό θέμα νομίζω αυτό το οποίο συζητάμε σήμερα και η χρονική στιγμή είναι και κατάλληλη διότι την περασμένη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζει την ε, συνέχεια του ε, μέσου διευκόλυνσης για την Τουρκία για τους πρόσφυγες και την περασμένη εβδομάδα επιτύχαμε την παράταση. Το πολίτικο έγραψε γι' αυτό. Η... Εμείς το μάθαμε από το πολίτικο, παρότι είμαστε τμήμα της Δημοσιονομικής Αρχής. Παρ' όλα αυτά είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή για να αξιολογήσουμε αυτά τα καταπιστεύματα. Ο κατεπήγον χαρακτήρας των καταπιστευμάτων αυτών πώς ε, συνδέεται με την ακαιρεότητα του προϋπολογισμού και πώς τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου διαφυλάσσονται σε ό,τι αφορά τη λειτουργία αυτών των καταπιστευμάτων. Το πρώτο συμπέρασμα της μελέτης για τις δραστηριότητε των καταπιστευμάτων είναι ότι το Κοινοβούλιο εκπληρεί τις, προϋπο... τις υποχρεώσεις του και ο προϋπολογισμός της Ένωσης το ίδιο σε ό,τι αφορά τις ε, πιστώσεις που δίνονται σε αυτά τα καταπιστεύματα. Όμως τα κράτη-μέλη δεν πληρούν πάντα τις δικές τους υποχρεώσεις. Το δεύτερο το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι αυτή η μελέτη και γι' αυτό σας συνιστώ να την διαβάσετε όλοι σας θερμά, μας δίνει στοιχεία για την εφαρμογή, καθώς και συστάσεις για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη λειτουργία αυτών των ταμείων. Η μελέτη καταλήγει ξεκάθαρα ότι αυτά τα καταπιστευματικά ταμεία αποτελούν κίνδυνο για την ακαιρεότητα του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι οι δημοκρατικές ε, δικλίδες επίσης τίθενται ένα αμφιβόλο. Φυσικά. Αυτό είναι σωστό το συμπέρασμα και μας δίνει, δείχνει ότι ο διακυβερνητικός χαρακτήρας λειτουργίας της Ένωσης δεν είναι καλός όταν υπάρχει Εάν η Ένωση έχει προνόμια σε κάποιους τομείς, σε κάποιες πολιτικές, αυτό που δεν είναι αποδεκτό είναι ότι δεν υπάρχει αρκετή χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της Ένωσης και εφευρίσκουμε τα ταμεία, τα καταπιστεύματα. Επομένω, η λύση είναι σαφή. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρμοδιότητα σε, μία, σε ένα τομέα και περιμένουν η εθνική πολιτική, τα κράτη-μέλη κτλ. Ε, να δώσει, να κάνει κάποια πράγματα. Αν περιμένουμε λοιπόν να κάνει κάποια πράγματα η Ένωση, εφόσον έχει αρμοδιότητε, εφόσον υπάρχουν αυτέ οι προσδοκίε, θα πρέπει να υπάρχουν αρκετοί πόροι στον προπολογισμό τη Ένωση. Το να μην υπάρχει αρκετή προμήθεια, αρκετέ προβλέψει ε, από τον προπολογισμό της, για τον προπολογισμό τη Ένωση και να εφευρίσκουμε τα καταπιστεύματα δεν είναι σωστό. Ποιε είναι οι σωστέ λύσει επαρκής προπολογισμό σε ένα επαρκές επίπεδο με επαρκή ευελιξία και επαρκή περιθώρια για αναπάντηχες περιστάσεις. Οι... Κάποιες από τις εξελίξεις από το 2014 τις περιμέναμε. Όχι, δεν τις περιμέναμε. Θα έχουμε αναπάντηχες εξελίξεις ε, στο επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Προφανώς. Και επομένως, ή θα ξαναϊοθετήσουμε ένα πουδουπού το οποίο ανταποκρίνεται στις ανάγκες μας από Πρώτου του 2021 ή θα έχουμε έναν επαρκή ενα επαρκέ επαρκές πουδουπού από 1η Πρώτου 21 μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2028, 27 συγγνώμη, ή δεν θα έχουμε τον, το επαρκέ πουδουπού και τότε δεν θα μπορούν ε, δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί ε, στις προσδοκίες των πολιτών κτλ. Ή θα μάθουμε από το παρελθόν και θα υιοθετήσουμε ένα επαρκές πουδουπού, επαρκή περιθώρια, επαρκή ευελιξία και αρκετά στεναρό έτσι με επαρκές, ε, επαρκείς ε, πιστώσεις. Επίσης, ο κατεπήγον χαρακτήρας των καταπιστευμάτων. Αν κοιτάξουμε αυτό το μέσο για την Τουρκία. Εκατομμύρια σύρων προσφύγων στην Τουρκία. Αυτό το μέσο, αυτή η διευκόλυνση ήταν σωστή απόφαση. Μας βοήθησε να δώσουμε βοήθεια στους πρόσφυγες στην Τουρκία και να εμποδίσουμε την ε, λαθρομετανάστευση στην Ευρώπη. Ήταν κατεπήγον, ναι ήταν. Εάν κοιτάμε όμως το Ταμείο για την Αφρική, όπου τα κράτη-μέλη δεν πληρούν τις υποχρεώσεις του, όπου ε, ο βαθμός εφαρμογή είναι πολύ χαμηλός, ήταν σωστό να αποφασίσουμε έτσι βιαστικά για αυτό το καταπίστευμα. Όχι. Ήτανε κατεπήγον, όχι. Χρειαζόμαστε μια μακροπρόθεσμη πολιτική για την Αφρική. Χρειάζονται καλέ συνθήκες διαβίωση οι Αφρικανοί. Είμαστε πέρυσι ε, με την Επιτροπή Προπολογισμών στην Αφρική και πήγαμε και ήταν το πρώτο της ε, την Πήγαμε στη Μέση Ανατολή. Ξέρουμε ότι έχουμε υποχρεώσει. Ε, ο προπολογισμό τη Ένωση δίνει λεφτά εκεί και αυτά είναι το κατάλληλο εργαλείο. Φυσικά θα πρέπει να υποστηρίξουμε και την Αφρική, αλλά μέσω του προπολογισμού τη Ένωση. Το καταπίστευμα για την Αφρική δεν ήταν κατεπήγον. Το είπα. Και αν η Κομισιόν θεωρεί ότι ήταν κατεπήγον, τότε πρέπει να πω ότι ήταν αποτυχία, γιατί δεν οδήγησε σε καμία ουσιαστική έλεγχη επιτέλους, ε, επιτόπου. Ε, το Ταμείο για την Τουρκία ήταν κατεπήγον. Αυτό ήταν. Και μας βοήθησε, όπως είπα, να σταματήσουμε τη ροή των λαθρομεταναστών. Των προσφύγων αλλά και των λαθρομεταναστών κυρίως. Το επόμενο σημείο, που είναι το πιο σημαντικό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ενεπλάκει καθόλου στην λήψη των αποφάσεων για τα καταπιστεύματα. Όταν δημιουργήθηκαν, όταν συστήθηκαν αυτά τα καταπιστεύματα, χρειάστηκε να υιοθετήσουμε σχέδια διορθωτικού προϋπολογισμού για αυτά τα, λόγω αυτών των ταμείων. Είναι σαν να φορολογήσει χωρίς να εκπροσωπήσει. Ε, δεν είναι ισορροπημένο, δεν λέμε τίποτα και όμως επηρέασε τον προϋπολογισμό και είχαμε απλώς την ευκαιρία να πούμε ναι. Και μας ε, πίεσαν κιόλα να το πούμε και γρήγορα, σας παρακαλούμε μας λένε, πέστε το γρήγορα γιατί είναι και πολύ επίγον. Φυσικά αυτό δεν θα πρέπει να γίνει το modus vivendi, ο κανόνας που λειτουργούν τα θεσμικά όργανα. Να το πω ξεκάθαρα. Το δικαίωμα της ε, σύμφωνης γνώμης και συμφωνία για τη σύνταξη, για τη σύσταση αυτών των καταπιστευμάτων είναι κάτι που πρέπει να έχει το Κοινοβούλιο. Εάν προκύψει μια κατεπίγουσα ανα, ε, ανάγκη και δημιουργηθεί ένα το καταπίστευμα, εντάξει, σύμφωνοι, να γίνει. Αλλά θα πρέπει να λειτουργήσει, να εμπλακεί το Κοινοβούλιο από την αρχή. Όχι έτσι όπως έγινε με, την με το Ταμείο για την Αφρική. Και ο έλεγχος του Κοινοβουλίου θα πρέπει να υπάρχει βρισκόμαστε στι συνεδριάσει του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά δεν ξέρουμε καθόλου για τίποτα για τη λειτουργική επιτροπή, το Operational Committee. Θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια απέναντι στο Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετέχει και να ενημερώνεται για ό,τι συμβαίνει στι ε, λειτουργικέ αυτέ επιτροπέ σε καθημερινή βάση. Γιατί μιλάμε για τα λεφτά των Ευρωπαίων φορολογουμένων τα οποία ξοδεύονται εκεί. Οι δύο τελευταίε μου παρατηρήσει για να κλείσω και να θέσω βασικά δύο ερωτήσει προς την Επιτροπή ή και προς την Επιτροπή. Θεωρείτε ότι η ένταξη των καταπιστευμάτων αυτών στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το, για το επόμενο πουδουπού υπάρχει τέτοια περίπτωση να συμβεί. Πώς θα εξελιχθούν αυτά τα καταπιστεύματα στο επόμενο πουδουπού. Και η δεύτερη ερώτησή μου είναι ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές αν κοιτάξουμε αυτά τα καταπιστεύματα, από την εμπειρία σας, τι μπορείτε να μας πείτε, τι πήγε καλά, τι θα συνεχίζατε όπως, ε, όπως σήμερα και τι πρέπει να βελτιωθεί κατά τη γνώμη σας Κομισιόν. Δε, δεδομένου του γεγονότος ότι εμείς έχουμε ευθύνη για το προϋπολογισμό, αναγνωρίζετε ότι ο ρόλος του Κοινοβουλίου δεν ήταν ε, επαρκής και ότι τα καταπιστεύματα δεν έδωσαν αυτό που υποσχέθηκαν ότι θα δώσουν. Ποιε είναι οι βέλτιε πρακτικέ από τη διαχείριση, από την εφαρμογή αυτών των καταπιστευμάτων. Θα ήθελα να τα ακούσω αυτά τα πράγματα από την Κομισιόν. Αυτά, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι, ευχαριστώ για την προσοχή, για την προσοχή σας. Περιμένω τη συζήτηση τώρα, με μεγάλο ενδιαφέρον. Ευχαριστώ. Αυτά τα καταπιστεύματα δείχνουν πραγματικά ότι δεν υπάρχει αρκετή ευελιξία στον προπολογισμό μας. Ήρθε εδώ η πρόεδρος της Επιτροπής ΔΕΒΕ, η κυρία Γκάρδια Θαμπάλ. Θα μας κάνει μία συμπληρωματική εισαγωγή μετά από αυτό που ακούσαμε τον κύριο Μουρεσάν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όντως, συμπληρωματικά σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Μουρεσάν. Προφανώς συμφωνώ απόλυτα με την αξιολόγηση που μας έκανε. Όταν άρχισαν να εμφανίζονται όλα αυτά τα εργαλεία τα οποία βρίσκονται εκτός προπολογισμού, αυτό ο γαλαξία από έξω ε, δημοσιονομικά μέσα μας είπαν ότι ήταν για να υλοποιηθούν τρεις στόχοι ή για να λυθούν τρία προβλήματα. Καταρχά, μα είπαν ότι θα πρέπει να δώσουμε μια πάρα πολύ γρήγορη απάντηση σε μια κατεπίγουσα κατάσταση. Δεύτερον, για να έχουμε μεγαλύτερη ε, ταχύτητα στην εφαρμογή αυτών των ε, εργαλείων. Και τρίτον, για να υπάρχουν, να δοθούν επιπλέον λεφτά από τα κράτη-μέλη. Και όμως, τι προκύπτει από αυτή τη μελέτη, ότι αυτοί οι τρεις στόχοι δεν υλοποιήθηκαν. Επομένω, η προστιθέμενη αξία αυτού του πράγματος δεν αποδείχτηκε. Και γι' αυτό ακριβώς ε, δεν υπάρχει και η προστιθέμενη αξία που θα έπρεπε να υπάρχει. Και όχι μόνο δεν υπάρχει, από την μελέτη προκύπτει ότι δημιουργούνται και δύο προβλήματα. Πρώτον, ότι το Κοινοβούλιο αυτό που είπε το Κοινοβούλιο ξεκάθαρα, ότι ως Κοινοβούλιο εμείς πρέπει να ελέγχουμε και να ελέγχουμε κυρίως τι χρηματοδοτείται και τι ε, προγράμματα και τι project προωθούνται μέσω αυτών των καταπιστευμάτων. Δεύτερον, υπάρχει μια πιθανή σύγκρουση συμφερόντων εδώ. Γιατί οι οργανώσεις ή οι οντότητες οι οποίες ε, βρίσκονται ε, και επιλέγουν αυτά τα project βρίσκονται στην μέσα στην όλη διαδικασία και επιλέγουν αυτά τα project, συχνά συμμετέχουν σε αυτά τα project. Σύγκρουση συμφερόντων επομένω. Υπάρχουν και δέκα συμπεράσματα έτσι, που προκύπτουν από την ε, έκθεση αυτή, που αν όντω υλοποιηθούν θα βελτιώσουν πολύ τη διαχείριση αυτών των ε, εργαλείων που βρίσκονται εκτό ε, προπολογισμού. Όπω είπε και ο κ. Μουρεσάν, τι θα κάνουμε στο επόμενο πουδουπού, αν είναι πιο ευρύ αυτό το επόμενο πουδουπού και μπορεί να εντάξει όλα αυτά τα εργαλεία και μάλιστα είναι αρκετά ευέλικτο ούτω ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις κατεπίγουσες καταστάσεις που θα αντιμετωπίσουμε τα επόμενα χρόνια, τότε δεν έχει κανένα νόημα να έχουμε αυτά τα έκτακτα ας πούμε, εργαλεία εκτός προπολογισμού και να αντιμετωπίζουμε όλα αυτά τα προβλήματα που βλέπουμε. Πολύ ωραία. Εμείς αυτά ξέρουμε, περιμένουμε να ακούσουμε και άλλες πληροφορίες. Τα αποτελέσματα της μελέτης δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να επιβεβαιώνουν τις ε, αμφιβολίες και τις κριτικές που είχαμε απέναντι σε αυτά τα καταπιστεύματα. Ευχαριστώ. Merci, Ευχαριστώ κύριε Γκουαρία Θαβάλ. Πολύ ωραία. Πρέπει να κλείσουμε αυτό το σημείο οπωσδήποτε στις 10 η ώρα. Και προτείνω τώρα η παρουσίαση να γίνει μέσα σε 10 λεπτά παρακαλώ. Ξέρω ότι οι εισηγητές μπορούν να κάνουν περιλήψεις πάρα πολύ καλές. Ε, συνεχεία, η Κομισιόν θα έχει 5 λεπτά, ούτω ώστε να έχουμε τελικά ακόμα 15 λεπτά για τη συζήτηση. Πολύ ωραία. Ο κύριος Καρέρα και ο κύριος Νούνες Φερέρ είναι αυτοί που θα πάρουν το λόγο. Ε, ο κύριος Καρέρα και μετά ο κύριος Φερέρ. Ευχαριστώ πολύ τους ευρωβουλευτές, ε, όλους σας. Ε, πραγματικά είναι μεγάλη χαρά για μένα που μου προσφέρετε η ευκαιρία να σας παρουσιάσω την έρευνά μας. Η ε, μελέτη αυτή μας ανατέθηκε από την Γενική Διεύθυνση IPOL. Έχουμε λοιπόν εδώ τους ερευνητές οι οποίοι διεξήγαγαν αυτή την έρευνα. Και σε 10 λεπτά θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε τα βασικά σημεία της μελέτης μας, η οποία είναι ιδιαίτερα εμβριθής και εμπεριστατωμένη. Στόχος μας είναι το θέμα της διαχείρισης, να έχουμε έτσι και μια γενική επισκόπηση των καταπιστευματικών ταμείων, του μηχανισμού για τις πρόσφυγες στην Τουρκία. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι όχι να υπάρξει μια ποιοτική αξιολόγηση των προγραμμάτων, Άρα δηλαδή δεν πρόκειται για μια μελέτη με τη μορφή ελέγχου. Το επίκεντρο της αξιολόγησής μας ε, είναι να εξετάσουμε την προσθέμενη αξία έχοντας κατά νου κυρίως ε, τους, ε, τις συνθήκες και τις διατάξεις για καλή νομοθετική πράξη, για καλή νομοθεσία. Ε, αρμόδια αρχή είναι η Επιτροπή Προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ στην, ε, στον πίνακα αυτό βλέπουμε όλες τις μελέτες, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές αλλαγέ. Έχουμε το μηχανισμό στήριξης για την Τουρκία. Αυτό δεν είναι πιστευματικό ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά το συμπεριλάβαμε στις αναλύσει μας ε, γιατί είναι ένα ειδικό εργαλείο για περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Δεν μπορεί όμως να προσμετρηθεί στα κλασικά ε, καταπιστευματικά ταμεία. Ο δημοσιονομικός κανονισμός προβλέπει τη δυνατότητα να συστήνονται αυτά τα ταμεία, υπό ποιε προποθέσει μπορούν να συστηθούν. Η προστιθέμενη αξία έχει σχέση με εθνικά προγράμματα, εθνικά συμφέροντα, έκτακτες περιπτώσεις. Παίζει ρόλο αν υπάρχει κάποια έκτακτη περίπτωση η οποία να αιτιολογεί την ε, σύσταση του Ταμείου. Αναφέρθηκε το θέμα της προσθέμενης αξίας, αλλά και η ευελιξία, η παρουσία. Το θέμα είναι με ποιο κόστος. Ναι, ευελιξία, σωστά, αλλά με ποιο κόστος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο και βεβαίως και ο ρόλος των κρατών μελών αναφέρθηκε ότι είναι πολύ σημαντικός. Το βασικό ερώτημα που τίθεται στη μελέτη αυτή είναι ο βαθμός στον οποίο αυτά τα ταμεία θεωρούνται το πιο κατάλληλο εργαλείο σε μια συγκεκριμένη περίπτωση. Υπάρχει άραγε πιεστική ανάγκη, υπάρχει έκτακτη ανάγκη. Πώς μπορούμε να αξιολογήσουμε την προσθέμενη αξία. Εδώ λοιπόν το ελεγκτικό συνέδριο παρουσιάζει, έχει μια ε, πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη για το καταπιστευματικό ταμείο Μπεκού, όπου καταλήγει η μελέτη ότι αυτό το ταμείο ήταν το το κατάλληλο. Αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να έχει προσφέρει πιο ουσιαστική ανάλυση των προαπαιτούμενων ε, και κατά πόσον καλύπτονται στην περίπτωση αυτού του Ταμείου του Μπεκού τα προαπαιτούμενα τα καταπιστευματικά ταμεία για την Αφρική αναφέρθηκαν. Υπήρχε άραγε ανάγκη να συσταθούν αυτά τα ταμεία για την Αφρική. Η μετανάστευση από την Αφρική ήταν πολύ μεγάλη ήδη πριν από το 2015. Δεν ξέρω λοιπόν ήταν έκτακτη ανάγκη αφού υπήρχε έτσι και αλλιώ ε, η διαπίστωση. Τα αίτια είναι ένα θέμα που έχει άμεση σχέση με την ανάπτυξη. Είναι ένα θέμα μακροπρόθεσμο. Γι' αυτό αυτό λοιπόν, ε, το κατά πόσον υπήρχε αυτή η έκτακτη ανάγκη, αυτό ε, είναι αμφίβολο. επανερχόμεθα σε θέματα διαχείρισης και λογοδοσίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει καθεστώς παρατηρητή. Ε, όμως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσκαλείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Θεωρούμε ότι μια πολύ καλή πρακτική που πρέπει να συνεχιστεί. Βέβαια, το θέμα, το σημαντικό, παραμένει στις επιχειρησιακές λειτουργικές επιτροπές, οι οποίες αποφασίζουν για τα προγράμματα. Εδώ διαπιστώνουμε κάποια ασάφεια. Δηλαδή, όταν πρόκειται για τα κριτήρια επιλεξιμότητας, ε, είναι μια φαιά ζώνη που ενδεχομένως να αποθαρρύνει κάποιους ετούντες και επίση ε, αναφέρθηκε και προηγουμένω η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στα κράτη-μέλη ως δωρητέ και στα κράτη-μέλη ως ε, μέλη που εφαρμόζουν τα προγράμματα, αυτή η διαχωριστική γραμμή δεν είναι σαφή ενδεχομένω να υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Και υπάρχει και το ερώτημα κατά πόσον ο εταίρο που επιλέγεται είναι πράγματι και ο βέλτιστος για την εφαρμογή ενό κινητούν προγράμματος ή μια δράση. Η μια δραση η εξετάζει και το θέμα τη δημοκρατική λογοδοσία, εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων. Αυτό που μα ενδιαφέρει είναι η συνεχή λογοδοσία σε σχέση με αυτά τα ταμεία, δημοκρατία δημοκρατική λογοδεσία και, το, και ο τρόπος με τον οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να εμπλακεί στην αξιολόγηση των πράξεων. Υπάρχει ένα κενό στον έλεγχο των αποτελεσμάτων, κατά πόσον υπάρχει συμμόρφωση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και με το κράτος δικαίου, ε, κατά πόσον αυτά τα ταμεία ε, δημιουργούν ε, πράγματι προβλήματα στις χώρες που δεν διασφαλίζουν ανθρώπινα δικαιώματα και κράτος δικαίου. Την προηγούμενη εβδομάδα το Ελεγκτικό Συνέδριο κατέθεσε σε μια μελέτη για την Τουρκία και επισήμανε το πόσο δύσκολο είναι λόγω των προβλημάτων επιβολή ε, κράτου δικαίου σε αυτή τη χώρα και δημοκρατική λογοδοσία. Είναι πολύ δύσκολο το ταμείο που έχει συσταθεί για την Τουρκία να ε, επιδιώξει το στόχο του. Δυστυχώ δεν έχουμε χρόνο για να σα παρουσιάσω τα διάφορα ταμεία. Η μελέτη παρουσιάζει πολλέ πληροφορίε όπω ε, το ποιοι εφαρμόζουν τα προγράμματα οι τομείς, ε, τα θέματα που χρηματοδοτούνται από κάθε ταμείο. Ένα από τα βασικά μηνύματα που εκπέμπει η μελέτη είναι ότι τα ταμεία δεν είναι υπαρκτά, δεν υπάρχουν από μόνα τους, αλλά είναι ένα κεντρικό στοιχείο της εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι τα μέσα της εξωτερικής πολιτικής ε, για την ε, μετανάστευση ε, κατ' ουσίαν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με βάση τις συνθήκες θα πρέπει να συμμετέχει στις αποφάσεις. Η μελέτη λοιπόν επισημαίνει ότι αυτός ο, αυτά τα επιπρόσθετα εργαλεία του προϋπολογισμού κατ' ουσίαν ε, αμφισβητούν το ρόλο που προβλέπεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τις συνθήκες. Γιατί, διότι υπάρχει αυτό το στοιχείο της έκτακτης ανάγκης που είναι καθοριστικό για τη σύσταση ταμείων το γεγονός ότι μπορούμε να επενδύσουμε στην ανάπτυξη για να προλάβουμε τη μετανάστευση, αυτή είναι λάθος άποψη. Ε, η μελέτη επισημαίνει επίσης ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο να επιτρέψουμε στην ανάπτυξη, σε συζητήσεις, στην εργασία, ανάπτυξη, να παρισφρήσει μια άποψη που είναι κατ' ουσίαν άποψη των Υπουργείων Εσωτερικών η ανάπτυξη και η συνεργασία για την ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι εις βάρος της μετανάστευσης αλλά κατ' ουσίαν θα πρέπει να εξυπηρετεί τα θεματολόγια των Υπουργείων Εσωτερικών. Η Τουρκία, παραδείγματο χάρη. Εκεί ποια είναι η στρατηγική εξόδου. Εφόσον ή εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση δώσει τόσα δισεκατομμύρια στην Τουρκία, τότε τι θα προσφέρει στην Αφρική. Και πώ θα ξεφύγει από αυτό τον κύκλο η Ευρωπαϊκή Ένωση, από ένα φαύλο κύκλο ε, Προσφορά ε, κονδυλίων χρημάτων, οπότε δεν ξέρουμε πού καταλήγουν αυτά τα κονδύλια και ποια είναι η αποτελεσματικότητά του, ποια είναι η προστιθέμενη αξία που προσφέρουν. Περνάμε στι συστάσεις. Πράγματι ε, είναι ένα νομοθετικό εργαλείο, αλλά ο διαμεσολαβητή λέει ότι όσον αφορά την Τουρκία, ανεξάρτητα από τη φύση του μέσου, του εργαλείου, αν είναι πολιτικό ή χρηματοδοτικό, παρόλα αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να ελέγχει εντελεχώς ε, τις επιπτώσεις ε, αυτών των ταμείων. Να γίνει ταξιολόγηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να εντοπίζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι σε μια συγκεκριμένη χώρα Επίσης, ε, θέσαμε το θέμα των ε, συντακτικών ε, συμφωνιών. Η μελέτη επισημαίνει ότι υπάρχουν κάποιες ελπιδοφόρες πρακτικές το Ταμείο του Χάρη Μαδάτη για τη Συρία είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα, θετικό παράδειγμα για το πώς μπορούν να συνταχτούν οι συντακτικές συμφωνίες, συστατικές μάλλον συμφωνίες που θα μπορούσαν να αποτελέσουν πηγή έμπνευση για τα καταπιστευματικά ταμεία. Τώρα, όσον αφορά τη συνεργασία με, τη, με τα κράτη-μέλη. Πάλι αυτό το Ταμείο για την κρίση τη Συρίας είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα. Δεν πρέπει να είναι αυτό η προτεραιότητά μας, γιατί κατ' ουσίαν αυτά στην πράξη σημαίνουν ότι ε, συγκεκριμένα συμφέροντα συγκεκριμένων κρατών μελών κυριαρχούν μάλιστα εις βάρος άλλων αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί να υπάρχει προτεραιότητα για τέτοια μορφή ή ε, εξουσιοδότηση, να εκχωρούμε για εκχώρηση της συνεργασίας. Παραδείγματο χάρη στο καταπιστευματικό ταμείο για την Αφρική κάναμε μία μελέτη για την Αιθιοπία και τι είδαμε, και είδαμε μία μελέτη που τη χειρίζεται κατ' ουσίαν η Ιταλία η οποία έχει στόχο να περιορίσει τη μετανάστευση ή αν θέλετε ε, αυτό το καταψευματικό ταμείο για την Κολυμπία συμφέρει, είναι προς όφελος ε, της ε, Ισπανίας. Όμως υπάρχει και ενωσιακή αξία και αυτή θα πρέπει να προβληθεί να υπάρχει μεγαλύτερη δημοκρατική λογοδοσία. Ένα ισχυρότερο πλαίσιο που θα καθορίζει το ποιε πρέπει να είναι επιπτώσει επιτόπου και με τον τρόπο αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη θα μπορούν να εντάσσονται καλύτερα στα προγράμματα αυτά, να μην έχουμε δηλαδή στο τέλος ε, πόρους που εκταμιεύονται και είναι αντίθετοι με τους στόχους του Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τελευταία τώρα διαφάνεια. Ζητάμε την συνεχιζόμενη και εκ των υστέρων αξιολόγηση των ταμείων, ε, των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων, του κράτου δικαίου. Είναι πολύ απαραίτητο κάθε ταμείο να προσαρμόζεται σε αυτά τα θέματα, στους κινδύνους και στους, ε, στην πραγματικότητα που επικρατεί σε κάθε περίπτωση. Βλέπουμε ότι κάποια κονδύλια που διοχετεύονται για ή σε κυβερνήσεις, τα κονδύλια αυτά κατ' ουσίαν ενέχουν ε, σε υφέρπουσα μορφή και τον κίνδυνο να υπονομευτεί το κράτος δικαίου. Ε, υπάρχουν παραδείγματα στα Ηνωμένα Έθνη και στην Παγκόσμια Τράπεζα και εκεί ε, είδαμε ότι θα μπορούσε να υπάρχει ένα μια ενιαία πύλη και σε εμά στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα ταμεία, γιατί υπάρχει στα Ηνωμένα Έθνη, παραδείγματος χάρη. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φερέρ δεν χρειάζεται να μιλήσει, έχει παραιτηθεί από το δικαίωμα λόγου. Μάλλον ναι. Πολύ ωραία. Η άλλη πλευρά τώρα, η οποία θα επρασπιστεί τη θέση της. Ο κατηγορούμενος έχει το λόγο, η Κομισιόν δηλαδή. Ευχαριστούμε Πρόεδρε. Έχετε πέντε λεφτά, ε, όχι παραπάνω. Είναι άδικο, γιατί ε, αυτοί που μας κατηγορούσαν είχαν δέκα λεφτά. Εγώ ε, είμαι πρόεδρος ε, στην Επιτροπή ε, Μαντάτ για την Αφρική, Συρία και στη Λειτουργική Επιτροπή για την Αφρική. Λοιπόν, δεν θεωρώ ότι αυτά που μας περιγράψαν ήταν ακριβή. Πιστεύω ότι τα καταπιστεύματα δημιουργήθηκαν ως μέσα για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Βοήθειας το 2012 μέσω του δημοσιονομικού κανονισμού μέσα σε πλαίσιο νομιμότητας και είναι η καλύτερη εφεύρεση ίσως που έχει υπάρξει την πρόσφατη ιστορία της ε, οικονομικής αρχιτεκτονικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά τίποτα δεν είναι τέλειο και νομίζω ότι η έκθεση προφανώς τονίζει ορισμένα πολύ σημαντικά πράγματα. Ε, είμαστε έτοιμοι να τα δεχτούμε. Και επίση τα τέσσερα καταπιστεύματα τα οποία υπάρχουν μέχρι στιγμή και πολύ σωστά είπατε ότι ε, ο μηχανισμό ε, για του πρόσφυγε για την Τουρκία ε, είναι ένα μηχανισμό συντονισμού, δεν είναι καταπίστευμα. Α το συζητήσουμε χωριστά. Αλλά τα υπόλοιπα τέσσερα δημιουργήθηκαν με διαφορετικά σενάρια και διαφορετικέ συνθήκε, ακόμα και πολιτικέ, διαφορετικέ πολιτικέ συνθήκε. Επομένω, νομίζω ότι θα πρέπει να διδαχτούμε και θα πρέπει να κοιτάξουμε ποιε είναι οι βαλτέ πρακτικέ. Όμω, πιστεύω ότι όντως υπάρχει κατεπίγουσα ανάγκη. Όταν δύο... Ε, στο, όταν στο Λίβανο, στην Τουρκία, ε, ζουν δύο εκατομμύρια στα στρατόπεδα, όταν ένα εκατομμύριο άτομα φεύγουν από τη Συρία, από την Λιβύη, συγγνώμη, για να έρθουν στις ε, όχθες της Ευρώπης και νομίζω ότι τα καταπιστεύματα ήταν πολύ γρήγορα στη λειτουργία τους για να αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματα. Φυσικά θα πρέπει να δούμε πώς γίνεται αυτό. Και η έκθεση πολύ σωστά τονίζει δύο βασικά θέματα. Πρώτον, είναι ο ποιοτικό έλεγχος. Φυσικά, ποτέ δεν υπάρχει αρκετός ποιοτικό έλεγχος των αποτελεσμάτων και αρκετή πρόβλεψη ε, εκ των προτέρων και εκ των υστέρων έλεγχος, ας πούμε. Παρ' όλα αυτά, εφαρμόσουμε το ίδιο σύστημα ποιοτικού ελέγχου και αξιολόγηση και παρακολούθηση ε, που θα χρησιμοποιούσαμε σε οποιοδήποτε άλλο ευρωπαϊκό project το οποίο ε, χρηματοδοτείται από τον προπολογισμό ή από το Ευρωπαϊκό Ταμείο ανάπτυξη. Και αν χρειάζεται απόδειξη για του λόγου του αληθέ, να σα πω ότι για το καταπίστευμα μαντάτ, ναι, μόνο φέτο έχουμε ε, τρεις μελέτες συγγνώμη, τρία project τα οποία χρηματοδοτούνται. Πήγατε στον, στην Ιορδανία και είδατε κάποια από αυτά τα project ε, με, τα ίδια σα τα μάτια. Βλέπετε τι γίνεται και εσεί ε, πήγατε και η Κοντ και η Άφετ και είδατε κάποια project στην Μέση Ανατολή και στην Αφρική. Και έχετε πιστεί, πιστεύω, από τις επιδόσεις ε, και αποτελέσματα των project. Φυσικά Είμαστε προσανατολισμένοι στα αποτελέσματα, όπως και οτιδήποτε άλλο χρηματοδοτούμε εξωτερικά. Ε, και πιστεύω ότι σε ό,τι αφορά τον ποιοτικό έλεγχο, το σύστημα υπάρχει. Φυσικά το σύστημα χρήση βελτίωσης. Αλλά αν θέλετε να βελτιώσουμε το, το σύστημα, θα πρέπει να το ε, βελτιώσουμε συνολικά, όχι μόνο για τα καταπιστεύματα. Επίσης, η συμμετοχή του Κοινοβουλίου και ο έλεγχος του Κοινοβουλίου. Τα καταπιστεύματα αποτελούνται από τι εισφορέ από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη, τον νοσιακό προπολογισμό λοιπόν, και μια τρίτη συνεισφορά από ε, την, ε, τις των κρατών μελών και τρίτων χωρών, Νορβηγία, Τουρκία κτλ. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, για την περίπτωση του Μαντάτ αποφασίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση τις ίδιε διαδικασίε με οποιοδήποτε άλλο project που χρηματοδοτούμε, όπω παραδείγματο χάρη τη διαδικασία επιτροπολογία με πλήρη κοινοβουλευτικό έλεγχο, όπως για οποιοδήποτε άλλο project. Εν συνεχεία, σε ό,τι αφορά τα ίδια τα καταπιστεύματα, φυσικά είμαστε έτοιμοι να εμπλέξουμε το Κοινοβούλιο ακόμα περισσότερο. Υπάρχει συμφωνία ότι τα μέλη του Κοινοβουλίου συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο των Καταπιστευμάτων και εγώ προσωπικά, αν μου επιτρέψετε την παρατήρηση, θα ήθελα αυτή η συμμετοχή να ήταν πιο έτσι, ενεργή. Δεύτερον, συμφωνήσαμε ότι στο νέο δημοσιονομικό κανονισμό θα υπάρχει μία έγκριση του Κοινοβουλίου πριν από τη δημιουργία νέων θεματικών ε, καταπιστευμάτων και θα υπάρχει και πρώτερη διαβούλευση με το Κοινοβούλιο πριν από τη δημιουργία ε, καταπιστευμάτων κατεπήγοντος και για καταστάσεις αφού λήξει η κατεπήγουσα ανάγκη. Επομένως υπάρχει συμμετοχή του Κοινοβουλίου. Αλλά ούτω ή άλλω έχουμε έρθει σε επαφή τον Ιούνιο του 2017, εκ των προτέρων δηλαδή. Ε, μια ερωτική σύνοδο είχαμε για το καταπίστευμα Μαντάπ για τη Συρία. Και είχαμε αντιπροσωπείε που πήγαν και είδαν το project. Επίση, σα ενημερώσαμε για τη Βόρεια Αφρική, ε, για το αφρικανικό καταπιστεύμα, στην Επιτροπή Πέτη, στην Επιτροπή Ντέβε, στην Επιτροπή Λίπε το 2017. Επομένω, νομίζω δεν μπορείτε να μα κατηγορείτε ότι δεν ε, δεχόμαστε τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Ακόμα ένα λεπτό, Πρόεδρε, να πω και κάτι άλλο. Υπάρχουν δύο επιχειρήματα τα οποία ε, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικά. Καταρχά, επί χρόνια, ατελείωτα χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτούσε ε, καταπιστεύματα της, ε, του ΟΗΕ και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Αυτό σημαίνει κόστος. Κοιτάξτε, τα, τα, τις λειτουργικές δαπάνες. Δεν υπήρχε καμία, κανένας έλεγχος από εμά και δεν μπορούσαμε να επηρεάσουμε τα project και ότι κάνουν αυτά τα project. Πιστεύω λοιπόν ότι τα ευρωπαϊκά καταπιστεύματα, όσο ατελεί και να είναι, μας δίνουν μεγαλύτερες εγγύσεις. Και νομίζω ότι η προτίμηση που έχετε ε, για ε, χωρισμένη συνεργασία ε, υπάρχει για να ενισχύσει την ε, διαφάνεια. Γιατί οι δικές μας υπηρεσίες όχι μόνο είναι παρούσες και ξέρουν, αλλά είναι οργανισμοί και υπηρεσίες που είναι πιο ανοιχτές για... και πιο διαφανείς ας πούμε, από, τις, από τους οργανισμούς του ΟΗΕ κτλ. Δεύτερον, ε, συμφωνώ με τον εισηγητή που λέει ότι καλύτερο θα ήταν να δώσουμε επαρκή χρηματοδότηση στον τίτλο 4. Καλύτερα θα ήταν να ενσωματώσουμε τα λεφτά αυτά στο που Και ελπίζω να σα ακούσουν από το 2021 και μετά. Αλλά προ το παρόν δυστυχώ δεν σα ακούν τα κράτη-μέλη. Και προ το παρόν δεν έχουμε μηχανισμού οι οποίοι να εξυπηρετούν ως πλατφόρμα συντονισμού ανάμεσα σε αυτά που κάνουν τα κράτη-μέλη ε, με τη διμερή τους ε, βοήθεια και αυτό που κάνουν τα καταπιστεύματα. Ε, ας πούμε ένα κράτος μέλος το οποίο δίνει 10 εκατομμύρια ε, σε ένα καταπίστευμα ε, θέλει πολύ περισσότερο να συντονίσει εκείνο ας πούμε ε, τη δική του βοήθεια για την Αφρική, παραδείγματο χάρη, παρά να το κάνει μέσω ενό καταπιστεύματο. Και τέλο, έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο έχει να κάνει με, το γεωγραφ... με τη γεωγραφική πτυχή των προγραμμάτων και της χρηματοδότησης. Θα θυμάστε όταν το κουμπάνε κοντά στα σύνορα ε, Τουρκίας-Συρίας. Ε, ήταν υπό ε, την πολιορκία του Ντάεσ. Και 200.000 άτομα από εκεί πήγανε προς τα τουρκικά σύνορα. Προς τις τουρκικές αρχές. Και το... Αποδείχθηκε ότι το χρηματοδοτικό σύστημα δεν ήταν αρκετά ευέλικτο. Γιατί εμεί, α πούμε, ε, ε, η Συρία, ο Λίβανος κτλ. εποφελούνταν. Η Τουρκία υποφελείται από το πρωταξιακό εργαλείο. Ε, οι άλλες τρεις χώρες, η, η Ορδανία κτλ, ε, από την αναπτυξιακή βοήθεια. Αλλά όλα αυτά τα μέσα μαζί δεν μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες των 200.000 ανθρώπων. Με το καταπίστευμα το οποίο ε, φτιάξαμε τώρα έχουμε ένα ευέλικτο εργαλείο το οποίο μπορεί να αντιμετωπίσει, τελευταία είναι αυτά που λέω, τις ανάγκες των ε, προσφύγων και μεταναστών σε κατεπίγουσες ανάγκες όπου ε, υπάρχει πρόβλημα. Παραδείγματο χάρη η κρίση στη Συρία. Χρηματοδοτούμε λοιπόν project όχι μόνο στον Ιράν, στο Λίβανο, στη Συρία, αλλά στην Αρμενία, Σερβία, όπου υπάρχουν ε, Σύριοι πρόσφυγε. Είναι η ευελιξία που έχουμε. Και δουλεύω ε, εδώ 24 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν ξέρω κανέναν άλλο μηχανισμό ο οποίο μπορεί να παρέμβει τόσο γρήγορα, τόσο ευέλικτα και τόσο αποτελεσματικά όσο αυτό ο μηχανισμό. Πιστέψτε με, ε, είναι επιλόγω τιμή το λέω. Ευχαριστώ και τώρα θα δώσουμε το λόγο στους συναδέλφους που θέλουν να πάρουν το λόγο. Παρακαλώ, λακωνικά όμως. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό και κάτι. Ποιος θέλει να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κατά τη γνώμη μου, η αλήθεια είναι ότι τα καταπιστεύματα ιδρύθηκαν για διαφορετικούς λόγους σε κάθε μέρος, σε διαφορετικές στιγμές και έχουν καταλήξει να γίνει μια συνήθεια. Και το πρόβλημα είναι η ευελιξία, όπως υπόθηκε. Και αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας ε, όταν ε, συστήνουμε νέα καταπιστεύματα. Όταν κοιτάμε το καταπίστευμα για την ε, Αφρική, το θέμα ήταν η ορατότητα για τους ε, υπουργού στο Συμβούλιο ή το καταπίστευμα για τη Τουρκία. Ήταν αποτέλεσμα μιας πολιτικής απόφασης. Ήταν... Ήμουν στη Τουρκία εκείνη την εβδομάδα, μίλησα με διάφορους πολιτικούς. Ε, είχαν πρόβλημα με όλη αυτή τη ροή ε, προσφύγων και ή θέλανε να πληρώσουμε γι' αυτό. Το αν ήταν σωστή απόφαση ήταν το κάτι άλλο. Κάτι έπρεπε να κάνουμε πάντως. Και το αποτέλεσμα ήταν η ίδρυση του ε, Ταμείου. Το Ταμείο Μπέκου ε, γύρισε από την Αφρική πριν από λίγες εβδομάδες. Αυτό το ε, Ταμείο είναι ακριβώς ε, το είδος Ταμείου που θα έπρεπε να συσταθεί σε κατάσταση έκτατης ανάγκης όταν το κράτος δεν ε, μπορεί να ε, παράγει αποτελέσματα. Ήμουν εκεί στην ε, ε, Λαϊκή Δημοκρατία της, Αφρικής, της Κεντρικής Αφρικής και ένα από τα προβλήματα των ταμείων είναι ότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα για πολύ μικρά project. Ε, Μίλησα με εκπροσώπους ε, ΜΚΟ και τους ρώτησα πώς ε, χρηματοδοτούνται. Και αποδεικνύεται ότι δίνουμε χρήματα σε ε, οργανισμούς που έχουν εποπτικό ρόλο, αλλά όχι σε μικρούς οργανισμούς. Πρέπει λοιπόν να το έχουμε υπόψη μας αυτό. Στην Κεντρική Αφρική πρέπει να έχουμε υπόψη μας και να λαμβάνουμε υπόψη μας το ε, ρίσκο. Σε ό,τι αφορά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, αν η Κομισιόν είναι ε, απογοητευμένη με τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου, θα πω ότι μου ζητήθηκε να πάω στο Μπαγκή, το Μπέκου, ε, με πέντε μέρες μόνο προειδοποίηση. Ξέρω ότι η Κομισιόν είχε προβλέψει αυτή την συνεδρίαση τη συνάντηση πολύ πριν. Γιατί ειδοποιήθηκα τελευταία στιγμή. Σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη, είναι και αυτό ένα θέμα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας για να αλλάξουν τα πράγματα στο μέλλον. Κατά τη γνώμη μου, σε κάποιες περιπτώσεις, ναι, χρειάζονται καταπιστεύματα. Το αν χρειαζόμασταν ένα καταπίστευμα για την Αφρική για να αντιμετωπίσουμε το θέμα της μετανάστασης, δεν είμαι σίγουρη. Αυτό σημαίνει ότι παίρνουμε χρήματα από τα project για την ανάπτυξη και τα χρησιμοποιούμε αλλού. Σε ό,τι αφορά τα νέα ταμεία, λοιπόν, πρέπει να είμαστε αυστηροί, να ξέρουμε πού διαθέτουμε τα χρήματα, να υπάρχει ορατότητα, έλεγχο και να διασφαλίσουμε την απαραίτητη ευελιξία για να έχουμε και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ο κύριος Κολμέλη έχει το λόγο. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να πω κάποια θέματα που είναι θέματα αρχής. Κοιτάξτε, σε αυτή την Επιτροπή πολύ συχνά συζητάμε για την απαραίτητη διαφάνεια που πρέπει να χαρακτηρίζει κυρίως τον προϋπολογισμό. Είμαστε λοιπόν αναγκασμένοι να δεχτούμε ότι αυτά τα καταπιστευματικά ταμεία δεν συμβάλλουν σε μεγαλύτερη διαφάνεια. Συμβαίνει το αντίθετο. Και το δεύτερο που πολλοί το είπαν είναι ότι αυτά τα ταμεία είναι πολύ σημαντικά έτσι ώστε να μπορούμε να αντιδράσουμε γρήγορα και σωστά. Δείτε λοιπόν το ερώτημα κατά πόσον ο προϋπολογισμός μας είναι συντεταγμένος με τέτοιο τρόπο ώστε να πληρεί αυτές τις προποθέσεις. Φοβάμαι πως όχι. Άρα πρέπει να σκεφτούμε το τι πρέπει να αλλάξουμε στον προϋπολογισμό έτσι με βάση τον προϋπολογισμό να μπορούμε να αντιδράσουμε σωστά και γρήγορα. Το δεύτερο ισχύει το εξή ότι σε ειδικέ περιπτώσεις, σε έκτακτε περιπτώσει, πράγματι πρέπει να χορηγούμε βοήθεια, αυτό δεν συζητιέται. Νομίζω όμως ότι μερικές φορές η βοήθεια αυτή καθίσταται απαραίτητη. Ξέρετε γιατί. Γιατί μας δείπει η απαραίτητη στρατηγική για να μπορέσουμε έγκαιρα να εντοπίσουμε τα προβλήματα. Αν κανείς εντόπιζε έγκαιρα τα προβλήματα, τότε δεν θα προέκυπταν πολλές έκτακτες καταστάσεις. Ως εκ τούτου, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να μεριμνήσουμε έτσι ώστε ειδικά στον τομέα και στα προβλήματα που έχουν σχέση με τη μετανάστευση να επεξεργαστούμε μία μακροπνοή και μακροχρόνια στρατηγική η οποία δυστυχώς εξακολουθεί να λείπει. Ευχαριστώ πολύ. Uh, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κατά τη γνώμη μου είναι προφανές ότι όποιο και αν είναι ο προπολογισμό που υιοθετούμε, όποιο μηχανισμό επιλέγουμε, ποτέ δεν θα μπορούμε να προβλέψουμε ε, όλες τις ε, περιστάσεις που θα προκύψουν. Είναι λοιπόν χρήσιμο να Υπάρχουν ευέλικτα εργαλεία που επιτρέπουν να αντιμετωπίσουν έκτακτες ανάγκες που ποτέ δεν μπορούν να ε, προβλεφθούν στο 100%. Όταν υπάρχει ε, ελληματική λογοδοσία και βλέπω το πίνακα στη σελίδα 45 του εγγράφου ε, δείχνει ξεκάθαρα την απουσία του κοινοβουλευτικού ελέγχου στην όλη διαδικασία αυτό μας καθιστά ευάλωτους, καθιστά την Κομισιόν ευάλωτη. Σε ε, περιστάσεις που θα προκύψουν καταχρήσεις, γιατί όπου υπάρχει χρήμα και εξουσία υπάρχουν καταχρήσεις. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα, να αντιμετωπίσουμε την έλλειψη ε, δημοκρατικής λογοδοσίας, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι τα κονδύλια που χρειάζονται για έκτακτες ανάγκες είναι όντως αποτελεσματικά και δεν, είναι, δεν συμμετέχουν απλώς σε ένα μηχανισμό που προσπαθούν να υπονομεύσουν τους θεσμούς που προσπαθούμε να συστήσουμε. Είναι απαραίτητος ο δημοκρατικός είναι, εύκολο, είναι δύσκολο, αλλά είναι απαραίτητο ε, μακροπρόθεσμα. Ευχαριστώ πολύ. Πράγματι, βλέπουμε ότι με αυτά τα ταμεία προσπαθούμε να καλύψουμε το κενό, την απουσία ε, ευελιξίας. Και το παράδοξο είναι ότι η ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υλοποιήσει πρακτική πολιτικές που δεν τηρούν τους βασικούς δημοσιονομικούς κανόνες. Οι δημοσιονομικές κανόνες για τη Τουρκία θα εμφανιστούν ε, στον προϋπολογισμό, δεν πρόκειται για καταπίστευμα, αλλά θα χρησιμοποιήσουμε τα κονδύλια. Τρία δισεκατομμύρια οι δαπάνε, αλλά θα εμφανιστούν στον προπολογισμό μόνο ένα ε, δισεκατομμύριο. Πιστεύω λοιπόν ότι υπάρχει κενό εδώ, δεν υπάρχει διαφάνεια και σε ό,τι αφορά τα καταπιστεύματα, πιστεύω ότι όταν συστήνεται τέτοιο ταμείο αυτό επιτρέπει στους πολιτικούς να δείχνουν ότι κάνουν κάτι, κάνουν κάτι για την Αφρική. Πολύ καλό αυτό για τις συνεντεύξεις τύπου, τις επίσημες ανακοινώσεις, αλλά στην πράξη δεν υπάρχει απαραίτητη αποτελεσματικότητα. Και ο προϋπολογισμός θα μας επιτρέπει να ε, αντιμετωπίσουμε αυτές τις έκτακτες ανάγκες. Μιλήσατε για τα κονδύλια που δίνουν η Νορβηγία και η, ε, η Ελβετία. Πολύ σημαντικά ποσά που δεν εμφανίζονται όμως στον προϋπολογισμό διατίθενται απευθείας σε ε, κάποιες χώρες που επωφελούνται από την πολιτική συνοχής. Τι συμβαίνει με τα καταπιστεύματα. Για μία ακόμη φορά δεν υπάρχει διαφάνεια. Όταν προσπαθούμε να εξηγήσουμε ότι το Brexit θα μπορούσε να οδηγήσει στην απώλεια 14 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά ε, η το οποίο θα αντισταθμιστεί από τα κονδύλια της Νορβηγίας και της Ελβετίας. Αυτό δεν εμφανίζεται πουθενά όμως. Γιατί υπάρχουν ειδικά συγκεκριμένα κανάλια που ε, έχουν ως αποτέλεσμα αυτά τα κονδύλια να οδηγούνται σε συγκεκριμένες χώρες και δεν εμφανίζονται αυτά τα κονδύλια στον περιπολογισμό. Θα μπορούσατε να μας το εξηγήσετε αυτό. Και ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, ο κύριος Φιλιμπερτό, ήθελε να πάρει το λόγο για πολύ λίγο χρόνο δυστυχώς. Ναι, θα είμαι σύντομο. Θα σε δύο σημεία τα οποία αναφέρθηκαν στη συζήτηση. Καταρχήν, τη χρήση των κονδυλίων για την ανάπτυξη για άλλους πολιτικούς στόχους όμως. Θα ήθελα από τη μία να σας πω ότι είμαστε υποχρεωμένοι με βάση το άρθρο 21 της συνθήκης να εξασφαλίσουμε τη συνέπεια της εξωτερικής δράσης Δηλαδή η συνεισφορά των διαφόρων πολιτικών στην ανάπτυξη και άλλων ε, με συνεπή τρόπο, υπ' αυτή, την, αυτή την έννοια πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι που το καταπιστευματικό ταμείο συνεισφέρει σε μια πιο συνολική δράση Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τις ε, χώρες εταίρους, ειδικά σε περιπτώσεις κρίσης. Όμως, απ' την άλλη, φυσικά δεν είναι οι στόχοι των Υπουργείων Εσωτερικών που πρέπει να εξυπηρετηθούν εδώ. Ε, το Ταμείο για την Αφρική προστατεύει τους ε, πρόσφυγες, τις μεταναστευτικές ροές, την ασφάλεια των συνόρων που το ζητούν και οι χώρες εταίροι. Γιατί οι πρώτες είναι αυτές που πλήττονται από τις ε, ροές μεταναστών προσφύγων συγγνώμη, και μεταναστών μέσα από τα σύνορα. Η επανένταξη των μεταναστών, η στήριξη σε δραστηριότητες που παράγουν εισόδημα, όλες αυτές είναι αναπτυξιακές δράσεις και δεν νομίζω ότι μπορούμε να θεωρήσουμε ότι σφετεριζόμαστε κονδύλια και τα πήγαινουμε αλλού. Ένα άλλο που μας κατηγορήσανε είναι η σύγκρουση συμφερόντων. Νομίζω ότι έχει νόημα να δράμε ενιαίο τρόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη όταν προσφέρει μία σειρά εργαλείων που είναι αναπτυξιακά, εμπορίου, ε, τεχνικής βοήθειας, capacity building, οικοδόμηση δυναμικού προ τρίτε χώρε, ούτω ώστε να συνεργαστούμε με τις τρίτε χώρε. Είναι σημαντικός αυτός ο στόχος στην στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωση σε ό,τι αφορά το εξωτερικό. Ευχαριστώ. Είμαστε υποχρεωμένοι να κλείσουμε εδώ και να περάσουμε στο επόμενο σημείο, τουλάχιστον αυτό που θα ήθελα να πω στους διάφορους ενδιαφερόμενους είναι ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να μπορέσουμε να πούμε τι δράση κάνει η Ευρώπη απέναντι στις μεταναστευτικές ροές. Δεν μπορούμε να πούμε ότι μέσα από αυτά τα ταμεία, τα καταπιστεύματα δηλαδή, ε, ότι δεν υπάρχει εξυπνάδα εκεί σίγουρα, αλλά δεν είναι βανάγνωστα αυτά τα ταμεία, ας πούμε. Δεν τα καταλαβαίνουμε. Όταν γίνεται μια συζήτηση ή όταν ας πούμε ε, γίνουν του χρόνου οι εκλογές. Θα πρέπει να πούμε κάποια επιχειρήματα, θα πρέπει να δείξουμε ξεκάθαρα τι κάνουμε. Ας πούμε το, το καταπίστευμα για την Αφρική. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Έχουμε διάφορες δράσεις για να προσπαθήσουμε να κλείσουμε ας πούμε τους κρουνούς της μετανάστευσης. Αλλά ε, όλα αυτά δεν φαίνονται προς τα έξω. Υπάρχει μια ανάγκη διαφάνειας εδώ και μια ανάγκη, ανάγκη δημοκρατικής νομιμότητας. Γιατί κάθε φορά ε, επιλέγουμε, ε, ε, εφευρίσκουμε ένα steering board, ένα, μια κατευθύνουσα ας πούμε επιτροπή κτλ. Όπου είναι παρούσες όλες οι χώρες, όλες οι, πρε, οι πρεσβείες κτλ. Δεν νομίζω όμως ότι είναι τόσο μεγάλη προσθέμενη αξία αυτού του steering board. Ευχαριστώ λοιπόν τους δύο εμπειρογνώμονες, δεν θα πούμε τίποτα άλλο. Μας είπαν πολλά με την ανάλυση τους και τις συστάσεις τους. Ε, αυτό που είναι καλό είναι ότι έχουμε τη δυνατότητα να βελτιωθούμε, να βελτιωθούμε, να βελτιώσουμε τα πράγματα. Θα πάμε τώρα στο μηχανισμό ε, για την Τουρκία. Έτσι. Θα μιλήσουμε τώρα για αυτό το θέμα θα θυμάται ο Γενικό Συγητή τι συζητήσει που είχαμε ε, στη συνδιαλλαγή για τον προπολογισμό, όπου διρωτώμεθα αν αυτό ο μηχανισμό δεν θα έπρεπε να υπάρχει στο σχέδιο προπολογισμού το 2018. Το θυμάστε, μα είπαν όχι. Όχι, δεν χρειάζεται. Και δυόμισι μήνε μετά, μετά από την αρχή του έτου 2018, ορίστε που βρισκόμαστε. Η Κομισιόν την περασμένη εβδομάδα πρότεινε να παρατείνουμε το μηχανισμό για την Τουρκία, ε, να δώσουμε 3 δισεκατομμύρια ακόμα για το 18 για το 18-19, όπως κάναμε για το 16-17. Η χρηματοδότηση θα γίνει το ίδιο τρόπο, δηλαδή 1 δισεκατομμύριο από τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση και 2 δισεκατομμύρια από τα κράτη-μέλη. Θα προσθέσουμε και την Νορβηγία και την Ελβετία προφανώ εδώ. Η Κομισιόν υιοθέτησε μια απόφαση για αυτό το θέμα και λυπόμαστε που δεν ε, μα διαβουλευτήκατε, αυτό που σα έλεγε ο κ. Μουρισάν πριν από λίγο, ή τουλάχιστον ενημερωθούμε έστω για το πώς η Κομισιόν σκόπευε να τροφοδοτήσει αυτό το 1 δισεκατομμύριο, ή μάλλον να πάρει αυτό το 1 δισεκατομμύριο από τον προπολογισμό. Πού θα το έπαιρνε. Θα έπρεπε να κάνουμε ένα διάλογο, τόσο ώστε οι απόψει του Κοινοβουλίου να, μπορούν, να μπορέσουν να ενσωματωθούν πριν ληφθεί τελική απόφαση. Χωρίς να πάρουμε απόφαση, χωρίς ε, ε, τη σύμφωνη γνώμη, ενώ είμαστε ο ένας από τους δύο βραχίονες ε, του δημοσιονομικού. Είμαστε η, ε, η μία από τις δύο δημοσιονομικές αρχές ε, δίνω το λόγο στον εκπρόσωπο της ε, Κομισιόν, υπεύθυνη για το θέμα αυτό. Πολύ ωραία. Θα παρουσιάσω με μεγάλες λεπτομέρειες την πρόταση αυτή για την παράταση του μηχανισμού για την Τουρκία, του μηχανισμού για τους πρόσφυγες δηλαδή για την Τουρκία. Να σας πω καταρχήν ότι ε, ο Επίτροπος Έτιγκερ στην παρουσίαση που έγινε ε, και στην συζήτηση για, το επόμενο πολιτεύσιμο πολιτεσμό-συνομικό ε, πλαίσιο στο Κοινοβούλιο ήταν ο πρώτος ο οποίος ανήγγειλε την απόφαση της Κομισιόν και το Κοινοβούλιο ενημερώθηκε. Δηλαδή την ίδια μέρα, για να μην σας πω και νωρίτερα, από το Συμβούλιο. Ναι, νομίζω ότι το Συμβούλιο ε, ενημερώθηκε την επόμενη μέρα στο Κορεπέρ. Νομίζω λοιπόν ο Επίτροπο έδειξε τη σημασία που δίδεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αναγγέλλοντα την απόφαση τη Κομισιόν αμέσω μετά την ε, συνεδρίαση του Σώματο ε, των Επιτρόπων στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου. Και τώρα θα πάω στα αγγλικά. Ο μηχανισμό αυτό για την Τουρκία ήταν ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο εκτός της Ευρώπης για τους πρόσφυγες. Αυτό λοιπόν επιβεβαιώνεται από τη δεύτερη έκθεση για το μηχανισμό που εγκρίθηκε την προηγούμενη εβδομάδα κατά την ένατη επιτροπή της καθήλυνα αρμόδια, ένα συνεδρίας καθήλυνα αρμόδιας επιτροπής που έλαβε χώρα κάποια στιγμή το Μάρτιο. Εμείς καταλήγουμε στο εξή. Αυτός ο μηχανισμός ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικός και θα σας το εξηγήσω αυτό όχι μόνο για αυτά που επιτυγχάνει επιτόπου αλλά και διότι έχει κατορθώσει να τον οικειοποιηθούν όλα τα κράτη-μέλη και να υπάρξει συντονισμός δράσεων των κρατών μελών. Κύριε Πρόεδρε, η ανάλυση μας όσον αφορά τη λειτουργία αυτής της κατευθυντήρης επιτροπής είναι ε, ιδιαίτερα θετική, προσφέρει η Επιτροπή προς τη θέμενη αξία και όσοι συμμετέχουν αισθάνονται ότι και συμμετέχουν στη διαδικασία λήψη αποφάσεων. Θέλω λοιπόν να συντονίσουν όχι μόνο αυτά που υπάρχουν σε ενωσιακό επίπεδο, αλλά και σε αυτά που συμβαίνουν στην Τουρκία. Και ο συνάδελφός μου παρακατήμενος θα επανέλθει από αυτού. Όσον αφορά ε, τη δήλωση Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία 18 Μαρτίου προβλέπεται η εκταμείευση άλλων τριών δις στο πλαίσιο του μηχανισμού για την Τουρκία, Βεβαίως ε, στο βαθμό που θα χρησιμοποιηθούν ε, στο έπακρο αυτά τα κονδύλια και υπό την προπόθεση ότι θα καλύπτονται και οι προποθέσει. Τα τρία δις ε, πλέον έχουν προσημειωθεί. Έχουμε 72 προγράμματα που έχουν επιλογή. 1,5 δις έχουν ήδη εκταμιευτεί και αυτός είναι ο λόγος ε, γιατί παρότι υπάρχει, υπάρχουν λόγοι να επικρίνουμε την Τουρκία για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κράτους δικαιού, παρόλα αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρίνει ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να προτείνουμε την παράταση του μηχανισμού. Κυρίως με το σκεπτικό ότι η Τουρκία έχει τηρήσει τις δεσμεύσεις της με βάση αυτά που αποφασίστηκαν στις 26 Μαρτίου και σε σχέση πάντα με τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει για θέματα προσφύγων. Γι' αυτό λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα η Επιτροπή αποφάσισε να παρατείνει το μηχανισμό, τη λειτουργία του μηχανισμού και θα μου επιτρέψετε να δώσω το λόγο στον κύριο Φεράν που είναι ε, διευθυντής ε, και αρμόδιος για θέματα Τουρκίας και ο οποίος θα σας δώσει και μια πολιτική εξήγηση για το όλο θέμα και μετά θα επανέλθω εγώ, ε, θα κάνω μια μικρή ανακεφαλαίωση και θα επισημάνω τα δημοσιονομικά θέματα. Στο πολύ θα προσπαθήσω να συνοψίσω τα βασικά επιτέγματα του μηχανισμού. Τα στοιχεία αυτά έχουν δημοσιευθεί στην ε, έκθεση που αφορούν το μηχανισμό την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτά τα επιτέγματα ε, αποτέλεσαν δικείμενο εξηγής ε, στην Διοικητική Επιτροπή στις 29 Μαρτίου. Εκφράστηκε τότε και η ξεκάθαρη επιθυμία για διαφάνεια στο, ως προς το Κοινοβούλιο. Έχουμε προσθέσει, ε, αποδείξει τόπου ότι υπάρχει προστιθέμενη ε, αξία. Πάνω από 1,2 εκατομμύρια προσφύγων αποφελήθηκαν από τη βοήθεια, κυρίως στο μης εκπαίδευσης και της ε, υγείας. Μέχρι τώρα στην εκπαίδευση έχουμε ε, χάρη στις δράσεις μας πάνω από 300.000 παιδιά έχουν επιστρέψει στο σχολείο στη Τουρκία, έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό, κατάρτιση, ε, μαθήματα ε, τουρκικών, βοήθεια στο τομέα της υγείας, άμεση βοήθεια. Μέχρι τώρα συστήσαμε 12 κινητές μονάδες υγείας 760.000 ε, επισκέψεις, ε, έχουν γίνει εμβολιασμοί, μεταξύ άλλων. Αυτά τα βασικά επιτεύγματα που θα ήθελα να υπογραμμίσω σχετικά με την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού. Η κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκία συνεχίζει να υλοποιείται και επιβεβαιώθηκε από τα κράτη-μέλη ομόφωνα και θεωρήσαμε ότι είχε έρθει η ώρα να ε, εκταμιέσουμε το, ε, τη δεύτερη ε, δόση του μηχανισμού. Ε, υπήρχε έκτακτη ανάγκη, θα σας εξηγήσω γιατί. Όπως σας είπα, ένα από τα βασικά επιτεύγματα παρατηρήθηκε, διαπιστώθηκε στο τομέα της εκπαίδευσης. Είναι σημαντικό για να μην χαθεί μια ολόκληρη γενιά παιδιών. Ε, με το ε, τουρκικό Υπουργείο Παιδείας. Υπάρχει συμβόλαιο που λύγει στις 3, ε, σύμβαση που λύγει στις 3 Οκτωβρίου. Χρειάζονται προετοιμασίες προκειμένου να μπορέσουμε να ε, υπογράψουμε την παράταση αυτής της συμφωνίας και χρειαζόμαστε απόφαση Τώρα, προκειμένου όλες οι διαδικασίες, στις οποίες συμμετέχετε κι εσείς, να οδηγήσουν στην διόρθωση του προϋπολογισμού του 2018 προκειμένου να γίνει εγκαίρωση ή απαραίτητη εκταμίευση. Ο διορθωτικός προϋπολογισμός καλό θα ήταν να εγκριθεί ε, στην Ολομέλεια σας τον Ιούλιο. Γι' αυτό το λόγο ε, πήραμε αυτή την απόφαση, η οποία και κοινοποιήθηκε στις 9 Μαρτίου. Οι συμμετέχοντες έλαβαν την ενημέρωση ότι η Κομισιόν θα ε, υιοθετήσει αυτή την απόφαση. Σε ό,τι αφορά το προπολογισμό θα ξαναδώσω το λόγο στην συνάδελφο σχετικά με τις πηγές των κονδυλίων. Γνωρίζετε ότι όταν κάναμε την παρουσίαση της πρότασης της Κομισιόν στο Συμβούλιο, υπήρχαν πολλές αντιδράσεις από αρκετά κράτη-μέλη που ε, δεν συμφωνούσαν. Η Κομισιόν θεώρησε ότι δεν θα ήταν η καλύτερη προσέγγιση, μιας και αυτό θα σήμαινε ότι θα ε, χρησιμοποιούσαμε μεγάλο κομμάτι του δημοσιονομικού του προϋπολογισμού που προβλεπόταν για άλλους ε, σκοπούς. Όπως ξέρετε, υπάρχουν ανάγκες που απορρέουν από τη κρίση στη Συρία. Η Ευρώπη πρέπει να ανταποκριθεί και όπως γνωρίζετε πρέπει να υποστηρίξουμε με τον προπολογισμό ε, μας και την απασχόληση και την ανανάπτυξη. Προβλέπονται κονδύλια για την ε, υποστήριξη της απασχόλησης των για την αντιμετώπιση των αναγκών σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και την μετανάστευση. Γι' αυτό το λόγο η Κομισιόν πρότεινε να ε, ε, να χρησιμοποιηθούν ένα εκατομμύριο από το προπολογισμό της, Ευρωπαϊκής, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δύο εκατομμύρια από τα κράτη-μέλη αυτός ο μηχανισμός δεν αφορά την αποστολή χρημάτων στη Τουρκία, αλλά την, ε, ε, την αντιμετώπιση των βασικών αναγκών των προσφύγων στη Τουρκία. Πιστεύουμε ότι η αποτελεσματικότητα, η αποτελεσματική υλοποίηση της συμφωνίας σε ό,τι αφορά τις ροές μεταναστών και προσφύγων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτούν μια άμεση απάντηση εκ μέρους μας και αυτό προσπαθούμε να επιτύχουμε με την πρότασή μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Καλβίνιο, κυρία ε, Φεράν. Σας ευχαριστώ πολύ και στις δύο. Θα ξαναδώσω το λόγο στον Γενικό Εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπατε στην εισαγωγή σας, όταν διαπραγματευόμασταν τον προπολογισμό για το 2018, ξέραμε ότι θα προέκυπεται αυτό το ζήτημα και ότι το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Κομισιόν θα έπρεπε να αποφασίσουν από κοινού αν θα συνεχιστεί ο μηχανισμός στήριξης για την Τουρκία, για τους πρόσφυγες στην Τουρκία ή όχι. Ε, καλώς ήρθατε ε, στο Κοινοβούλιο σήμερα το ε, πρωί. Ε, το εκτιμούμε που είστε εδώ σήμερα. Θα ήθελα να σημειώσω τρία πράγματα. Πρώτο απ' όλα η συνεργασία ανάμεσα στην Κομισιόν και το Κοινοβούλιο. Δεύτερον, ο ρόλος του Κοινοβουλίου. Τρίτον, η χρηματοδότηση του μηχανισμού για τους πρόσφυγες στη Τουρκία σε ό,τι αφορά τη συνεργασία Κοινοβουλίου Κομισιόν. Κατά τη γνώμη μου, αυτή η απόφαση και το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού που θα μας ε, προταθεί θα είναι από τους πιο σημαντικούς διορθωτικούς προπολογισμού των τελευταίων ετών. Το ποσό είναι σημαντικό, η προσοχή των, του κοινού είναι ουσιαστική σημασία. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να συνεργαστούμε ε, με ειλικρινή τρόπο, όπως γνωρίζετε όταν ξεκίνησε ο μηχανισμός, όταν ε, εμείς ενημερωθήκαμε από δημοσιεύσεις στο τύπο. Μην το ξανακάνετε αυτό σας παρακαλώ. Ξέρουμε ότι υπήρχε έκτακτη ανάγκη, αλλά μην το ξανακάνετε στο μέλλον. Δεν, το, δεν σημαίνει αυτό ότι, δεν θα το, ότι θα το δεχτούμε, αλλά ενημερώστε ε, με, τον, ε, με επαρκή τρόπο το κοινοβούλιο, το οποίο πρέπει να συμμετέχει με το κατάλληλο τρόπο. Η Κομισιόν, ναι, ενημέρωσε το Κοινοβούλιο αμέσως μετά τη λήψη της απόφασης από το Σώμα Επιτρόπων. Ήταν κατάλληλη στιγμή, αλλά δεν ήταν σωστό που ε, δημοσιεύτηκε πρώτα η απόφαση στο τύπο, εγώ το ε, διάβασα εκείνο το πρωί από το, στο πολίτικο, έτσι έμαθα για την απόφαση. Ε, ενώ το Κοινοβούλιο είναι τμήμα της αρχής προπολογισμού. Αν μπορείτε να μας δώσετε περισσότερες στοιχεία για το Ποιο γέρευσε στοιχεία στο τύπο σχετικά με αυτή την απόφαση θα το εκτιμούσαμε. Εξαιτίας της ε, ουσιαστικής σημασίας της συνεργασίας μας, σκεφτόμουν ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει περιθώριο προκειμένου να υπάρξει η απαραίτητη ευελιξία στην υλοποίηση του, του μηχανισμού στήριξης. Όταν μου τέθηκε το ερώτημα, ε, είπα ότι πρέπει να υπάρξει τέτοιο περιθώριο και στην περίπτωση της ε, Τουρκίας. Πρέπει να συνεργαστούμε, έχουμε ευθύνη, είναι φυσικά απαραίτητη η διαφάνεια και πρέπει να συμμετέχουμε. Δεύτερον, Σήμερα το πρωί συζητήσαμε για μια μελέτη για τη διαχείριση των καταπιστευμάτων και ε, αναφέρθηκε ο μηχανισμός στήριξης για τους πρόσφυγες στην Τουρκία. Και οι συνάδελφοι δεν αμφισβήτησαν τη σημασία αυτού του μηχανισμού. Και σίγουρα επιτόπου ο μηχανισμός αυτός ήταν αποτελεσματικός, αλλά σε ό,τι αφορά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, την ε, δημοκρατική λογοδοσία. Το Κοινοβούλιο θέτει στην Κομισιόν κάποια ερωτήματα. Γιατί δεν πρότεινε το Κοινοβούλιο να συμμετέχει στην Επιτροπή ε, τη Διοικητική Επιτροπή του ε, Μηχανισμού και τρίτον σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση. Πολλές φορές συζητήσαμε για τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε ε, από κοινού. Έχουμε κάποιες προτεραιότητες που πρέπει να χρηματοδοτηθούν Ε, προβλήματα κάποιων ε, project ε, για την υλοποίησή τους. Φυσικά, πριν δούμε το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού της Κομισιόν, δεν μπορούμε να εκφράσουμε κάποια γνώμη, αλλά σίγουρα οι καινούριες προτεραιότητες χρειάζονται νέες χρηματοδοτήσεις. Καταφέραμε να αφήσουμε περιθώριο 250 εκατομμυρίων. Και συνολικά 1,6 δισεκατομμύριο είναι το περιθώριο. Αυτό αφήνει περιθώριο 3,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πιστεύω λοιπόν ότι το ένα δισεκατομμύριο πρέπει να προέρχεται από νέα κονδύλια και όχι από ανακατανομή κονδυλίων, γιατί όσο και αν είναι η πίεση, είναι ε, καλύτερο ε, να διαθέτουμε νέα κονδύλια για ε, νέες προτεραιότητες. Αυτά είχα να σας πω. Ευχαριστώ πολύ την Κομισιόν για την παρουσίαση της εδώ και είμαι ανυπόμονος να λάβουμε περαιτέρω ενημέρωση σχετικά με αυτά τα ζητήματα και να συνεργαστούμε κάτι που είναι πολύ σημαντικό δεδομένης της πολιτικής σημασίας αυτού του εγχειρήματος. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Δελανού. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ απόλυτα με τις ε, παρατηρήσεις του κυρίου Μουρεσάν. Έβαλε το δάκτυλο επί των τύπων των ήλων. Τα κράτη να οργανώσουν την κοινή πολιτική εκτός των κανόνων λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό δηλαδή, σημαίνει ότι η Κομισιόν και οι συνομοθέτες ε, Συμβούλιο και Κοινοβούλιο να του αφήνουν εκτός, ε, δημιουργεί πρόβλημα. Ε, και ειδικά όταν βάζουν το χέρι, από το, όταν βάζουν το χέρι στο Γκορβανά, ας πούμε, τότε σημαίνει ότι δεν υπάρχει πια εμπιστοσύνη. Δεν νομίζω ότι πρέπει να δεχτούμε αυτήν την κατάσταση. Και νομίζω ότι πρέπει να σας πω σήμερα ότι περάσαμε την κόκκινη γραμμή. Πρέπει να επανέλθουμε σε πράγματα πιο κανονικά. Το θέμα των προσφύγων δεν λύνεται με την ε, συμφωνία με την Τουρκία. Είναι ένα παγκόσμιο θέμα, συνολικό θέμα, πρέπει να αντιμετωπίσουμε συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένω, αυτό το συνολικό του προβλήματο σημαίνει ότι όλα τα θέματα που συνδέονται με του μετανάστε θα πρέπει να ενσωματωθούν και να επιληθούν και να χρηματοδοτηθούν από τον προπολογισμό τη Ένωση. Πρέπει να το κάνουμε αυτό. Πρέπει να μην έχουμε διάφορες μικροπολιτικές ας πούμε, ε, οι οποίες ε, περιφέρονται ας πούμε άσχετες μεταξύ τους. Ας πούμε. Θα πρέπει να λειτουργεί η Ένωση κανονικά με τους συνομοθέτες μαζί που έχουν κοινή ευθύνη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Άλλη, ένα λεπτό. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω για όλες τις λεπτομέρειες που ακούσαμε για την παράταση του μηχανισμού στήριξη των προσφύγων στην Τουρκία. Αυτή η δεύτερη περίοδος δεν θα είναι και πολύ διαφορετική από την πρώτη περίοδο. Προκύπτει από την απόφαση που ελήφθη. Σε ό,τι αφορά, ούτε σε ό,τι αφορά την διάρκεια, ούτε σε ό,τι αφορά το μοντέλο χρηματοδότηση. Το μοντέλο είναι ακριβώ το ίδιο. Δηλαδή, ένα τμήμα από τον προπολογισμό τη Ένωση και ένα άλλο τμήμα από συνεισφορέ των κρατών μελών. Η κατάσταση των προσφύγων στην Τουρκία αυτή τη στιγμή δεν έχει αλλάξει σε σχέση με τη στιγμή, χρονική στιγμή που ξεκίνησε να λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός. Ο αριθμός των προσφύγων έχει φτάσει και έχουν ξεπεράσει τα 3,5 εκατομμύρια άτομα. Και 284.000 παιδιά γεννήθηκαν στο μεταξύ. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξουμε το πώς εφαρμόζουμε το μηχανισμό αυτό σε σχέση με την πρώτη φάση και τι πρέπει να κάνουμε ούτω ώστε να λύσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν. Λαμβάνοντας υπόψη τα διδάγματα που πήραμε από τα λάθη του παρελθόντος, πώς μπορούμε λοιπόν, πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την εφαρμογή του μηχανισμού αυτού σε αυτή τη δεύτερη φάση. Ερωτήσεις λοιπόν. Οι βασικές αρχές θα πρέπει να είναι η ταχύτητα, η αποτελεσματικότητα, και η καλή ή χρηστή οικονομική διακυβέρνηση. Μιλάμε για 3 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο. Δώσαμε ήδη για την περίοδο 16-17. Αυτές οι βασικές αρχές στην πρώτη φάση έγιναν σεβαστές. Τώρα, το 2017 τα κράτη-μέλη έδωσαν περίπου 1,5 δις ευρώ. Το 97% έχουν ήδη εκταμιευθεί από αυτά τα 1,5 δις. Έτσι. Περιμένουμε λοιπόν την κινητοποίηση του, των υπόλοιπων κονδυλίων για την περίοδο 2018-2019. Η καταληκτική ημερομηνία το 2021 υποτίθεται. Υπάρχει δυνατότητα να βελτιώσουμε την ταχύτητα και την πειθαρχία σε ό,τι αφορά την αποδέσμευση των κονδυλίων στην δεύτερη φάση. Και τρίτον, τι γίνεται με την αποτελεσματικότητα του Ταμείου. Ε, μπορείτε να μας πείτε κάποια λόγια. Κυρία Γκρέσλερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ έχω ενοχληθεί από αυτή τη συζήτηση γιατί είχα την εντύπωση ότι όσον αφορά αυτή τη ε, δεύτερη δόση τελικά ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα. Η Τουρκία εντωμεταξύ όχι μόνο έχει ξεκινήσει πόλεμο αλλά και η ίδια προκαλεί μετακινήσεις και πρόσφυγες. Με ενδιαφέρει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη τελική ανάλυση πώς το βλέπει αυτό. Η Τουρκία δεν είναι πια ίδια, έχει αλλάξει ρόλο. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τώρα τι κάνουμε. Επιβραβεύουμε αυτόν που προκαλεί προβλήματα. Ως ε, Επιτροπή Προϋπολογισμών επισκεφτήκαμε επιτόπου την κατάσταση. Ε, βέβαια η Τουρκία συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά βλέπουμε επίσης ότι η Τουρκία έχει στα χέρια της ένα πολύ σημαντικό δημοσιονομικό μέσο. δείτε λοιπόν το εξή ερώτημα. Ακούμε για σχολικά κτίρια, για ιατρική περιθάλψη. Τα έχουμε ακούσει αυτά πολλές φορές. Αλλά είμαστε ειλικρινά σίγουροι ότι και εμείς δεν συγχρηματοδοτούμε τον πόλεμο κατά της Συρίας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για αυτή τη σημαντική ερώτηση. Η κυρία Γκουάρδια Θαβάλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, πολύ γρήγορα, γιατί όλοι γνωρίζουμε πόσα, πόσους πρόσφυγες έχει φιλοξενήσει η Τουρκία. Ε, το βασικό είναι ότι η Ευρώπη δεν ήθελε να έρθουν σε εμά, έτσι. Επομένως, τουλάχιστον μου φαίνεται λογικό να προσπαθήσουμε να δώσουμε μια οικονομική βοήθεια για να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην υγεία αυτοί οι άνθρωποι, καθώς και μια στέγη πάνω το κεφάλι τους. Τέλος. Όπως είπε η κυρία Κρέσλερ, είναι αλήθεια ότι η σχέση με την Τουρκία είναι πάρα πολύ ευαίσθητη. Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία ε, υπαναχώρησε. Ε, οι ΜΚΟ και οι εθελοντέ που δουλεύουν εκεί δεν είναι οι καλύτεροι, δεν υπάρχει ελευθερία τύπου και όλα αυτά μας, μας δημιουργούν πολλές αμφιβολίες, απροθυμία αν θέλετε, να εκταμιευθούν αυτά τα κονδύλια να δοθούν αυτά τα κονδύλια. Όμως είπατε, υπάρχουν όμως εκεί, είναι εκεί οι πρόσφυγες, υποφέρουν και υποφέρουν συχνά και γιατί ε, είναι αδρανή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένω, κάτι πρέπει να κάνουμε, τουλάχιστον να χρηματοδοτήσουμε. Θα πρέπει να βάλουμε δύο, δύο βασικά κριτήρια λοιπόν. Πρώτον, συνθήκε πολύ λεπτομερεί. Πολύ λεπτομερεί για να ξέρουμε τι κάνουμε με αυτά τα λεφτά και να είμαστε σίγουροι ότι και το τελευταίο σεντ από αυτό το ταμείο πηγαίνει για τους πρόσφυγες. Και να μην έχουν τάσεις οι Τούρκοι έτσι, να χρησιμοποιούν αυτά τα λεφτά για άλλα πράγματα. Δεύτερον, για τη χρηματοδότηση. Αυτά, αυτό το ένα δις είναι το όριο που πρέπει να βάλουμε. Δεν μπορούμε να πάμε πιο πέρα, έτσι. Εάν θέλετε αυτά τα τρία ε, δισεκατομμύρια να τα δώσουμε πάντω από τον κοινοτικό προπολογισμό, θα πρέπει να αλλάξει το πουδουπού. Γιατί δεν μπορεί, δεν γίνεται έτσι με το σημερινό πουδουπού να δοθούν από τον προπολογισμό τη Ένωση. Λοιπόν, θα σα δώσω το λόγο σε αυτού που τον ζητήσατε, αλλά σα παρακαλώ πολύ πολύ γρήγορα. Ο κ. Κολμάιε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Στη Γερμανία έχουμε ένα αστείο που το λέμε, το χρησιμοποιούμε όταν πρόκειται για θέματα χρόνου. Δηλαδή το αστιάκι είναι το εξή, ότι φέτος τα Χριστούγεννα θα έρθουν πολύ νωρί. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Λοιπόν, εγώ ε, θεωρώ ότι η συμφωνία με την ε, Τουρκία εκπνέει η εξέπνευσε στις 3 Οκτωβρίου. Αυτό το ξέραμε όμως εκ των προτέρων. Γι' αυτό λοιπόν θα σας πω για άλλη μια φορά ότι χρειαζόμαστε επιτέλους μια σαφή στρατηγική, ένα σαφή στόχο για το τι ακριβώς χρειαζόμαστε ως προς το μεταναστευτικό. Προφανώς και θέλουμε να βοηθήσουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως έχει ήδη βοηθήσει. Ε, και εγώ εντάξει λέω να βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο. Όμως μόνο εφόσον παράλληλα υπάρχει και ένα σαφής πολιτικός στόχος. Αν δεν υπάρχει σαφής πολιτικός στόχος τελικά κάθε χρόνο θα καταβάλουμε περισσότερα κονδύλια, θα πληρώνουμε περισσότερο για καταβλισμούς, για αιστείες κρίσης και σε τελική ανάλυση δεν θα ξέρουμε ποιος είναι ο στόχος μας. Γι' αυτό λοιπόν σας λέω ότι χρειαζόμαστε απαραίτητα στόχους. Και για μένα είναι σημαντικό άλλο ένα ερώτημα. Υπάρχει μια συμφωνία με την Τουρκία της τάξης των περίπου 3 δις ευρώ. 1,85 δις έχουν ήδη καταβληθεί. Πριν τώρα αποφασίσουμε για άλλο ένα δις, θέλω να αποφασίσω γιατί το υπόλοιπο από τα τρία δεν έχει καταβληθεί και αν τελικά θα καταβληθεί θέλω να γνωρίζω πότε. Αυτά είναι σημαντικά στοιχεία. Να μας τα πείτε σήμερα, όχι να μας τα πείτε μετά από κάποιους μήνες. Ο κύριος ε, Ομπαρτ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν να πω ότι αυτά που είπε η συνάδελφός μας, η προαλήσα σα, συμφωνώ απόλυτα με αυτά. Δεν χρειάζεται να τα παραλαμβάνουμε. Νομίζω βέβαια είναι απόλυτα σαφές ότι υπάρχει μια επίγουσα ανθρωπιστική ανάγκη έκτακτη περίπτωση, πήγουσα ανάγκη όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεπλάκησε αυτό το μηχανισμό. Από όλα λοιπόν που έχω ακούσει, έχω δει και με όσους ε, έχω μιλήσει και με την ΟΝΤΙΡ, η ΟΝΤΙΡ ε, πολύ καλή δουλειά κάνει, πρέπει να το πούμε αυτό, ο οργανισμός ΟΝΤΙΡ ε, γιατί ε, ο βασικός σκοπός αυτού του οργανισμού είναι να καλύπτει ανθρωπιστικές ανάγκες. Όμως, επιτρέψτε μου να ε, κρούσω λιγάκι και τον κόντονα του κινδύνου. Υπάρχει κίνδυνος η Ευρωπαϊκή Ένωση να εμπλακεί σε μία χρηματοδότηση στο δίνεκές. Ε, δεν ξέρω τώρα ποια θα είναι η στρατηγική, αλλά ελπίζω και επιθυμώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει και μια στρατηγική εξόδου από αυτό το φαύλο κύκλο. Φυσικά, δύο τελευταίες παρεμβάσεις. Πάρα πολύ γρήγορα. Ο κύριος Ντεπχέ πρώτος και καλύτερο. Πολύ σύντομα, Πρόεδρε. Πάντα θεωρούσε, παρότι δεν ήταν δημοφιλές, ότι η συμφωνία υπεργολαβίας που έχουμε συνάψει με την Τουρκία για να ασχοληθεί με τους μετανάστες που δεν τους θέλουμε, δεν θέλουμε να τους έχουμε εδώ πέρα, ήταν κάτι που πρέπει να υποστηρίξουμε. Έτσι, μια και είμαστε σε μια λεπτή κατάσταση στο εσωτερικό της Ένωσης. Έχω λοιπόν δύο ερωτήσεις προς την Κομισιόν. Ε, προς την κατεύθυνση που μας είπε και ο προηγούμενος ομιλητή Τη στιγμή που πληρώσαμε την πρώτη δόση των τριών δις, έτσι, όλοι ξέραμε τι θα συνέβαινε. Και τη στιγμή τη πρόταση προπολογισμού για το 2018 η Κομισιόν δεν ενσωμάτωσε αυτή την πρόταση, έτσι, στον προπολογισμό. Έτσι, κάναμε, λε και δεν υπήρχε. Όμω το ξέραμε ότι θα υπήρχαν και άλλε δύο δόσει, έτσι. Λέω στην Κομισιόν λοιπόν. Έχουμε την αίσθηση ότι δεν υπήρχε προβλεψιμότητα εδώ πέρα, έτσι, και μας βάζετε πρώτα τελεσμένων. Ε, δεύτερη ερώτηση. Τελικά, για πόσο καιρό θα πληρώνουμε. Ποιο είναι το όριο. Από ποια στιγμή και μετά θα πούμε με ένα τμήμα αυτών των προσφύγων ε, δεν είναι πια πρόσφυγες, ε, αλλά είναι τμήμα ε, αυτής της συμφωνίας υπεργολαβίας. Για πόσο καιρό τέλο πάντων θα συνεχιστεί. Κύριε Ντριάντ, η τελευταία ομιλήτρια. Σύντομα πρέπει να το δούμε πιο μακροπρόθεσμα. Εμείς το βλέπουμε πολύ ε, κοντόθωρα, έτσι. Δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι η Ευρώπη δεν θέλουν να πάρουν αυτούς τους ε, πρόσφυγες, είναι πρόθυμοι ή το κάνουν πολύ αργά, επομένως πρέπει να αρχίσουμε να κοιτάμε πιο μακροπρόθεσμα, μια προσέγγιση πιο μακροπρόθεσμη. Γιατί εκεί είναι το σημείο κλειδί. Ε, θέλουν τα κράτη-μέλη να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν, εάν θα το κάνουν έστω και αυτό. Θα πρέπει να βρούμε λύσεις ε, για να λύσουμε τη σύγκρουση ε, και να ε, βοηθάμε τους ανθρώπους αυτούς να μην φεύγουν από τη χώρα προέλευσής τους. Θέλουμε μια πιο μακροπρόθεσμη, μια πιο ολιστική προσέγγιση. Ευχαριστώ. το εξής ζήτημα. Αν μπορούσαμε να είχαμε συζητήσει αυτό το θέμα όταν συζητήθηκε το προπολογισμό του 18, θα ήταν καλύτερα. Σήμερα, αν αυτά τα χρήματα θα διατεθούν από ε, ανακατανομή κονδυλίων, από νέα κονδύλια, τι να πω, θα θέλαμε μια απάντηση από την Κομισιόν. Παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση. Σημειώνουμε τις παρατηρήσεις και προτάσεις όλων. Πιστεύω ότι ουσιαστικά το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν συμφωνούν ως προς τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν και ότι πρέπει να βρεθεί απαραίτητη ε, ισορροπία στην αντιμετώπιση αυτών των αναγκών. Σε ό,τι αφορά τη λογοθεσία και τη διαφάνεια, συμφωνούμε απόλυτα με το Κοινοβούλιο ότι χρειάζεται να ενισχυθούν. Γι' αυτό το λόγο επιμείναμε και καλέσαμε το Κοινοβούλιο σε όλες τις συναντήσεις στις οποίες συζητάμε τις λεπτομέρειες της ε, υλοποίησης του μηχανισμού και στις 9 Μαρτίου ήδη είχε ανακοινωθεί ότι ε, ετοιμάζει αυτή την ε, απόφαση η Κομισιόν. Επίσης, αποστέλουμε στο Κοινοβούλιο κάθε μήνα εκθέσεις υλοποίησης και ε, φροντίζουμε να δίνουμε όσες περισσότερες λεπτομέρειες γίνεται στην ετήσια έκθεση. Ευπρόσδεκτες οι ε, προτάσεις, αλλά όσο αφορά την ενημέρωση, έκανα ό,τι μπορούσα. Κάνουμε το μέγιστο δυνατό. Αν χρειάζεται κάτι, χρειάζεστε κάτι παραπάνω, πείτε το. Ε, μηνιαίες εκθέσεις, λεπτομερείς εκθέσεις, ε, αιτήσεις εκθέσεις. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε για να υπάρχει περισσότερη λογοδοσία, περισσότερη ε, διαφάνεια σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του μηχανισμού. Το ο μηχανισμός αυτός είναι νέο νομικό εργαλείο και στην πράξη υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι συντονισμού και υλοποίηση, αλλά ουσιαστικά χρησιμοποιούμε ε, κονδύλια από την ανθρωπιστική βοήθεια, από την προενταξιακή βοήθεια και χρησιμοποιούμε τους κανόνες ε, του προϋπολογισμού σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση. Πράγματι, στις διαπραγματεύσεις ε, ήταν να πάρουν το ζήτημα αυτό και συμφωνούμε πλήρως με το Κοινοβούλιο ότι τα ε, ε, κονδύλια πρέπει να προέρθουν από τα ε, περιθώρια του που αφήνει ο προπολογισμό όσο περισσότερο γίνεται. Στην ουσία πρόκειται για ανθρωπιστική βοήθεια και για τα υπόλοιπα πρέπει να ε, πρόκειται για νέα κονδύλια που προέρχονται από τα περιθώρια. Τρίτον, σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα και τις σχετικές προκλήσεις. Όπως σας είπα προηγουμένως, όπως είπατε, ε, κάποια από σας είπατε, είναι ευαίσθητη η σχέση μας με την Τουρκία και γι' αυτό την ώρα που ε, αυξάνουμε τη χρηματοδότηση, ελήφθη πολιτική απόφαση να ε, μειωθούν τα κονδύλια που διατίθενται στην προενταξιακή βοήθεια εν μέρη για τον προπολογισμό αυτού του έτους και εν μέρη για τον προπολογισμό του επόμενου έτους. Προσπαθούμε να βρούμε την απαραίτητη ισορροπία χρησιμοποιώντας τα εφιστάμενα εργαλεία και αντιμετωπίζοντα τις διάφορες προτεραιότητες. Συμφωνούμε πλήρως με το Κοινοβούλιο ότι πρέπει να φροντίζουμε τα ε, κονδύλια αυτού του μηχανισμού να πηγαίνουν για τους πρόσφυγες. Η πολιτική αυτή πρόκληση έχει σχέση και με το, τη χρονική στιγμή. Αν ε, κινηθούμε υπερβολικά νωρίς, υπάρχει ρίσκο να μην τηρηθούν, να μην αντιμετωπιστούν όλα τα κριτήρια. Άμα ε, δραστηριοποιηθούν πολύ αργά θα είναι και αυτό πρόβλημα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα κονδύλια που μπορούν να διατεθούν για αυτό το μηχανισμό. να μην ξεπεράσουμε τα όρια χρηματοδότησης του φετινού προϋπολογισμού και πρέπει να βρεθεί απαραίτητη ισορροπία με ε, λεπτομερή ενημέρωση να ξέρουμε πότε θα έχουν εξαντληθεί τα 3 δισεκατομμύρια και τι σκοπεύουμε να κάνουμε στο μέλλον. Όπως και να πρέπει να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με επικοδομητικό τρόπο προκειμένου να βρούμε μία λύση, όχι μόνο για τώρα, αλλά όπως ε, είπατε να ε, σκεφτούμε να εξετάσουμε μία ε, μακροπρόθεσμη λύση, την οποία δεν θα βρούμε σήμερα, αλλά θα πρέπει να το συζητήσουμε για να ε, υπάρχει ένα ε, σταθερό πλαίσιο στο μέλλον. Θα επανέλθουμε σε αυτό. Κυρία Φεράν, πολύ σύντομα παρακαλώ, γιατί ε, έχουμε αργήσει. Τρία σημεία πολύ σύντομα για την ε, πολιτική κατάσταση των σχέσεων με την Τουρκία και η θέση του μηχανισμού στο εσωτερικό, η εκτέλεση και τη στρατηγική εξόδου που υπάρχει και την προετοιμάζουμε. Λοιπόν, καταρχά, ο μηχανισμό δεν είναι μία ανταμοιβή για την Τουρκία. Έτσι, είναι σαφέ ότι το, τα λεφτά πάνε για του πρόσφυγε. Και ήταν μόνο ένα τμήμα των συνολικών σχέσεων που έχουμε με την Τουρκία. Ο Επίτροπο Χαν ήταν εχθέ στην Ολομέλεια τη ομάδα τη ΑΦΕΤ για να παρουσιάσει το στρατηγικό διάλογο για το μέλλον του προεταξιακού εργαλείου και η Κομισιόν προτείνει μία περικοπή 750 εκατομμυρίων ε, μέσα στα επόμενα τρία χρόνια. Ο μηχανισμός δεν αφορά, δεν πηγαίνει δηλαδή ε, στο κράτος, στο τουρκικό, αλλά στους πρόσφυγες. Σε ό,τι αφορά την εκτέλεση. Μία γρήγορη και αποτελεσματική εκτέλεση με πλήρη σεβασμό των αρχών καλής ε, και χρηστής οικονομικής διαχείρισης είναι η βάση της διαχείρισης του, ε, του μηχανισμού. Το ελεκτικό συνέδριο ετοιμάζει ένα, μια έκθεση ελέγχου που θα είναι έτοιμη πριν το καλοκαίρι και που θα δίνει όλες τις εγγυήσει για να είμαστε σίγουροι ότι σε, σεβόμαστε τις αρχές της χρηστής οικονομικής διαχείρισης ή όχι. Δεν έχουμε ακόμα την έκθεση. Ε, είναι τμήμα της ε, προσεκτικής παρακολούθησης εκτέλεσης ε, του μηχανισμού. Έχουμε εξοδέψει ένα δισεκατομμύριο 850 εκατομμύρια ευρώ μέχρι στιγμής. Γιατί όχι περισσότερο, γιατί ε, σεβόμαστε τους κανόνες χρηστής οικονομικής διαχείρισης και με σεβασμό των κανόνων της Ένωσης ξοδεύοντα ξοδεύοντας δόση-δόση. Όλα τα συμβόλαια έχουν υπογραφεί. Αυτό σημαίνει ότι το σύνολο των κονδυλίων είναι σε φάση χρησιμοποίηση. Φυσικά οι τελικέ πληρωμέ δεν θα δοθούν παρά μόνο όταν τα project ολοκληρωθούν. Και στα πλαίσια των project έχουμε project για υποδομέ, όπω την ε, ε, οικοδόμηση δύο νοσοκομείων. Η τελική πληρωμή για αυτά τα νοσοκομεία δεν θα καταβληθεί πριν το 2020-2021. Η καταληκτική ημερομηνία για τις πληρωμές είναι 2021 αλλά όλα τα προγράμματα έχουν ε, ήδη ξεκινήσει και δεν υπάρχουν ε, κι άλλες ε, πιστώσεις ανάληψη υποχρεώσεων. Λοιπόν, αυτό που είπαμε ήταν ότι δεν θα έπρεπε να έχουμε μηχανισμό για τους, για πρόσφυγες για την Τουρκία, θα πρέπει να έχουμε κονδύλια για τους πρόσφυγες της Συρίας τελεία. Ο κύριος Μουρεσάν. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την Επιτροπή που ήρθε. Καταρχήν ε, νομίζω ότι όλα αυτά που είπαν οι συνάδελφοι είναι πολύ σημαντικά. Εμείς θέλουμε να εμπλακούμε σε αυτό, να δούμε λιγάκι τον διορθωτικό προϋπολογισμό και να μπορέσουμε και να καλύψουμε τις, να δούμε να καλύπτονται οι προϋποθέσεις που έχει ορίσει το Κοινοβούλιο για όλο αυτό το θέμα. Κύριος Τζέτη, εσείς που ασχοληθείτε με τον προπολογισμό το 2019, Ξέρετε ότι θα έχετε πιστώσει για το μηχανισμό για τους πρόσφυγες από τη Συρία στην Τουρκία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τους διάφορους ομιλητές και θα περάσουμε στην ψηφοφορία. Παρακαλώ βάλτε τις ηλεκτρονικές σας κάρτες ε, στο μηχανάκι. Θα κάνουμε μία πρώτη δοκιμή. Ψηφίζουμε τώρα. Ψήφισαν όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Πολύ ωραία. Πρώτη ψηφοφορία. Έχουμε τον προϋπολογισμό 2018. Θα δώσω το λόγο στο Γενικό Εισηγητή για να μας παρουσιάσει το σχέδιο για τη μεταφορά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σύντομα είναι μια μεταφορά που δεν ήταν καθόλου προβληματική το 2017 ε, λόγω της, ε, λόγω της ε, αργής νομικής βάσης ε, για την υιοθέτηση των 580 εκατομμυρίων πιστώσεων προβλέπαμε ότι θα καλύπταμε το κόστος για το πρόγραμμα. Από την γραμμή για τον προπολογισμό πήγαμε στην επιχειρησιακή γραμμή για το, την πρώτη προκήρυξη διαγωνισμού. Στο μεταξύ, ο οργανισμός έχει αρχίσει να εφαρμόζει την ε, πρωτοβουλία. Ε, μιλάμε για ένα ποσό συνολικά 724.123 για να καλυφθούν τα επιπλέον ε, λειτουργικά έξοδα. 347.000 ευρώ καλύπτονται από το SFIC και 377 θα επιστραφούν από το Wi-Fi, από την επιχειρησιακή γραμμή αυτή. Περί αυτού πρόκειται. Έχουμε λάβει γραπτές παρατηρήσεις από την Κομισιόν σε όλες τις ερωτήσεις που είχαμε. Επομένως, συστήνω να ψηφίσουμε υπέρ της μεταφοράς αυτής, που είναι συνέπεια της υιοθέτησης της νομικής φάσης ε, για το Wi-Fi, για το πρόγραμμα της Ένωσης. Ψηφίσουμε. Αυτά τα Wi-Fi και μαλακίε. Εγκρίνεται. Ε, δύο αποχές, δύο ψήφοι κατά, 29 ψήφοι υπέρ. Εγκρίνεται. Πολύ ωραία. Και τώρα έχουμε μια ψηφοφορία για την ε, έδρα, τον καθορισμό της έδρας της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών. Έχουμε μια πρώτη τροπολογία. Τροπολογία υπαριθμών 9. Και την τροπολογία υπαριθμών 5. Τις ψηφίζουμε. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 1. Με μία προφορική τροπολογία του εισηγητή υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός υπαριθμών 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Θα το επαληθεύσουμε ε, ηλεκτρονικά, παρακαλώ. Ψηφίζουμε τώρα. Ψήφισαν όλοι. Πέρας προφορία. Εγκρίνεται. 19 ψήφι υπέρ, 13 κατά. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Για το σύνολο του κειμένου, όπως το τροποποίησαμε, με ονομαστική κλίση. Ψηφίζουμε τώρα ηλεκτρονικά. Πέρας εγκρίνεται με 28 ψήφους υπέρ, 4 ψήφους κατά και μία αποχή. Και τώρα, έκθεση ομάρζη για την εδαφική συνοχή, κοινωνική συνοχή και οικονομική συνοχή και για την 7 έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μάλιστα θα ήθελα να σας ε, τονίσω ότι σε ό,τι αφορά τον κατάλογο ψηφοφορίας που δόθηκε για αυτή την γνωμοδότηση, ε, θα ήθελα να σας ζητήσω να σημειώσετε τις εξή διευκρινήσεις. Καταρχάς, διάφορες χωριστές ψήφοι, ε, ψηφοφορίες ζητήθηκαν για τις παραγράφους που καλύπτονται από συμβιβασμού. Πρόκειται για τις τροπολογίες 6, 25 και 28. Δεύτερη διευκρίνηση, η τροπολογία 14 δεν είναι συμβατή με το συμβιβασμό υπαριθμών 2 και κατά συνέπεια καταπίπτει εάν ο συμβιβασμός αυτός υιοθετηθεί. Υπάρχουν σχόλια. Δεν βλέπω. Πολύ ωραία. Θα περάσουμε τώρα στην ψηφοφορία. Έχετε το λόγο. Να σας εξηγήσω ότι διάβασα το κείμενο και στην παράγραφο 1, εάν ο συμβιβασμός υιοθετηθεί, θέλω να αποσύρω την ε, τροπολογία 6 που είναι δική μου. Πολύ ωραία, την αποσύρατε την 6. Ευχαριστούμε. Θα κερδίσουμε και χρόνο. Για το συμβασμό 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9 με χωριστή ψηφοφορία, πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, θα το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε τώρα. Ψήφισαν όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με 18 ψήφους κατά, 12 ψήφους υπέρ. Για το δεύτερο τμήμα παρακαλώ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι είναι η ίδια κατάσταση όπως και για το πρώτο τμήμα. Απορρίπτεται. Τροπολογία 10. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβασμός 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στην τροπολογία 15 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 16, υπέρ, κατά, αποχές, θα το επαληθεύσουμε χρονικά. Ψηφίζεται τώρα. Πέρας φοφορίας. απορρίπτεται 17 ψηφί κατά, 14 ψηφί υπέρ και μία αποχή. Τροπολογία 17, υπέρ, κατά, αποχές θα επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίσουμε τώρα. Λήξη της ψηφοφορίας απορρίπτεται με 16 ψήφους κατά. Συμβιβασμός 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 25. Υπέρ. Κατά. Ε, ε, αποχές. Εγκρίνεται. Συμβασμός 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε στη τροπολογία στο συμβασμό 6 Υπέρ. Κατά. Οι αποχές εγκρίνεται. Περνάμε λοιπόν στο δεύτερο μέρος της τροπολογίας 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα επαληφθέσουμε ηλεκτρονικά για το δεύτερο κομμάτι του, της Υπολογίας ε, 28, έναρξη της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με 19 ψήφους κατά. Ε, τροπολογία 31. Υπέρ κατά. Αποχές. Ε, απορρίπτεται. Τροπολογία 32 με δύο τμήματα. Για το πρώτο κομμάτι υπέρ. Κατά ηλεκτρονική επαλήθευση, έναρξη της ψηφοφορίας. Πέρασε της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με 18 ψήφους ε, κατά δεύτερο τμήμα. Αν καταπίπτει το πρώτο κομμάτι, καταπίπτει και το δεύτερο. Τροπολογία 33 λοιπόν, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται τροπολογία 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται για το σύνολο του κειμένου με ονομαστική ψηφοφορία έναρξη της ψηφοφορίας πέρας εγκρίνεται με 29 ψήφους υπέρ 4 ψήφους ε, κατά ε, συγχαρητήρια σε ό,τι αφορά τα άλλα κομμάτια. Δεν υπάρχει αίτημα μεταφοράς. Δίνω λοιπόν το λόγο στην Μόνικα Αλμέγερ. Σε ό,τι αφορά τα διάφορα ε, σχέδια κτηριακής πολιτικής και, κυρίως, και πρώτα απ' όλα τη μεταφορά του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων στο Άμστερνταν. Κύριε Πρόεδρε, προτείνω να ξεκινήσουμε με τα πιο εύκολα και μετά να ολοκληρώσουμε με τα πιο δύσκολα. Ε, γιατί άμα ξεπετάξουμε τα εύκολα μετά θα έχουμε χρόνο για συζήτηση. Αυτό που είναι λοιπόν αρκετά απλό, εκνευρίζει βέβαια, αλλά αυτό που είναι απλό είναι το σπίτι της Ευρώπης στη Στοκχόλμη παρά την ε, έρευνα που έγινε στην ε, αγορά, γιατί στη Στοκχόλμη υπάρχει μια ευημερούσα αγορά στα κτίρια. Ήταν πολύ δύσκολο να βρούμε ένα κτίριο το οποίο να μας ικανοποιεί και να ικανοποιεί και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε αναγκασμένοι το κτίριο που έχουμε τώρα να παρατείνουμε τη μίσθωσή του για τρία χρόνια και μετά ίσως να έχουμε την ευκαιρία να βρούμε κάτι πιο κατάλληλο, κάτι καινούριο. Το κόστος ε, είναι υψηλότερο από ότι καθότι τα νίκια αυξήθηκαν κατά πολύ στη Στοκχόλμη. Και έτσι λοιπόν η αύξηση που βλέπετε δεν είναι πάνω από την αύξηση της αγοράς, είναι κάτω από την αύξηση της αγοράς, αλλά παρόλα αυτά περισσότερα χρήματα από ό,τι πληρώνουμε μέχρι ε, σήμερα. Η Κομισιόν αναλαμβάνει τις 681 περίπου χιλιάδες και το Κοινοβούλιο περίπου τις 464 χιλιάδες. Εγώ δεν βλέπω να υπάρχει πρόβλημα, γι' αυτό και παρακαλώ να συνενέσετε. Ευχαριστώ πολύ. Donc, euh, Μας παρουσιάσατε λοιπόν το ε, κομμάτι που αφορά τη Στοχόλμη. Θέλετε να ψηφίσουμε τώρα, ναι, για τη Στοχόλμη. Ε, θετική ε, τοποθέτηση της εισηγητή. Ε, γίνεται ηλεκτρονική ψηφοφορία, έναρξη. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται με 25 ψήφους ε, υπέρ, 3 ε, κατά και 2 αποχές. Το Άμστερνταμ. Για την Κένια έχουμε 4 κομμάτια, στα πούμε. Ε, για την Κένια έχουμε ήδη μια πρωτοπληροφορία που πήραμε από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Ως εκ τούτου αυτά που μας προτείνονται δεν διαφέρουν και πολύ από αυτά που μας είχαν δοθεί στην ενημέρωση. Εκτός τότε έχουμε τώρα κάποιες περισσότερες ε, λεπτομέρειες το, η συνολική έκταση είναι περίπου 4.000 τόσα τετραγωνικά μέτρα. Αυτό το κτίριο το μοιράζεται η Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία, η ΙΜΠΕ ε, και άλλοι ε, αναλόγως τα ε, κατανεμηθούν και οι θέσεις, πάσκευση, οι θέσεις στάθμευσης, γιατί εκεί συμμετέχουν πάρα πολλοί, η Unifor, η ΕΙΜΕ, πάρα πολλοί σε 33 τετραγωνικά μέτρα ανάτομο και το ετήσιο μίστημα είναι περίπου 600 τόσες ε, χιλιάδες με τη αριθμική προσαρμογή του 3%. Αυτό το βρίσκω λίγο πρόβλημα, αλλά ξέρετε στο Ναϊρόμπι δεν υπάρχουν ε, πολλές ε, δυνατότητες ε, να βρει κανείς κάτι άλλο που να του αρέσει. Και το κτίριο αυτό καλύπτει τις ε, προϋποθέσεις, υπάρχει κυρίως καλύτερη ασφάλεια και όπου υπάρχει καλύτερη ασφάλεια μειώνεται και το κόστος ασφάλειας, ως εκ τούτου αξίζει τον κόπο να ενοικιάσει κανείς αυτό το κτίριο. 2,6 εκατομμύρια είναι το κόστος εξοπλισμού και 13.000 ε, περίπου είναι το κόστος ε, της μετακόμισης, υπάρχει και ένα κόστος για τους συμβολογράφους, για ανακαινήσεις. Ως εκ τούτου θεωρώ ότι το ετήσιο συνολικό κόστος, αν τα υπολογίσει κανείς όλα είναι 1,7 περίπου εκατομμύρια ευρώ. Σας προτείνω να συμφωνήσετε γιατί το όλο σχέδιο όχι μόνο είναι λογικό αλλά έχουμε ενημερωθεί και σωστά από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Ευχαριστώ πολύ για αυτές τις διευκρινήσεις. Ε, είστε υπέρ αυτής της, ε, του, αυτού ε, της επιχείρησης στη Κένια, κύριε Ντεμπρέ. Μία ερώτηση προς τη συνάδελφο. Βλέπουμε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης έχει στη διάθεσή της γραφεία ε, ε, ε, με 4.000 περίπου 200 τετραγωνικά και υπάρχουν άτομα από την UNAFOR, από την ομάδα για το κέρδος της Αφρικής και τώρα θέλουμε ένα καινούριο κτίριο 15.000 τετραγωνικών. Πολλαπλασιάζουμε την επιφάνεια επί δηλαδή. Θα ήθελα να ξέρω αν αυτό δικαιολογείται από ε, συμφωνίες που έχουν ήδη συναφθεί με άλλες υπηρεσίες που θα μπορούσαν να καλύψουν ένα μέρος του ενοικίου γιατί πολλαπλασιάζουμε την ε, επιφάνεια επί τρία. Δεν είμαι κατά, αλλά θέλω να ξέρω αν υπάρχουν ε, συμφωνίες που έχουν συναφθεί με άλλους θεσμούς για να δικαιολογηθεί μια τέτοια αύξηση. Δεν ξέρω αν ο εισηγητή έχει αυτές τις πληροφορίες, θα ήθελα να γνωρίζω τι συμβαίνει ακριβώς. Κοιτάξτε, περίπου 4.000 είναι τα τετραγωνικά μέτρα. 4.200 κάτι. Και έχουν... Εκεί βρίσκονται η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και έχουμε συνάψει και συμβάσεις με τους υπόλοιπους ε, για το τι χώρο θα καταλάβουν εκείνοι. Άρα δηλαδή ε, τον χώρο αυτό το μοιραζόμαστε. Έχουμε τώρα περισσότερους συνεργάτες εκεί, η Κομισιόν έχει 84, έχουμε άλλους 9 από τις αντιπροσωπείες, από τη Σομαλία, και από διάφορους άλλους φορείς, 2-10 συνεργάτες, 33,11 τετραγωνικά μέτρα ανάτομο. Δηλαδή, αν θέλετε, ο μέσος όρος. Ο μέσος όρος αυτού που συνηθίζεται και μάλιστα και κάτω από το μέσο όρο ε, που προβλέπεται για τις ε, αντιπροσωπείες. Μπορείς να επαναλάβεις γιατί δεν άκουσα τι είπες. Συμφωνώ μόνικα με αυτό που είπες τώρα μόλις. 84 υπάλληλοι, άτομα από την αντιπροσωπεία για τη Σομαλία, αλλά αυτοί βρίσκονται σε ένα κτίριο αυτή τη στιγμή 4.200 τετραγωνικών. Και τώρα ζητάμε ένα κτίριο 15.000 τετραγωνικών. Όχι. Είναι τεράστιο ε, κτίριο, το οποίο όμως δεν ε, χρησιμοποιούμε εξ ολοκλήρου. Θα νοικιάσουμε τέσσερις ορόφους. Τα υπόλοιποι όροφοι δεν θα είναι δικοί μας. Θα χρησιμοποιήσουμε 4.372 τετραγωνικά, έτσι δεν είναι. Κοιτάξτε, πρόκειται για το εξής. Ε, τέσσερις ε, ορόφους του νέου κτηρίου θα τους ε, προσφέρουμε δεν θέλουμε να έχουμε όλο το κτίριο, μόνο τέσσερις ορόφους. Και αν υπάρξουν περισσότερες ανάγκες, ε, αυτό θα πρέπει να μας το πει η υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Μέχρι τώρα μιλάμε για τέσσερις ορόφους ε, από τους 20. Τους υπόλοιπους ορόφους δεν τους θέλουμε. Θα νοικιάσουμε ε, αυτά τα 4.300 τετραγωνικά. Ναι τους τέσσερις αυτούς ορόφους. Ε, οι υπόλοιποι όροφοι ανήκουν σε άλλον. Εντάξει. Ηλεκτρονική ψηφοφορία θα γίνει. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται με 27 ψήφους υπέρ, 3 κατά και 2 αποχές. Θα μιλήσουμε επιτέλους για το Άμστερνταμ. Ναι. Ναι, θα μιλήσουμε για το Άμστερνταμ. Αξιότιμε Πρόεδρε, τώρα λοιπόν θα μιλήσουμε για το Άμστερνταμ. Έχω και εγώ να κάνω κάποιες ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, την τελευταία φορά είχα σκίσει κριτική στην Ολλανδική κυβέρνηση και πρέπει να σας πω ότι εντωμεταξύ η κατάσταση έχει βελτιωθεί κατά πολύ. Ε, ισχύει το εξή λοιπόν. Πρώτον, έχουμε ένα φάκελο που μας έχει κατατεθεί και ο φάκελος αυτός ε, είναι αυτά που προτείνει η Ολλανδική κυβέρνηση στους ε, συνεργάτες της. Δηλαδή, η Ολλανδική κυβέρνηση θα αναλάβει το κόστος μεταφοράς όσο και το κόστος του μεταβατικού κτηρίου. Επίσης, το κόστος για το νέο κτίριο στο βαθμό που ε, το κτίριο αυτό δεν πρέπει να ε, ανακαινιστεί ειδικά για μας. Κατόπιν τούτου 20 χρόνια θα είναι ε, ο χρόνος μίσθωσης και θα έχουμε και τη δυνατότητα παράτασης του μισθώματος και του μισθωτηρίου. Αν τελικά προκύψει κάποιο άλλο κόστος θα επιβαρύνει την Ολλανδική κυβέρνηση. Σας τα λέω όλα με πολλές λεπτομέρειες και οι δύο συμφωνούν, τα δύο αντισυμβαλόμενα μέρη συμφωνούν ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούν να καταγγείλουν τη σύμβαση. Ε, στο βαθμό παραδείγματος χάρη η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίζει να μετακομίσει κάπου αλλού. Στην περίπτωση αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, πρέπει να ειδοποιήσει έξι μήνες ε, νωρίτερα και βεβαίως μπορεί να υπάρξει και κάποια έκτακτη ανάγκη που καθιστά άκυρη τη σύμβαση. Ε, αυτό είναι απαραίτητο. Το έχουμε προσθέσει ο ρήτρα γιατί την τελευταία φορά είχαμε κάνει ένα μεγάλο λάθος ε, και δεν είχαμε τη δυνατότητα καταγγελίας της σύμβαση και ήμασταν αναγκασμένοι να καλύπτουμε εμείς το κόστος ή να βρούμε έναν υπενικιαστή. Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Το 2019 είναι το έτος ε, ενέγερση 15 Δεκάτου του 19 θα μπούμε μέσα αν καθυστερήσουμε το κόστος θα, το αναλάβει η Ολλανδική κυβέρνηση 31.000 περίπου τετραγωνικά ε, μέτρα θα είναι η έκταση 26.000 περίπου για τα γραφεία 5.000 ε, περίπου τετραγωνικά μέτρα συνεδριακό κέντρο ε, χωρίς στάθμευσης Επίσης προβλέπεται το κτίριο μπορεί κανείς ε, να το προσπελάσει και με ε, δημόσια μέσα μεταφοράς. Αυτή τη στιγμή 1103 είναι οι συνεργάτες που θα εγκαθισταθούν εκεί. Εν τω μεταξύ η Ολλανδική κυβέρνηση έχει πάρα πολλούς συνεργάτες που έχουν οικογένεια και παιδιά και γι' αυτό το λόγο έχει κάνει μια επιπρόσθετη προσφορά, δηλαδή να βοηθήσει στα σχολεία, στους χώρους στάθμευσης, που σημαίνει ότι στην περίπτωση ελληνική κυβέρνηση καλύπτει πλήρω τι απαιτήσει μα. Κατά τα άλλα, αν οι συνάδελφοι έχουν πάρει κάποιε άλλε πληροφορίε, εγώ να σα πω ότι δεν έχω πάρει άλλε πληροφορίε. 28,5 περίπου τετραγωνικά μέτρα η έκταση ανά άτομο, κάτω δηλαδή από το μέσο όρο, κάτω από αυτό που κατ' ουσίαν απαιτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και 8,668 880 είναι ε, το πραγματικό κόστος ε, το κόστος συντήρησης είναι 1,8 εκατομμύρια, 1,2 ε, εκατομμύρια για το κτίριο και κατά τα άλλα 650.000 για άλλα, άλλες εργασίες συντήρησης. 320 ευρώ ε, αυτό συμπεριλαμβανόταν στη συντήρηση και νομίζω ότι αυτό τώρα είναι πλέον το ε, κόστος το οποίο μας αφορά. Οι λειτουργικές δαπάνες 3,141. Αυτό βέβαια πρέπει να το καλύπτουμε εμείς για την καθαριότητα και την ασφάλεια. Καλύπτουμε επίσης τις δαπάνες για το φυσικό αέριο και για το ηλεκτρικό ρεύμα 13,67 είναι το πραγματικό κόστος και ενδιάμεσα υπάρχουν και άλλες δαπάνες τις οποίες οφείλουμε να αναλάβουμε εμείς και δεν ήταν αντικείμενο του διαγωνισμού. Η ΕΜΑ είναι ένας οργανισμός ο οποίος σε μεγάλο βαθμό αυτοχρηματοδοτείται. Ως εκ τούτου η ΕΜΑ, ο οργανισμός αυτός, ε, θα έχει 15 εκατομμύρια για την ε, κατασκευή, ένα κομμάτι θα το καλύψει μόνη της, ε, το μισθωτήριο συμβόλαιο θα είναι περίπου 20 έτη. Αυτά όλα λοιπόν σημαίνουν ότι αν συνυπολογίσει κανείς το σύνολο των ταπανών με catering, με ασφάλεια, με έπιπλα, εσωτερική, εσωτερικό εξοπλισμό, βίντεο και οτιδήποτε άλλο, 14,37 εκατομμύρια, από τα οποία βέβαια ένα μεγάλο κομμάτι καλύπτεται από τον ίδιο τον οργανισμό αίμα. Ως εκ τούτου θεωρώ θεωρώ ότι δεν προκύπτει επιπρόσθετη επιβάρυνση του προπολογισμού. Το κτίριο αυτό είναι πολύ πιο ευνοϊκό από το ε, κτίριο του Λονδίνου. Ως εκ τούτου θεωρώ ότι με αυτά τα οποία μας προσφέρονται μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι. Έχω όμως και τρία βασικά ερωτήματα και έχω ήδη επισημάνει Κομισιόν ότι θα θέσω αυτά τα τρία ερωτήματα. Το πρώτο ερώτημα είναι το εξής. Θα υπάρξει αυτή η διαδικασία ε, όπου η Ιταλία θα καταφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και έχουμε δικαιολογημένες ερωτήσεις των σκιωδών εισηγητών. Ε, μπορεί λοιπόν να συμβεί όλο το θέμα να αναβληθεί εκ νέου. Θα ήθελα να επισημάνω στους συναδέλφους ότι με τη νέα ρήτρα περί καταγγελίας ε, της σύμβοσης αυτό πια δεν μπορεί να συμβεί. Δηλαδή δεν θα παραμείνουμε στο κτίριο αυτό αν είμαστε αναγκασμένοι να φύγουμε. Αυτό που είχαμε ως πρόβλημα στην αίμα δεν θα επανεμφανιστεί. Μάθαμε το μάθημά μα. Όμως η παράκλησή μου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας ανακοινώσει ποιες είναι οι νομικές συνέπειες ή ποιες θα μπορούσαν να είναι οι νομικές συνέπειες από μια τέτοια διαδικασία, ε, τι ακριβώς ε, προβλέπεται για τους συναδέλφους. Οικονομικές ε, συνέπειες για το κτίριο δεν θα υπάρξουν, διότι όπως σας είπα έχουμε τη ρήτρα της καταγγελίας. Δεύτερο, seat agreement και τρίτο, τροπολογία των ε, Founding Regulation ε, που αυτή τη στιγμή τις ε, διατάξεις αυτές εξετάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος. Ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να μας δώσει, παρουσιάσει μια γενική εικόνα γιατί με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να αποφασίσουμε με μεγαλύτερη ασφάλεια. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Ολιβιέ Σάλ θα ήθελε να απαντήσει ερωτήσεις της παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ. On the, uh, on, on the, on the court case, uh, Για την περίπτωση του δικαστηρίου, δεν είναι κάτι το οποίο η Κομισιόν uh, έχει λόγο. Είναι μια διαδικασία ανάμεσα στις Ιταλικές Αρχές και το Συμβούλιο. Χρήσιμο θα ήταν να υπενθυμίσουμε λοιπόν ότι αυτό απορρέει από το περίεργο πλαίσιο μέσα στο οποίο ξεκίνησε η διαδικασία. Μιλάμε για την, ε, με την κατάσταση ενός οργανισμού που είναι κάτι διαφορετικό από την κλασική διαδικασία, όταν δημιουργείται δηλαδή ένας νέος οργανισμός, ένας νέος φορέας. Και όπως ξέρουμε όλοι, με βάση τη διαδικασία η οποία εγκρίθηκε από τα κράτη-μέλη την περασμένη άνοιξη και τις διάφορες προσφορές ε, που προέκυψαν από τις πρωτεύουσε, τα διάφορα τα 27 κράτη-μέλη έφτασαν σε πολιτική συμφωνία τον Νοέμβριο του 2017 για τις δύο νέες έδρες. Και εκεί το νομικό κείμενο που υποβλήθηκε από την Κομισιόν αποκτά αξία, γιατί αυτή η πολιτική συμφωνία πρέπει να επιβεβαιωθεί μέσω ενός νομικού κειμένου. Γι' αυτό η Κομισιόν υπέβαλε τις δύο προτάσεις πέρυσι τον Νοέμβριο του 2017, δηλαδή τροποποιώντας την έδρα για τον ιδρυτικό κανονισμό για την ε, EMA και το, την EBA, την Τραπεζική Αρχή και την Αρχή Φαρμάκων. Η Ολομέλεια ψήφισε την α, ε, περασμένη εβδομάδα ε, έκθεση Λαβιόλα για την ΕΜΑ και επιβεβαίωσε την τροποποίηση, την αλλαγή της έδρας της ΕΜΑ, δηλαδή στο Άμστερνταμ. Ο άλλος τρόπος για να, να επιβεβαιωθεί αυτή η πολιτική συμφωνία μέσω νομικού κινημένου είναι μια συμφωνία στην περίπτωση της ΕΜΑ έχει προχωρήσει η δουλειά πολύ καλά. Υπάρχουν έντονες συζητήσεις μεταξύ των Ολλανδικών αρχών και την ίδια την ΕΜΑ και περιμένουμε τελεσφόρηση των συζητήσεων τις επόμενες μέρες, οι εβδομάδες το πολύ. Και φυσικά η συμφωνία αυτή των πρωτεύουσών, εν θα επιβεβαιώσει τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν ήδη συμφωνηθεί και που απεικονίζονται επίσης και στο φάκελο. Το σημαντικό που πρέπει να τονίσουμε και να, για να απαντήσω και στην ερώτηση της ηγήτριας είναι ότι τα βασικά, ένα από τα βασικά στοιχεία που τα τρία θεσμικά όργανα προσπαθούν να εξασφαλίσουν είναι να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει συνέχεια των εργασιών της ΕΜΑ. Εξού και τρέχουν αυτές οι παράλληλες διαδικασίες. Ε, υπάρχει νομική τροποποίηση της ιδρυτικής πράξης, δηλαδή. Υπάρχουν οι συζητήσεις μεταξύ πρωτεύουσα και αίμα και υπάρχει και η ανάγκη να προχωρήσουμε γρήγορα πάνω στο ίδιο το φάκελο. Εξού λοιπόν και η προσπάθεια αυτή για να γίνουν τα απαραίτητα βήματα, ούτω ώστε να γίνει μια ομαλή με την κατάσταση. Ελπίζω αυτέ οι εξηγήσει να είναι επαρκεί για την Επιτροπή σα, ούτω ώστε να δώσει το πράσινο φω για το κτίριο τη ΕΜΑ, για το φάκελο αυτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο εκπρόσωπο τη ΕΜΑ θέλει να πάρει το λόγο. Παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν έχω να προσθέσω και πολλά στα όσα είπε ο εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι όλε οι πτυχέ ε, προοδεύουν καλά. Η συμφωνία για την έδρα, έχουμε κάποια ίσονα θέματα να επιλύσουμε, αλλά είναι θέμα ημερών για να επιληθούν. Έχουμε και αυτή την ε, steering committee με την ε, Ολλανδία, δηλαδή την ε, συνάντηση της Διευθύνουσας Επιτροπής με την Ολλανδία και θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα. Σε ό,τι αφορά τα, την προσωρινή έδρα, το προσωρινό κτίριο και όλες τις εργασίες που πρέπει να ξεκινήσουν για να ετοιμαστούν τα τελικά, η τελική έδρα, το τελικό κτίριο, πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν καθυστερήσεις και σε αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τις διευκρινήσεις σας. Λοιπόν, ο κύριος Γιώτη. Ο κύριος Βιώτη, παρακαλώ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Χολμάιρ για την ακρίβεια, για όλες τις λεπτομέρειες που μας έδωσε και που μελέτησε όλες τις συμβάσεις τόσο προσεκτικά για τις διάφορες έδρες, έτσι. Φυσικά, δεν θέλω να μπω τώρα στο θέμα της διαδικασίας αυτή με την Ιταλική κυβέρνηση καθόλου. Θέλω ε, για την, το, το, το μισθωτήριο συμβόλαιων. να κάνω τι εξής ερωτήσεις, Τρει ερωτήσει. Καταρχά, το χρόνο παράδοσης. Γιατί προβλεπόταν αρχικά για τον Οκτώβριο, 1η Οκτώβριο. Και τώρα μιλάμε για 15 Νοεμβρίου, έτσι, του 2019, παράδοση του κτηρίου. Ποια είναι η νομική βάση ε, επί της οποίας άλλαξε αυτή η ημερομηνία. Δεύτερον, υπάρχει ένα δεύτερο στοιχείο στο συμβόλαιο μεταξύ ΑΜΑ και κατοχωρών. Μιλάμε για 15 Νοεμβρίου, εκτός και αν ε, συμβεί κάτι έκτακτο, ας πούμε, εκτός ελέγχου. Ποιες είναι αυτές. Δύο είναι τα μέρη στην τελική. Είναι η αίμα και οι κάτω χώρε. Μιλάμε για φυσικέ καταστροφέ, απρόβλεπε κτλ. ή μιλάμε για καθυστέρηση από του εργολάβου που οφείλονται στο γεγονό ότι οι ίδιοι με καθυστερούν ή θα καθυστερήσουν. Και, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει σε περίπτωση καθυστερημένη παράδοση να υπάρχει κύρωση έτσι, για τον εργολάβο. Τρίτον, τρίτον, τελευταίο ερώτημα για μια ε, ρήτρα πιθανής ανανέωσης του ενοικίου. Κανονικά νοικιάζουμε για 20 χρόνια, έτσι. Το είπε και ε, η κυρία Χολμάιερ, ότι μπορεί να ανανεωθεί αυτόματα. Με βάση τα έγγραφα της ΕΜΑ, ε, δεν θα πρέπει κανονικά να αλλάξει η έδρα. Έχει προβλεφθεί μία ρήτρα για ε, να μην ε, αυξηθεί υπερβολικά το μίσθωμα μετά το, 2039. Έχει προβλεφθεί μια τέτοια ρήτρα παγώματος του μισθωτηρίου. Merci, Madame Κυρία Χόφμαν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, εγώ αυτό που με εντυπωσιάζει είναι το εξής. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε αποφασίσει διαφορετικά, αλλά βέβαια δεν μπορέσαμε να επηρεάσουμε την απόφαση. Και ερχόμαστε τώρα αντιμέτωποι με την κατάσταση όσο έχει διαμορφωθεί. Όμως υπάρχει κάτι που δεν έχω καταλάβει και γι' αυτό ερωτώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πώς ακριβώς ε, αξιολογεί της, ε, την πιθανότητα η Ιταλία να δικαιωθεί στην προσφυγή της ε, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και ποιες θα μπορούσαν να είναι οι συνέπειες που θα προκύψουν από αυτό το ενδεχόμενο. Παρακαλώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τοποθετηθεί ακριβώς επ' αυτού. Πριν να δώσουμε το λόγο στην Κομισιόν, ποιος θέλει το λόγο, υπάρχει άλλος θέλει το λόγο, η Κομισιόν. Η κυρία Χολμάιερ νομίζω θέλει το λόγο. Το θέλετε? Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα για άλλη μια φορά να απευθυνθώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξέρω ότι δεν μπορείτε να πείτε ποια θα είναι η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, όμως σας ερωτώ, η διαδικασία ήταν νομότυπη, ήταν σωστή. Μιλήσαμε στο τηλέφωνο και εσείς μας είπατε με ανάγλυφο τρόπο ότι τα κράτη-μέλη συμφώνησαν για τη διαδικασία, ακολουθητέα διαδικασία ε, την, ε, το φθινόπερο. Αυτό είναι και μία απάντηση προς τον κύριο Γιώτη. Κοιτάξτε, αν καθυστερήσουν δεν θα υπάρξει πρόβλημα, γιατί από τον Νοέμβρη είναι η Ολλανδική κυβέρνηση, από την 1η Ιανουαρίου ήδη μάλιστα, ε, η οποία έχει αναλάβει το κόστος για το μεταβατικό κτίριο, που σημαίνει αν μας παραδώσουν το κτίριο Νοέμβρη ή Δεκέμβρη δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, γιατί έτσι και αλλιώ θα πληρώσει η Ολλανδική κυβέρνηση ανεξάρτητα με το πότε θα γίνει η μετακόμιση. Βέβαια θέλουμε και η Ολλανδική κυβέρνηση επιθυμεί διακαώς να γίνει μετακόμιση το συντομότερο δυνατόν διότι αυξάνεται το κόστος. Ως εκ τούτου, ε, παραλαμβάνω, η ίδια η Ολλανδική κυβέρνηση επιθυμεί να γίνει η μετακόμιση το συντομότερο δυνατόν. Για μας στον προπολογισμό δεν προκύπτει καμία τους δαπάνη διότι σας είπα τα αναλαμβάνει όλα η Ολλανδική κυβέρνηση. Μετά, έκπτωση ενοικίου. 8,8110 αυτό θα είναι το ενίκιο υπάρχει βέβαια τη μαριθμική αναπροσαρμογή ε, που ε, κατανέμονται και επιμερίζονται σε 20 χρόνια άρα από το 3% πάμε στο 6% προβλέπεται μία μείωση και έτσι κάθε χρόνο θα υπάρχει μείωση του κόστους. Ως εκ τούτου και εδώ δεν υπάρχει πρόβλημα. Και το τελευταίο που θέλω να πω προς τη συνάδελφο την κυρία Χόφμαν. Θεωρητικά, αν το Συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά, εγώ δεν θέλω να κάνω εικασίες, αλλά τουλάχιστον αυτή τη φορά δεν θα έχουμε κτηριακό πρόβλημα. Γιατί μετά τους έξι μήνες μπορούμε να καταγγείλουμε τη σύμβαση χωρίς να κληθούμε να καταβάλουμε αποζημίωση. Αυτό δηλαδή που αναγκαστήκαμε να κάνουμε στο Λονδίνο. Γι' αυτό σας λέω πολύ πιο ήρεμα, ναι, έτσι είναι τα πράγματα, γιατί αν συμβεί κάτι δεν θα επιβαρυνθούμε. Αλλιώ θα προέκυπταν τεράστια προβλήματα. Θεωρητικά βέβαια δεν θα προκύψει πρόβλημα αν, ακούσατε, αν ακούσετε αυτά που μου είπε και εμένα χθε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο τηλέφωνο. Μόνικα, να ψηφίσουμε. Η Κομισιόν θα ήθελε να πει κάτι τελευταίο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στα ερωτήματα που τέθηκαν. Χωρίς να ξεκινήσω καινούρια συζήτηση, όπως είπα προηγουμένως, τα κράτη-μέλη συμφώνησαν το προηγούμενο καλοκαίρι μια διαδικασία και όπως γνωρίζουμε τηρήθηκε αυτή η διαδικασία. Σε ό,τι αφορά την προσφύγη των Ιταλικών αρχών δεν έχουμε να πούμε, δεν μας πέφτει λόγος σε μια υπόθεση που αφορά ένα κράτος μέλος και το Συμβούλιο. Αυτό που προσπάθησα να πω προηγουμένως είναι ε, σημαντικό να, να επικεντρωθούμε στην νομική σαφήνια διευκρίνηση που θα επιφέρει η τροποποίηση του κανονισμού και τα, ε, οι διευκρινήσεις για το ε, σχέδιο αυτό περιλαμβάνονται στο φάκελο. Από την πλευρά μας δεν προβλέπουμε κάτι το τρομερό, τουλάχιστον όχι σε ό,τι αφορά την προπολογισμό, ε, μετά από αυτή την προσοχή των Ιταλικών Αρχών. Ευχαριστώ κύριο Πρόεδρο. Κύριε Εισηγήτρια. Κύριε Πρόεδρε, προτείνω να αποφασίσουμε λαμβάντας υπόψη ότι θα ολοκληρωθεί σύντομα η συμφωνία για τις έδρες και λαμβάντας υπόψη ότι θα εγκριθούν, θα εγκριθεί και ο ο περίφημος κανονισμός Founding, Founding Regulation, γι' αυτό προέβηνε σε αυτή τη συμφωνία με τους εισηγητές. Ωραία. Θα ψηφίσουμε ερχονικά λοιπόν, μια και άλλο δεν θέλει το λόγο, ψηφίζουμε τώρα. Gut für Italien. Ψηφίστηκαν, ε, ψήφισαν όλοι. Πέρας, εγκρίνεται με 15 ψήφους υπέρ, 7 κατά, 6 εποχές. Τώρα, για τη Ουάσιγκτον. Θα ψηφίσουμε σήμερα ή θα το αναβάλουμε το θέμα αυτό. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να παρακαλέσω, επειδή το όλο θέμα μας εστάλει μόλις πριν από λίγο, θα έλεγα να ψηφίσουμε την άλλη φορά, στην επόμενη συνεδρία. Λογικά φαίνονται όλα αυτά, αλλά παρόλα αυτά δεν έχουμε ακόμα συγκεκριμένες πληροφορίες ε, για τη σύμβαση. Ε, δεν θέλω να πω τίποτα, μπορεί να είναι 20, μπορεί να είναι 30 χρόνια, τα ποσοστά μπορεί να κυμαίνονται. Εγώ θα ήθελα λοιπόν από κοινού με τους σκιώδης ηγητές να το ξαναδούμε λιγάκι και το θέμα της σύμβασης και γι' αυτό παρακαλώ για μία παράταση δύο εβδομάδων και να αποφασίσουμε στην επόμενη συνεδρίαση ε, της Επιτροπής. Ε. Ευχαριστώ πολύ. Θα κερδίσουμε χρόνο λοιπόν. Την επόμενη φορά θα συζητήσουμε αυτό το θέμα. Τελειώσαμε με τις ψηφοφορίες. Σε ό,τι αφορά την κτηριακή πολιτική, Λάβαμε πληροφορίες που μας επιτρέπουν να εξετάσουμε τα επόμενα σχέδια στο μέλλον ή η συγγήτρια θεωρεί ότι δεν υπάρχει λόγος να γίνει συζήτηση σήμερα. Κυρία Συγήτρια, τίποτα δεν θέλετε να προσθέσετε, όχι. Θα εξετάσουμε λοιπόν τώρα ε, οι ψηφοφορίες έχουν λήξει και τώρα θα εξετάσουμε το θέμα που αφορά τον Οργανισμό για την ε, Ασφάλεια στο, στο κυβερνοχώρο. Ο εισηγητής δεν είναι παρόν, άρα ο κύριος Τυριοβίλκεν θα τον εκπροσωπήσει και θα παρουσιάσει το σχέδιο ψηφίματος. Κύριε Βόλκεν. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι, σήμερα αντικαθιστώ τον κύριο Γκάια, ο οποίος δυστυχώς έπρεπε να παραμείνει στην εκλογική του περιφέρεια. Ε, θα είμαι γρήγορος και σύντομος. Όπως ξέρετε, ο οργανισμός ΕΝΙΖΑ, ο οργανισμός για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, που αυτή τη στιγμή έχει έδρα στην Ελλάδα, διοικητικά βρίσκεται η έδρα της στο Ηράκλειο, αλλά η πραγματική λειτουργική έδρα είναι στην Αθήνα. Ε, υπάρχει μία πράξη περί κυβερνοασφάλειας και η Κομισιόν προτείνει να υπάρξει βελτίωση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Ως εκ τούτου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ένα σύστημα πιστοποίησης ε, και Κατόπιν τούτου ε, θα πρέπει ε, σε αυτό το πλαίσιο να συμμετέχει και ο ΕΝΙΖΑ. Η ενίσχυση του ρόλου του ΕΝΙΖΑ είναι ευκταία, τη χαιρετίζουμε και επίσης χαιρετίζουμε και το ότι προβλέπεται να προσληφθούν περισσότεροι υπάλληλοι. Μέχρι το 2020 ο οργανισμός ε, θα αποκτήσει 23 εκατομμύρια ευρώ και θα έχει 80 υπαλλήλους, το διπλάσιο αριθμό. Με αυτή τη νέα ε, εντολή θα τεθεί βέβαια και το θέμα της έντρας της, ε, του οργανισμού εκ νέου. Και αυτό για τον εξής λόγο, διότι έχει δύο έντρες. Αυτό δεν είναι παραγωγικό. Η, το σχέδιο της γνωμοδότησης προβλέπει η συμφωνία περί ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και τον οργανισμό να αναθεωρηθεί και μετά την αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί ε, κάλεσαν ε, σύσταν μια ειδική ομάδα εργασία ε, και ε, λένε ότι θα πρέπει να αξιολογηθούν αυτοί οι οργανισμοί. Μια τέτοια αξιολόγηση ε, κατ' ουσίαν θα καταλήξει, είμαστε σίγουροι, στο ότι οι δύο έδρες είναι αντιπαραγωγικό. Επίσης υπάρχει μια πρόταση για να προβλέπονται ιδιαίτερα κονδύλια για την έρευνα, έτσι ώστε στο μέλλον ο οργανισμός να μπορεί να διεξάγει τι δικές της έρευνε και να μπορεί επίση και να προσφέρει εμπειρογνωμοσύνη. Κατά τα άλλα προτείνεται και η ε, συμπερίληψη ενός εκπροσώπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Διοικητικό Συμβούλιο. Κατά τα άλλα, ο οργανισμός θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να καταφεύγει για μεταφράσεις και σε άλλους παρόχους, αν αυτή είναι πιο φτηνή. Αυτά από τον κύριο Γκάια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που αντικαταστήσατε τόσο αποτελεσματικά το Hans ε, Γκάιερ. Κύριε Όλμπριχτ, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μία πολύ σύντομη παρατήρηση εκ μέρους του κυρίου Σαλαμάνκου, που έπρεπε να φύγει από το Κοινοβούλιο σήμερα. Ο κύριος Σαλβαμάρ, συγγνώμη, ευχαριστεί τον κύριο Γκάιερ για τη γνωμοδότησή του και συμμερίζεται τα περισσότερα στοιχεία της. Θέλει να τονίσει τη σημασία της, ε, ενός προϋπολογισμού που θα βασίζεται στις επιδόσεις. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχουν συνέργειες και ενισχυμένη συνεργασία με του ΕΝΙΣΑ, με άλλες ε, υπηρεσίες, φορείς, ε, οργανισμούς, χωρίς να δημιουργούνται επικαλύψεις με τους κρατικούς εθνικούς φορείς. Αυτή είναι η βασική παρατήρηση του συναδέλφου. Και εγώ ευχαριστώ. Υπάρχουν άλλες ε, παρατηρήσεις. Όχι, από ό,τι βλέπω. Ο εισηγητής. Μετά από αυτά που είπε ο κύριος Όλμπριχτ, έχει να πει τίποτα. Όχι. Αν δεν υπάρχουν σχόλια θα κλείσουμε αυτό το σημείο. Να σας πω ότι η ημερομηνία για την κατάθεση τροπολογιών είναι 28 Μαρτίου στις 12 η ώρα. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή Προϋπολογισμών θα γίνει στις 16 Μαΐου και στην Ολομέλεια του Ιουνίου στο Στρασβούργο θα αποφανθεί το Κοινοβούλιο για την γνωμοδότηση αυτή. Πολύ ωραία. Και τώρα θα υποδεχτούμε τον κύριο, κύριο Ιαν Γκρέγκορ που είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Παρακαλώ να έρθει στο βήμα. Σας ευχαριστώ που ήρθατε μαζί μας. Θέλετε να μας Ήρθατε εδώ και να μας παρουσιάσετε το έγγραφο που υιοθέτησε στις 15 Φεβρουαρίου το ελεγκτικό συνέδριο με τίτλο «Το μέλλον των οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταρρύθμιση της λειτουργίας του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να μια πρόταση η οποία πηγαίνει, είναι αντίστοιχη με τις δικές μας κατευθυν, ε, ανησυχίες. Γιατί έχει κάποιες ιδιαιτερότητες ο προϋπολογισμός της Ένωσης σε σχέση με τις βασικές αρχές ενός προϋπολογισμού. Ως συνήθως ο κ. Γκρέγκορ παρουσίασε την ε, έκθεση αυτή στην Επιτροπή Κοντ το Φεβρουάριο και στο μεταξύ η Επιτροπή μας και η Ολομέλεια υιοθέτησαν τη θέση του Κοινοβουλίου για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο καθώς και για τους ίδιους πόρους και επομένως καλώ τον κύριο Γκρέγκορ να πάρει το λόγο. Έχουμε μια ωρίτσα στη διάθεσή μας. Θέλω να τελειώσουμε στις 12.30. Ε, Παρακαλώ έχει το λόγο. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο, Πρόεδρε. Αγαπητοί Ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι, να σας ε, υπενθυμίσω από την τελευταία φορά που ήρθα εδώ, έγινε το, ε, ήταν το 2004, ήταν η τελευταία μεγάλη, μάλλον η πρώτη μεγάλη διεύρυνση. Έκτοτε δεν έχω ένθει στην Επιτροπή σας. Σήμερα θα ήθελα λοιπόν να σας παρουσιάσω αυτό το ενημερωτικό έγγραφο του ελληνικτικού Συνεδρίου για το μέλλον του Πουδουπού. Το μέλλον των οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ουσιαστικά. Θα ήθελα να διατρέξω λοιπόν αυτές τις διαφάνειες. Ε, τι κάναμε στο μεταξύ στις 15 Φεβρουαρίου, ε, όπως σας είπαμε, ε, ετοιμάσαμε ένα σύντομο ενημερωτικό έγγραφο, το πρώτο ενημερωτικό έγγραφο. Το επόμενο θα το δημοσιεύσουμε τον Ιούνιο-Ιούλιο του 2018. Αυτή τη στιγμή ε, ε, δημοσιευθεί και η πρόταση της Κομισιόν. Ελπίζουμε που θα έχει δημοσιευθεί το Μάιο. Στο μεταξύ, έχουμε δημοσιεύσει ή θα δημοσιεύσουμε ακόμα τρία έγγραφα για το μέλλον του προπολογισμού. Ένα για το μέλλον της ΚΑΠ, ένα ενημερωτικό κείμενο για το μέλλον της κοινή γεωργικής πολιτικής, ε, που έχει δημοσιευθεί σήμερα το πρωί. Του επόμενου μήνε θα δημοσιεύσουμε ένα άλλο ενημερωτικό έγγραφο για την απλούστευση στον τομέα της ε, πολιτικής συνοχής. Ίσως να έχει δημοσιευθεί ήδη τώρα, πριν από κανένα μισάωρο μάλιστα, θα το δημοσιεύαμε, η απλούστευση των προγραμμάτων έρευνας και κοινοτομίας, επίσης άλλο ενημερωτικό κείμενο. Και τέλος, το δεύτερο εξάμεινο του 18 θα δημοσιεύσουμε μία γνωμοδότηση για την απόφαση για τους ίδιους πόρους και άλλες τομεακές νομοθεσίες για τα προγράμματα δαπανών. Για τους ελεγκτές είναι πάντα δύσκολο να παρουσιάζουμε ένα έγγραφο για το μέλλον με βάση την παρελθούσα μας εμπειρία. Προσπαθούμε όμως να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να δούμε τα καλά στοιχεία και χρησιμοποίησαμε δύο επιθεωρήσεις, κυρίως του 2014, για την καλύτερη χρήση των κοινωτικών κονδυλίων και για τα κενά και τις επικαλύψεις, καθώς και τις προκλήσεις στη διαχείριση και στα συστήματα ελέγχου. Ε, επίσης, έχουμε την ετήσια έκθεση του 2014, 2015 και 2016 και παραπέμπουμε και σε αυτές και χρησιμοποίησαμε ως σημείο αναφορά 16 ειδικέ εκθέσεις του 2015, 16, 17 και 18 καθώ και διάφορε άλλε νομοδοτήσει για του ε, δημοσιονομικού κανονισμούς, διάφορες νομοδοτήσει για του ίδιου πόρου, η απόφασή μα για τον, κανονισμό, τον κοινό κανονισμό ε, για την πολιτική συνοχή και τέλο, και σημαντικό κάνω και μια αναφορά στο ενημερωτικό μα έγγραφο για την ενδιάμεση αναθεώρηση του Πουδουπού. Προσπαθήσαμε λοιπόν μέσα αυτό το ενημερωτικό έγγραφο να εστιάσουμε σε ένα τμήμα του έγγραφου προβληματισμού της Κομισιόν που είναι το τμήμα για το μέλλον του προπολογισμού της Ένωσης και πώς θα λειτουργεί. Το σημείο 4,2 στο ενημερωτικό έγγραφο της Κομισιόν, αν δεν απατώμε. Και φυσικά υποστηρίζουμε την Κομισιόν, γιατί πάντα είναι λίγο δύσκολο και λεπτό να συμφωνήσουμε για το μέλλον των οικονομικών μας. Είναι μια λεπτή ισορροπία ανάμεσα στις ισχύουσες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις νέες προκλήσεις, τις εθνικές προτεραιότητες και την ε, ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, να λάβουμε υπόψη τους κανόνες για, τους, για τις δαπάνες και να είμαστε στοχευμένοι στα αποτελέσματα ανάμεσα στις επιχορηγήσεις και στα υπόλοιπα οικονομικά ε, μέσα χρηματοδότησης. Ε, σε όλους τους τομείς. Μεταξύ των προκλήσεων έχουμε την πιθανή αποχώρηση ενός κράτους μέλους που μας δημιουργεί επιπλέον δυσκολίες, πέρα από τις δυσκολίες που έχουμε συνήθως. Στην επόμενη διαφάνεια προσπαθούμε να αναγνωρίσουμε τις ε, καλές αρχές οι οποίες αναφέρονται από την Επιτροπή στο έγγραφο προβληματισμού της και προσπαθούμε να αναλύσουμε και να τις αντιμετωπίσουμε σε όλες τις φάσεις του δημοσιονομικού κύκλου. Θα σας ε, κατευθύνω λοιπόν στον τομέα της πρότασής μας. Για την προστιθέμενη αξία. Δεχόμαστε αυτό που λέει η Κομισιόν να υπάρχει ε, ως βασικός στόχος η ευρωπαϊκή η ενωσιακή, αν θέλετε, προσθέμενη αξία και να εστιάσουμε τον προπολογισμό μας στη, στους τομείς με την υψηλότερη προσθέμενη αξία και να μειώσουμε τις εγγύησεις και τα χρηματοδοτικά μέσα τα υπόλοιπα. Για την ε, πρόταση 1, ε, το να βρούμε την ενωσιακή προσθέμενη αξία, σε κάποιο βαθμό εδώ απεικονίζουμε το άρθρο 52, μάλλον παράγραφη 52-56 της θέσης του Κοινοβουλίου για το μελλοντικό πουδουπού. Και προτείνουμε να εφαρμόσουμε διάφορα πράγματα για να εξασφαλίσουμε την ουσιακή προστιθέμενη αξία. Θα πρέπει να εντοπίσουμε ευκαιρίε για να χρησιμοποιήσουμε τον προπολογισμό σωστά, ούτως ώστε να δημιουργηθεί αυτή η προστιθέμενη αξία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και να αξιολογήσουμε τις ε, προτάσεις για πιθανό ενωσιακό, ενωσιακή προστιθέμενη αξία για τα νέα προγράμματα δαπανών. Επίσης, να αναπτύξουμε περαιτέρω το, ένα πλαίσιο όπου θα μετράμε τις επιδόσεις των προγραμμάτων ε, δαπανών και παράλληλα πρέπει να αξιολογήσουμε τους κινδύνους καθώς και τα ωφέλη από τη χρήση των ενωσιακών οικονομικών μέσων και εργαλείων την έκθεση 19 ε, του 2016 την λαμβάνουμε υπόψη μας για τα χρηματοοικονομικά εργαλεία και θα πρέπει περιοδικά να αξιολογούμε την προσθέμενη αξία των διαφόρων α, ενωσιακών προγραμμάτων ως τμήμα ενός συνολικού πλαισ... Ε, μιας συνολικής αναθεώρησης των δημοσίων δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ενωσιακή προσθέμενη αξία επίσης βασίζεται στις προηγούμενες ε, γνωμοδοτήσεις, μία του 2010, Νομίζουμε ότι πρέπει να εστιάσουμε σε όλα τα τμήματα του, κύκλου, του δημοσιονομικού κύκλου, από την, το, το καθορισμό των προϊοτήτων, ε, ίδιους πόρους, μέχρι το κλείσιμο των προγραμμάτων. Και να δούμε κατά πόσο υπάρχουν αποτελέσματα. Επίσης σχολιάζουμε εν συντομία την καθαρή θέση, την καθαρή ισορροπία. Παράγραφος 51 ε, στην νομοδότησή μας. Για μας στηρίζουμε την ε, σύσταση της ομάδας υψηλού επίπεδου για τους ίδιους πόρους και υπάρχει ανάγκη να υπάρχει μεγαλύτερη ακρίβεια για τη σχέση κόστους-οφέλους για αυτή την καθαρι... Ε, σε αυτή την καθαρή θέση. Θα πρέπει ε, να απλουστεύσουμε αυτή την ιδέα της καθαρής θέσης, της καθαρής θέσης γιατί δεν είναι ξεκάθαρη θα πρέπει να πλουστεύουμε τον τρόπο με τον οποίο χορηγούμε τα κονδύλια στα κράτη-μέλη, αλλά επίση και ποια είναι τα πλεονεκτήματα από αυτό, και θα πρέπει να καταλάβουμε τα μη οικονομικά ωφέλη ποια είναι από την ε, συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευελιξία μέσα σε ένα σταθερό πλαίσιο το επόμενο. Το κείμενο τη Κομισιόν προτείνει να ξαναδούμε τι ε, διαφορετικέ πτυχέ του Πουδουπού ε, που καθορίζουν την ευελιξία, όπω τα δημοσιονομικά περιθώρια, τον αριθμό των τίτλων και τομέων, τη διάρκεια του MFF, του πολιτού δηλαδή του δημοσιονομικού πλαισίου και το πώ χρησιμοποιείται, η πρότασή μα είναι να βελτιώσουμε τον προπολογισμό τη Ένωση για να ανταποκρίνεται σε όλα αυτά. Ε, και αυτό ανταποκρά, ε, αντανακλά τη δική σας θέση. Βασιζόμαστε στο κεφάλαιο 2 της ετήσιας έκθεσης του 2016. Πιστεύουμε ότι θα... Εργαλεία ευελιξίας θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν κυρίως για πρόβλεπτα γεγονότα και πιθανά προβλήματα με τις ε, πληρωμές από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Και όχι να ασχολούμαστε με τις ε, απρόβλεπτες συνέπειες από καθυστερημένες πληρωμές. Επίσης, ε, υπάρχει ένα σύστημα αποθεματικών, ένα γενικό αποθεματικό με πιστώσεις και συγκεκριμένα αποθεματικά για κάθε τίτλο για να καλύπτουμε τα μακροπρόθεσμα, τις μακροπρόθεσμα υποχρεώσεις ε, δαπανών που σχετίζονται ε, με προγράμματα κτλ. Ε, πιθανές υποχρεώσεις, επίσης συγκεκριμένους κανόνες για τις μεταφορές από, τις, από το αποθεματικό στον υπολογισμό και μεταξύ των αποθεματικών. Πάμε τώρα στην πρόταση 3. Να εστιάσουμε σε ένα πιο πλήρες οικονομικό σχέδιο Παράγραφος 73 της εκδομοδής του Κοινοβουλίου, αυτό συνδέεται με αυτήν την παράγραφο, προτείνουμε λοιπόν το πουδουπού να συμπληρωθεί με ένα επιπλέον οικονομικό σχέδιο, το οποίο θα εστιάζει σε κάποιους ε, κινδύνους, ε, παραδείγματος χάρη ε, κάποιες ε, μεταβλητές ας πούμε, ε, υποχρεώσεις οι οποίες έχουν εκπληρωθεί, προχρηματοδότηση, υποχρεώσεις κτλ. Καθώς και προβλέψεις για πιο μακροπρόθεσμες πληρωμές. Προσπαθούμε να συγχρονιστούμε με την γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου και να τη λάβουμε υπόψη μα για να λάβουμε υπόψη και άλλε πηγέ χρηματοδότηση που θα χρησιμοποιηθούν για να εφαρμοστούν οι ενωσιακέ πολιτικέ από τα κράτη-μέλη, του διεθνεί οργανισμού και του ιδιωτικού φορεί. Και πιστεύουμε ότι αυτό το συνολικό ε, οικονομικό σχέδιο θα πρέπει να επικαιροποιείται ετησίως, ούτω ώστε οι σημαντικές αλλαγές στις ενωσιακές πολιτικές, ε, η πρόοδος στην εφαρμογή τους, οι αλλαγές κτλ. να ληφθούν υπόψη. Και αυτή η πρόταση βασίζεται κυρίως στο έγγραφο ενημέρωσης ε, για την ενδιάμεση αναθεώρηση του πουδουπού. Απλουστευμένοι κανόνες. Η Κομισιόν ε, το σκέφτεται πάρα πολύ καλά το έχει σκεφτεί πάρα πολύ καλά και μαζί λοιπόν θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το σύστημα πιο εύκολο στη διαχείριση, μειώνοντα τον αριθμό των προγραμμάτων δαπανών, των χρηματοδοτικών μέσων, να προστατεύσουμε του κανόνε, ούτω ώστε και στα έσοδα, να, σε περίπτωση που μπορούμε να σταματήσουμε του διορθωτικούς μηχανισμού ε, στον προπολογισμό τη Ένωση. Όπως σας ανέφερα προηγουμένως, ε, έχουμε ήδη καταθέσει κάποια άλλα έγγραφα που αφορούν στην απλούστευση. Πρόταση υπαριθμών 4. Είναι να ισχυθεί ε, το πλαίσιο της απόδοσης ε, και από αυτού θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο ε, για το ότι κάνει μνήμα του της ετήσιας έκθεσης του 2016 από εκεί αναφέρεται το θέμα της απόδοσης και θα ήθελα να επισημάνω ότι στόχος μας είναι να ε, περιοριστούν ε, οι δείκτες. Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 200 στόχους ε, και πάνω από 700 δείκτες για τις πολιτικές. Επειδή λοιπόν αυξάνεται ο αριθμό των προγραμμάτων δαπανών υπάρχει και ο κίνδυνος επικαλυψάρει, δηλαδή τίθεται η ανάγκη εξορθολογισμού. Επίσης θα ήθελα να επισημάνω ότι όταν συζητήσουμε συζητήσαμε για το κεφάλαιο υπαριθμών 4 ε, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκεί εστιάσαμε την προσοχή μας και στην ποιότητα των στοιχείων απόδοσης, στοιχεία τα οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει από τα κράτη-μέλη. Ε, Πάμε στην λογοδοσία, η οποία και αυτή καλύπτεται από το, ε, από το έγγραφο προβληματισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορά την ε, δημοκρατική και διαφανή διαδικασία στις αποφάσεις για τους μελλοντικούς προϋπολογισμούς. Κοινός στόχος είναι ε, να διατηρηθεί ο αριθμός των εργαλείων στο ελάχιστο. Πάμε στην πρόταση παριθμών 5 που αφορά στο 2000 14 εδώ αντικατοπτρίζεται, αν θέλετε, αντικατοπτρίζεται η παράγραφη 55-62 και αφορούν στην άποψη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει αποτελεσματική λογοδοσία και διαφάνεια. Αυτό να ισχύει για όλα τα στοιχεία ε, χρηματοδότησης να υπάρχει δημοκρατικός έλεγχος και ως γενικός κανόνας ε, όλοι οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να εντάσσονται μακροπρόθεσμα στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Δεν μπορούμε όλα αυτά να τα κάνουμε εν μια νυχτή. Και επιτρέψτε μου σύντομα να αναφερθώ και στις δικές μας τις αρχές που αναφέρονται τη σελίδα 16 της έκθεσής μας. Εκεί λοιπόν καθίσταται απαραίτητο να υπάρχει μια σαφής ε, ε, λογοδοσία, διαφάνεια, ε, η χρήση των κονδυλίων να προσφέρεται, να προσφέρεται από την ε, διαχείριση. Σας είπα, πλήρης δημοκρατικός έλεγχος έτσι ώστε να μπορούν να υπάρχουν διορθώσεις και βελτιώσεις του συστήματος. Επίσης, μια ισχυρή εντολή για ανεξάρτητο εξωτερικό έλεγχο και πρέπει να υπάρχει και εφαρμογή και παρακολούθηση των συστάσεων περί ελέγχων. Αυτές δηλαδή οι αρχές που αναφέρθηκαν ε, στην αναθεώρηση του 2014. Και τέλος αναφέρομαι στην τελευταία πρόταση η οποία συζητήθηκε συζητήθηκε περισσότερο με την Επιτροπή Ελέγχου ε, αποφασίσαμε να υπάρχει σαφής εντολή ε, δημόσιου ελέγχου. Ε, θεωρούμε ότι θα πρέπει όλοι οι φορείς να καλύπτουν τις δραστηριότητες τους με εξωτερικούς ελέγχους. Και εάν αυτό δεν ισχύει με την τρέχουσα νομοθεσία, θα πρέπει τουλάχιστον να δέχονται την εκπροσώπηση στους φορείς και στα συμβούλια ελέγχου. Γιατί κατά το παρελθόν υπήρξαν κάποια προβλήματα. Και τέλος, αυτή είναι η τελευταία διαφάνεια εκεί προτείνουμε, παρουσιάζουμε όλες μας τις προτάσεις και θέλω να προσθέσω ότι υπάρχει και μια σειρά άλλων εκθέσεων που έχουν δημοσιευτεί ανατομέα, γιατί εδώ βασιστήκαμε στις βασικές αρχές για τον προπλογισμό. Υπάρχει μια έκθεση για το πρασίνισμα. Εκεί δεχτήκαμε κριτική για τους νέους γεωργούς, για τον έλεγχο της αλίας, σημαντική έκθεση για το ρόλο των αρχών πιστοποίησης στην κοινή γεωργική πολιτική άλλη σημαντική πολιτική, πολιτική συνοχή. Εκεί δημοσιεύσα μια έκθεση για το Single Sky, για την ανεργία των νέων, ε, για τα αποθέματα ε, και κάποιες άλλες τομεακές εκθέσεις. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την παρουσίαση της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σε ό,τι αφορά το μελλοντικό προϋπολογισμό της Ένωσης καλό θα ήταν να είναι πιο ε, ξεκάθαροι, να καταλαβαίνουν καλύτερα πώς έχουν τα πράγματα οι Ευρωπαίοι πολίτες και να ξέρουν ποιες είναι οι δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή και στον συνηγητή του ε, πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου για μετά το 2020 και στον εισηγητή και συνηγητή των νέων ιδίων πόρων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω το ελεγκτικό συνέδριο για αυτή την παρουσίαση που αλλάζει λίγο την αντίληψη που έχουν κάποια μέλη του Κοινοβουλίου ότι το ελεκτικό συνέδριο επικεντρώνεται κυρίως στις διαδικασίες και όχι στα αποτελέσματα. Αυτή η έκθεση δείχνει ότι ε, δίνονται πολύ πιο λεπτομερή στοιχεία σε ό,τι αφορά το μέλλον των οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, φράσαμε τη θέση μας στην ε, γνωμοδότηση, κάναμε προτάσεις και περιμένουμε το, την απάντησή σας, η οποία είπατε θα δημοσιευτεί τον Ιούνιο-Ιούλιο. Και τότε θα αντιδράσουμε και πάλι όταν δημοσιευτεί το σχετικό έγγραφο. Καλό θα ήταν να γίνει μια ξεκάθαρη ανταλλαγή ε, πληροφοριών με το ελεγκτικό συνέδριο και υπάρχουν και άλλα στοιχεία που είναι σημαντικά για τη συζήτησή μας σε ό,τι αφορά το μελλοντικό πουδουπού και γενικώ το μέλλον του συστήματος. Γιατί όταν μιλάμε για το πολιτές δημοσιονομικό ε, πλαίσιο πιστεύουμε ότι μιλάμε απλώς για αριθμού, αλλά ουσιαστικά πρόκειται γενικά για το προπολογισμό και το μέλλον του. Και θα ήθελα να υπογραμμίσω κάποια στοιχεία. Πρώτα απ' όλα το θέμα της ε, αξία αξίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχετε δίκιο όταν λέτε ότι δεν πρόκειται για μία ακόμη πρόταση για το ποια είναι η προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ότι πρέπει να υπάρχει μια κοινή αντίληψη. Πρέπει να αποφασίσουμε τι εννοούμε. Το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, η Κομισιόν, γιατί στη συνέχεια... Τι νόημα έχει να συζητάμε συνέχεια για την ε, προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί να έχει ενδιαφέρον, αλλά νομίζω ότι δεν θα αλλάξουν πολλά. Δεύτερον, Υπάρχει κάτι πολύ ενδιαφέρον σε αυτό το έγγραφο. Κάποιοι ε, πολιτικοί στην ε, ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να διαβάσουν το εξή. Παραθέτω, πιστώσαμε την, ε, την ανάγκη συντονισμού των χρηματοδοτικών μέσων Και όσο αυξάνεται η ανάγκη για εγγύησει, τόσο αυξάνονται και οι κίνδυνοι στου οποίου εκτίθεται ο ευρωπαϊκό προπολογισμό. Πολύ συχνά μιλάμε για τι επιπτώσει του τριπλού Α και των αξιολογήσεων, αυτό συζητάμε, αλλά ουσιαστικά αυτό που βλέπουμε εδώ είναι ότι όταν περνάμε στο θέμα των εγγύσεων, τόσο περισσότερο αυξάνονται οι κίνδυνοι και οι επιπτώσεις στον προπολογισμό. Και να είμαι, για να είμαι πιο σαφής, τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι τράπεζα, είναι υπηρεσία, είναι επιχείρηση, είναι δημόσια αρχή. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, θα χρειαστεί να το ξεκαθαρίσουμε στο μέλλον. Γιατί θα περάσουμε σε ένα καινούριο σύστημα, στο πλαίσιο του οποίου εντάξει, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα είναι ακριβώ δημόσια αρχή, θα είναι, λειτουργεί κάπως σαν ε, τράπεζα και θα πρέπει να συζητάμε το θέμα των ε, χρηματοδοτικών εργαλείων. Και αυτό είναι μια απλοποιημένη εκδοχή. Στην πράξη πάντως οι κίνδυνοι αυξάνονται και ε, αντλούμε χρήματα από το δημόσιο κορβανά και ε, πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας αυτό. Είναι πολύ σημαντικό ότι, το ότι τονίζετε αυτό στο εγγραφό σας Χαιρόμαστε που το αναφέρετε. Ο συνάδελφος δεν είναι εδώ. Ε, μιλήσατε για το αποθεματικό. Ο ρόλος των αποθεματικών ποιος είναι. Πρόκειται για ένα ενιαίο αποθεματικό, για διάφορα αποθεματικά. Πρέπει να το σκεφτούμε αυτό. Είναι σημαντικό να υπάρχει ευελιξία. Πώς πρέπει, μπορούμε να φτάσουμε αυτή την απαραίτητη ευελιξία με πολύπλοκα εργαλεία χωρίς να χρησιμοποιούμε αποθεματικά. Πρέπει να επιλέξουμε την απλή ε, λύση και είναι ε, ενδιαφέρον ή ε, έχει ενδιαφέρον η αναφορά στο χρηματοδοτικό σχέδιο. Όχι το δημοσιονομικό σχέδιο, σχέδιο αλλά το χρηματοδοτικό σχέδιο. Νομίζω ότι η Κομισιόν προσπάθησε να ανταποκριθεί. Ε, η, πραγματική πρόκληση είναι οι διορθώσεις. Δεν πιστεύω ότι όλα τα κράτη-μέλη θα ε, συμφωνήσουν με τις διορθώσεις. Θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Και κάτι τελευταίο Ίσως πρόκειται για θέμα διατύπωσης μόνο, αλλά για μένα είναι σημαντικές οι διατυπώσεις, γιατί μιλάτε όχι μόνο για απο, ε, επίτευξη αποτελεσμάτων, αλλά για η επαλήθευσή τους. Αυτό είναι διαφορετικό, γιατί μπορούμε να επιτύχουμε αποτελέσματα και χωρίς να τα επαληθεύσουμε καθόλου, χωρίς να το αποδείξουμε. Και τότε μειώνεται η σημασία της επίτευξης των αποτελεσμάτων ε, την παρουσίασή σας ε, φαίνεται ότι δίνεται σημασία στην απόδειξη των ε, αποτελεσμάτων στους πολίτες, στις κυβερνήσεις. Είναι σημαντικό να επιτευχθούν τα αποτελέσματα, να αξιολογηθούν και στη συνέχεια να επαληθευθούν. Είναι ουσιαστική σημασίας και είναι πολύ ενδιαφέρον που αυτό το αναφέρει το ελεγκτικό σώμα το ότι πρέπει να ε, επαληθεύουμε την επίταξη αποτελεσμάτων. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα ακούσουμε την παρουσίαση ενός από τους δύο συνηγητές ε, των νέων ιδίων πόρων, τον Ζεράρ Ντεπρέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν νομίζω ότι ήδη οι πόροι αποτέλεσαν αντικείμενο μεγάλης προσοχής. Το καταλαβαίνω, γιατί το ελεγκτικό συνέδριο έχει ως ευθύνη κυρίως να συζητάει τον τρόπο με τον οποίο τα οικονομικά μέσα που υπάρχουν στη διάθεσή μας ε, χρησιμοποιούνται. Αν χρησιμοποιούνται σωστά και αν χρησιμοποιούνται με δικαιολογημένο τρόπο. Είδα παρόλα αυτά κάπου να εμφανίζεται όρος ήδη οι πόροι, έτσι. Αλλά ο εκπρόσωπο του ελεκτικού συνεδρίου τους ανέφερε χωρίς όμως να λέει τίποτα. Δεν ξέρω αν έχει σκεφτεί το θέμα αυτό το ελεκτικό συνέδριο. Θα ήθελα λοιπόν να πω δύο-τρία πραγματάκια. Καταρχά, θα ήθελα, αλλά να μην πρόσεξα κιόλα, να μα είχατε δώσει αυτό το έγγραφο πριν από δύο-τρει μήνε, τη στιγμή που ετοιμάζαμε την θέση μα για το μελλοντικό πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Γιατί γίνονται διάφορες ε, προτάσεις από πλευρά σας. Καλό θα ήταν να τις ξέρουμε αυτές τις προτάσεις. Νωρίτερα, και μια και το ελεκτικό συνέδριο είναι ένα σώμα προς υπηρεσία του Κοινοβουλίου, θα είχα εκτιμήσει το να μας είχατε στείλει αυτό το έγγραφο νωρίτερα. Γιατί υπάρχουν κάποιες σκέψεις πολύ έξυπνες, ειδικά για την ευελιξία, για τον τρόπο που θα οργανώσουμε αυτή την ευελιξία σε σχέση με το πώς την οργανώνουμε σήμερα. Αυτό ήταν το πρώτο που ήθελα να πω. Δεύτερον, έχετε μία προσέγγιση όπου λέτε ότι συγκεντρώνουμε τον προπολογισμό της Ένωσης ε, στους τομείς όπου υπάρχει μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία. Αλλά δεν την ορίζετε την προστιθέμενη αξία. Λέτε, εάν διάβασα καλά, ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας διαθεσμικός ορισμός της προστιθέμενης αξίας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συγκρίνουμε τα προγράμματα και μετά να δικαιολογήσουμε την κατανομή των πόρων. Αν είναι αλήθεια, ε, ας το φτιάξουμε αυτόν τον ορισμό. Γιατί το να επικαλούμαστε την ευρωπαϊκή ε, προστιθέμενη αξία αν δεν μπορούμε να την ορίσουμε. Και αν δεν συμφωνούμε τα διάφορα θεσμικά όργανα για το ποια είναι αυτή η περίφημη προστιθέμενη αξία, ε, χωρίς συγκεκριμένες παραμέτρους, τι νόημα έχει. Είναι απλώς ρητορία είναι σχήματα, ας πούμε, ε, απλώς ε, ρητορικά. Όταν μιλάτε για την ευρωπαϊκή προσθεμένη, ε, νοσιακή δηλαδή προσθεμένη αξία, στην πράξη τι σημαίνει, στο βαθμό που δεν έχουμε έναν ορισμό. Παραδείγματο χάρη για την πολιτική συνοχή. Τι είναι αυτή η ευρωπαϊκή προσθεμένη αξία. Εγώ το ξέρω ότι υπάρχει μια τέτοια ευρωπαϊκή προσθεμένη αξία, γιατί έχω το δικό μου ορισμό, τον προσωπικό ορισμό μου για την ευρωπαϊκή προσθεμένη αξία. Αλλά εσεί όταν μιλάτε για αυτή την έννοια, σε τι αντιστοιχεί. Ούτε για την ΚΑΠ, για την κοινή αγρο... Ε, ε, συγγνώμη, γεωργική πολιτική. Ποια είναι η ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία. Εντάξει, καλή είναι αυτή η ρητορία, αλλά δεν υπάρχει κοινά αποδεκτός ορισμός. Και πώς με βάση αυτό το έγγραφό σας μπορούμε να περάσουμε από τις συστάσεις σας σε κάτι πιο πρακτικό. Έτσι. Εσείς συστήνετε κάποια πράγματα απλώς, αλλά τίποτε άλλο. Υπάρχουν πάρα πολλές συστάσεις που θα ήθελα να τις συζητήσουμε. Παραδείγματος χάρη, μιλάτε για κάτι πολύ εντυπωσιακό. Μιλάτε για τη διάρκεια του πουδουπού και εφιστάτε την προσοχή στο εξή. Αν διαρκέσει το πουδουπού 7 χρόνια, θα πρέπει να θεωρήσουμε, να εξετάσουμε τις συνέπειες που έχει αυτό το πουδουπού 13 χρόνια μετά, λόγω της καθυστερημένης ε, πληρωμής ε, κάποιων προγραμμάτων, γενικά της καθυστέρησης των πληρωμών. Και όταν διαπραγματευόμαστε λοιπόν το πουδουπού, θα πρέπει να σκεφτόμαστε και τι θα συμβεί αργότερα, αύριο μεθαύριο, 13 χρόνια μετά, για να αποφύγουμε τις δραματικές καταστάσεις που αντιμετωπίσαμε πρόσφατα. Επομένως, μου άρεσαν οι γενικοί προσανατολισμοί που προτείνεται, αλλά έτσι όπως έχουν τα πράγματα, δεν έχουμε αρκετά στοιχεία στα χέρια μας στο βαθμό και μάλιστα δεν έχουμε μια αφετηρία κοινή, δηλαδή αυτή την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Δεν την ορίζουμε για να ε, ορίσουμε με αντικειμενικό τρόπο τους, ε, τις προτεραιότητες πάνω στις οποίες θα εστιαστεί ο προϋπολογισμός της Ένωσης και επίσης τα κριτήρια για να εκτιμήσουμε μετά τον τρόπο με τον οποίο δαπανώμε τα κονδύλια. Ευχαριστώ. Ακούσαμε τους δύο συνεισηγητές που είναι παρόντες. Η κυρία Γκουάρντια Θαβάλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, να ευχαριστήσω το ενεκτικό συνέδριο που μας ετοίμασε αυτή την ε, έκθεση και ευχαριστώ και τον κύριο Ντεπρέ για αυτά που είπε. Ο καλό θα ήταν, ε, σωστό είναι αυτό που είπε, ότι θα έπρεπε να το είχαμε αυτό το κείμενο νωρίτερα όταν κάναμε τις, τις συζητήσεις για το ΠΟΥΔΟΥΠΟΥ και το... τους ίδιους σπόρους. Εν πάση περιπτώσει, εδώ φτάσαμε ε, και στις μελλοντικέ μας διαπραγματεύσεις θα λάβουμε υπόψη το κείμενό σας. Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι γενικά συμμερίζομαι την ανάλυση και τα αποτελέσματα της έκθεσής σας. Αλλά έχω δύο προβλήματα. Πρώτον, στην πρώτη φάση, στον, στον καθορισμό των προτεραιοτήτων. Έτσι. Και αυτή είναι η πρώτη φάση, όπως λέει και το ελεκτικό συνέδριο, και στη δεύτερη φάση βάζουμε τα λεφτά. Αυτό το, το ζητάει το Κοινοβούλιο να το, να το κάνουμε, αυτέ τι δύο φάσει, αλλά δεν το θέλει το Συμβούλιο. Είναι πολύ σημαντικό για να έχουμε αυτή την ευελιξία και αυτά τα περιθέρια. Γιατί το ε, Συμβούλιο βάζει ένα όριο και επ' αυτού εμεί πρέπει να φτιάξουμε τι προτεραιότητε. Αυτό το όριο, αν είναι πολύ κάτω, έτσι πολύ χαμηλό, τελικά Απλώς πρέπει να χρησιμοποιούμε αυτό το 100% των ε, χρημάτων αυτών για να χρηματοδοτήσουμε τις προτεραιότητες που έχουμε. Και δεν έχουμε κανένα περιθώριο ε, για μελλοντικέ απρόβλεπτες καταστάσεις. Αν η συζήτηση γινόταν αλλιώ, να λέγαμε να οι προτεραιότητες και να τα λεφτά και έχουμε και κάποια στην πάντα ας πούμε για τα απρόβλεπτα θα ήταν πολύ καλύτερα. Τώρα, για την προσθέμενη αξία, να κάνω κι εγώ κανένα σχόλιο, συμφωνώ καταρχά με αυτά που άκουσα. Η προσθέμενη αξία είναι η ατέρμονη συζήτηση ποτέ δεν συμφωνούμε, ποτέ δεν έχουμε ένα ξεκάθαρο ορισμό. Δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να συμφωνήσουμε πάνω σε έναν ορισμό, γιατί η έννοια της προσθέμενης αξίας έχει πολλές ερμηνεύεται με διαφορετικού τρόπου. Υπάρχουν διάφορες απόψεις και τα κριτήρια που χρησιμοποιεί ο καθένα είναι τελείως διαφορετικά. Γι' αυτό μου φαίνεται επικίνδυνο να λέμε ότι ο, ο ενωσιακό προπολογισμό θα πρέπει να επικεντρώνεται σε εκείνα τα προγράμματα που έχουν υψηλή προστιθέμενη αξία. Είναι επικίνδυνο. Γιατί? Γιατί ανάλογα με τα κριτήρια, όταν κοιτάξουμε τον προπολογισμό με αυτή την υψηλή υποτίθεται προστιθέμενη αξία, με τον ορισμό που υπάρχει, ο, τότε ο σημερινό ε, ενωσιακό προπολογισμό είναι εκτό τόπου και χρόνου. Έτσι. Ο προπολογισμό όμω τη Ένωση ορίζει και την ουσία τη Ένωση. Γι' αυτό διαρωτώ με, ποιο είναι Ποιος να ποια είναι αυτή η προστιθέμενη αξία. Τελικά θα οδηγηθούμε σε μια φιλοσοφική συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα φτάσουμε ποτέ σε συγκεκριμένους δείχτες για να καθορίσουμε τον προϋπολογισμό για τα επόμενα χρόνια. Γιατί υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου γίνεται μια πολιτική χειρονομία ή θέλουμε να περάσουμε ένα πολιτικό μήνυμα κτλ. που δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να οριστεί με όρους προσθέμενης αξίας. Επομένω, ενδιαφέρουσα θα ήταν μια τέτοια συζήτηση για την προστιθέμενη αξία, αλλά είναι πολύ επικίνδυνο να κλείσουμε τη συζήτηση, να την κλειδώσουμε γύρω από την προστιθέμενη αξία και να μην πούμε τίποτα άλλο. Κάτι άλλο τώρα, ένα άλλο σχόλιο. Τα προβλήματα που είχαμε τι πληρωμέ. Ο κύριο Ντεπρέ εδώ είπε ότι οι πληρωμέ κάνουν ένα ε, πάνω κάτω ας πούμε. Πότε δίνουμε πολλά, πότε δίνουμε, λίγα, πότε δίνουμε λίγα λεφτά και θα πρέπει στο μέλλον κάπως να τις εξομαλύνουμε ας πούμε. Η εύκολη λύση θα ήταν να βάλουμε ένα υψηλό επίπεδο επαρκές ας πούμε για να σταματήσουμε με αυτή την ιστορία πάνω κάτω, πάνω κάτω οι πληρωμές. Ε, αλλά όμως ξέρετε ότι η πραγματικότητα δεν είναι έτσι και ε, με το Συμβούλιο διαπραγματευόμαστε και είναι πολύ δύσκολο να φτάσουμε σε αυτό το ιδανικό επίπεδο πληρωμών. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε ένα σύστημα αποθεματικού πληρωμών για εκείνες, τις πληρωμέ, για εκείνες τις περιπτώσεις που δεν χρησιμοποίησαμε όλα τα λεφτά και μπορούμε να πάρουμε ένα τμήμα και να τα βάλουμε σε ένα αποθεματικό για να τα χρησιμοποιήσουμε στο μέλλον. Για να αντιμετωπίσουμε μελλοντικέ ας πούμε πληρωμές για να μην καυγαδίζουμε μονίμως ας πούμε για το θέμα των πληρωμών. Ευχαριστώ. Merci. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Διστόφσκι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω στα τσέχικα, είναι καλύτερα. Μια και είμαι τσέχος. Θα ήθελα να ε, σας ευχαριστήσω για την παρουσίαση αυτού του ε, πλήρους και λεπτομερούς εγγράφου. Πράγματι αυτό το έγγραφο θα έπρεπε να το είχαμε λάβει νωρίτερα, αλλά είναι άλλο θέμα αυτό. Μιλάμε συχνά για την προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς στην Ελεγκτική Επιτροπή μιλάμε για τις επιπτώσεις του χρήματος που χρησιμοποιείται και για την ανάγκη ότι πρέπει να ελέγχουμε πού χρησιμοποιούνται τα χρήματα. Αυτό που είπε ο κύριος Όλμπριχτ, καμιά φορά το δεξί χέρι δεν ξέρει τι κάνει το αριστερό εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς διαθέτουμε χρήματα από διάφορα ταμεία για το ίδιο πράγμα. Στο τομέα της ε, γεωργίας, για παραδείγματος χάρη, από τη μία αντιμετωπίζουμε την κλιματική αλλαγή και από την άλλη ε, επενδύουμε στην αντικοποίηση της γεωργίας. Και νομίζω ότι εδώ εντοπίζεται η προστιθέμενη αξία και πρέπει να έχει ε, ουσιαστικό ρόλο στον επόμενο προϋπολογισμό Πρέπει να μιλάμε λοιπόν για τις επιπτώσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ε, λειτουργήσει ως ε, τράπεζα ή ως χρηματοδοτικός οργανισμός πώς θα πρέπει να διατεθούν ε, τα χρήματα σε πολυεθνικές, ε, σε μεγάλες επιχειρήσεις. Πρόκειται για την κινητήρια δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν πρέπει να επενδύσουμε 100 εκατομμύρια για ε, καλύτερο ψωμί, για καινοτομία. Το είπατε πολύ σωστά στη τελευταία διαφάνεια. Τα δύο επόμενα χρόνια θα είναι πολύ σημαντικά για να μας δοθούν διευκρινήσεις σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις, οι οποίες δεν αφορούν μόνο τους ίδιους πόρους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να εξαρτάται μόνο από τις ε, εισφορές των κρατών μέλων. Ε, στην Τσεχία ε, πάντα ακούγονται επικρίσεις. Εμείς πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ένα εξάρτητο σύστημα πόρων, που θα χρηματοδοτεί την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι πολύ καλό το έγγραφό σας και θα ήταν σημαντικό να ενισχύσουμε επιπλέον το σχετικό ε, κεφάλαιο για τη χρηματοδότηση, προκειμένου αυτό το έγγραφο τους επόμενους μήνες να μας επιτρέψει να ξανασυζητήσουμε αυτά τα θέματα. η κυρία Κρέσλε. Πάρα πολύ καλό το έγγραφο και ποτέ δεν είναι αργά. Άρα δηλαδή είναι σημαντικό η Επιτροπή Προϋπολογισμών ε, να αποφασίσει να κλείσει τα κενά που υπάρχουν στη λογοδοσία και να προσπαθήσει να ασκήσει επιρροή σε όλα τα κονδύλια τα οποία διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει το EDF να ενταχθεί στον προεπολισμό, το αναπτυξιακό δηλαδή ταμείο. Ε, δεν πρέπει να αφήσουμε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Και μετά η συζήτηση και για το νομισματικό ταμείο. Είναι σαφές ότι πρέπει να μπορεί να τοποθετείται το ελεγκτικό συνέδριο. Και μετά υπάρχουν άλλοι οργανισμοί που δεν ξέρουμε τίποτα. Παραδείγματο χάρη οργανισμός άμυνας. Ε, πολλοί είπαν ότι ε, η Επιτροπή Προπολογισμών πρέπει να επιληφθεί αυτού του θέματο γιατί χωρίς στην Επιτροπή Προπολογισμών δεν μπορεί κανεί να λειτουργήσει ούτε τον, του ελέγχου προπολογισμών ούτε οποιοδήποτε άλλο. Γι' αυτό λοιπόν ε, θεωρώ ότι υπάρχουν ε, κάποια ε, κομμάτια τα οποία δεν εντάσσονται στον νοσιακό προπολογισμό, είναι όμως πολύ σημαντικά. Άρα πρέπει να έχουμε ως ελεγκτή το ελεγκτικό συνέδριο και με τον τρόπο αυτό να μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα θέματα τα οποία δεν μπορούμε να επηρεάσουμε άμεσα. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να δούμε λιγάκι την σύσταση υπαριθμών 6 και Επιτροπή Προπολογισμού να επιληφθεί αυτή αυτής της ε, σύστασης της επαριθμών 6. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Και κάτι άλλο. Βρισκόμαστε κάτω υπό φοβερή πίεση. Εμείς ε, ως Επιτροπή Ελέγχου Ευρωπλογισμών όλο το χρόνο ασχολούμαστε με προγράμματα τα οποία μας τελικά δεν επιτυγχάνουν το στόχο τους. Υπήρξαν δύο τραγικοί έλεγχοι στον τομέα της Γεωργίας όσον αφορά το πρασίνισμα. Εκεί αναφερόταν 12 ε, δις κάθε χρόνο για το τίποτα και ε, επίσης και σε ένα άλλο πρόγραμμα 18 δις και εκεί δεν επιτεύχθηκε ο στόχος. Και πολλοί λένε τι να κάνουμε, έτσι έχουν τα πράγματα. Εγώ δεν είμαι κατά του να παρέχετε στήριξη, αλλά να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε με προγράμματα που πραγματικά δεν αποδίδουν. Νομίζω ότι και εδώ στο Κοινοβούλιο θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ε, κλείσουμε, να ε, καταργήσουμε κάποια προγράμματα. Αυτό επιτρέπεται από τον κανονισμό. Όσον αφορά τώρα τα χρηματοδοτικά εργαλεία, είμαι πολύ επικριτική από αυτού, γιατί εκεί ε, προβλέπονται πάρα πολλά μοντέλα χρηματοδότησης που δεν ξέρει ούτε το ελεγκτικό συνέδριο, ούτε εμείς τι ακριβώς γίνεται. Και κατόπιν υπάρχει και ένα άλλο βασικό ερώτημα για τα ραλ, τα ραλ αυτά, τα, αυτά που υπολείπονται και μεταφέρονται αυτά που υπολείπονται προς εκαθάριση. Ε, νομίζω ότι αυτά είναι ένα θέμα που πρέπει να το εξετάσουμε, να δούμε τι θα κάνουμε με το θέμα αυτό. Ε, ε, ευχαριστώ, πολύ για την παρουσίαση. Εγώ βασικά θέλω να ρωτήσω σχετικά με την ε, προστιθέμενη αξία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και για μένα αυτό που έχει επίσης ε, σημασία είναι το να ενισχυθεί το πλαίσιο απόδοσης. Εσείς έχετε καταθέσει συστάσεις ε, για να ενισχυθεί αυτό το πλαίσιο. Μία πρόταση είναι να συμμορφωθεί ο προγραμματισμός με τις στρατηγικές προτεραιότητες. Εγώ βέβαια πάντα σκέπτομαι ότι τώρα είμαστε στη διαδικασία προετοιμασίας του επόμενου πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου, αλλά δεν έχουμε την Ευρώπη 2030, δεν έχουμε δηλαδή το σαφές στρατηγικό έγγραφο και ως εκ τούτου θα πρέπει ε, το, το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και τον προϋπολογισμό μας να τα συνδέσουμε με αυτό το συγκεκριμένο έγγραφο. Ίσως πρέπει αυτά να τα προετοιμάσουμε παράλληλα και κατόπιν βέβαια με αυτή τη στρατική θα πρέπει να συζητήσουμε και την ε, προστιθέμενη αξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι πρέπει να γίνει έτσι ώστε να δημιουργήσουμε περισσότερες συνέργειες με τους εθνικούς προϋπολογισμούς γιατί με τον μικρό ενωσιακό προϋπολογισμό δεν μπορούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη επιρροή να μπορούμε να ασκούμε στους εθνικούς προϋπολογισμούς και με ενδιαφέρει και αυτό το τρίτο σημείο ε, το οποίο εσείς έχετε συμπεριλάβει στην διαφάνειά σας εκεί που ορίζεται την προστιθέμενη αξία. Πρόκειται για τις αιτήσιες αναφορές σχετικά με το ε, καθαρό προϋπολογισμό Δηλαδή η δική σας η άποψη είναι να συνδυαστούν αυτά με αναλύσεις ε, χρηματοδοτικών και μη χρηματοδοτικών ε, πλεονεκτημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί αυτή τη στιγμή αναλύουμε απλά το κόστος και το όφελος ε, και το τι εισέρχεται και τι εξέρχεται στον Ευρωπαϊκό Ευρωπολογισμό, το αποτέλεσμα εδώ όμως ποια είναι ακριβώς η ιδέα, τι πρέπει να προσθεθεί. Ίσως ε, το όφελος από την ε, ενίσχυση της νέας αγοράς και μετά μπορούμε να δούμε την ε, πυροή που η πολιτική συνοχής η οποία ενισχύει την κοινή αγορά και από αυτό ε, εποφελούνται κυρίως οι καθαροί συνεισφορείς στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Νομίζω ότι αυτό θα ε, βοηθήσει έτσι ώστε να υπάρξει μεγαλύτερο πλεονέκτημα από τον ενωσιακό προϋπολογισμό. Το τελευταίο που θέλω να πω έχει σχέση με το δημοσιονομικό σχέδιο, τον σχεδιασμό που προτείνεται Νομίζω ότι αυτό είναι απολύτως απαραίτητο, γιατί κάθε φορά υπάρχει αυτό το πρόβλημα ανάμεσα σε αυτό που προγραμματίζεται ανάμεσα σε αυτό που καταβάλλεται, προκύπτουν καθυστερήσεις στις πληρωμές. Ως εκ τούτου ε, χρειαζόμαστε και καλύτερη επικοινωνία με τα κράτη-μέλη. Πρέπει λοιπόν να ε, προβλεφθεί ένα ειδικό σύστημα ελέγχου ε, ηλεκτρονικό για να μπορούμε να ελέγχουμε σε επίπεδο κρατών μελών το τι γίνεται και μετά να γίνεται καλύτερος προγραμματισμός του ενωσιακού προϋπολογισμού. Ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω κάποιος άλλος να θέλει να λάβει το λόγο. Αν μου επιτρέπετε λοιπόν, θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια προσωπικά. Πρώτα απ' όλα για να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο για αυτή την παρουσίαση. Σημείωσα ότι δεν πρόκειται για οριστικό και ε, δουλειά για οριστικό έγγραφο. Πρόκειται για ενημερωτικό έγγραφο. Πολύπονται λοιπόν κάποιες εβδομάδες, κάποιοι μήνες για να προχωρήσουμε. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα ουσιαστικό ζήτημα το οποίο μας απασχολεί θα χρειαστούν σίγουρα και άλλες συναντήσεις με το ελεγκτικό συνέδριο για να ξεκαθαρίσουμε ε, ποιο θα είναι το όραμά μας, ποιες θα είναι οι πρακτικές που θα ακολουθούμε ως προς τον ε, προϋπολογισμό, γιατί ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Δεν τηρεί το θέμα, την αρχή της ε, ε, δημοσιονομικής ενότητες και επειδή δεν υπάρχει ευελιξία πρέπει να εφεύρουμε εργαλεία. Όταν, ε, επειδή δεν έχουμε ε, πόρους πρέπει να εφευρίσκουμε καινούρια εργαλεία με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα. Στην αρχή υπάρχουν, υπάρχει θετικός αντίκτυπος αλλά υπάρχουν κίνδυνοι κάποια στιγμή θα χρειαστεί να αναγνωρίσουμε απώλειες, ζημίες, οι οποίες θα έχουν επιπτώσεις στον προϋπολογισμό. Πώς μπορούμε λοιπόν να ξεφύγουμε από αυτό το δημοσιονομικό κατακαιρματισμό που δεν τον καθιστά και δεν καθιστά τον ε, το προϋπολογισμό καθόλου ευανάγνωστο ούτε από το Κοινοβούλιο ούτε από τους ε, πολίτες. Δεν τηρείται η δημοσιονομική οικουμενικότητα. Θα έπρεπε να εμφανίζονται όλες οι δαπάνες και όλα τα έσοδα το πρωί το είπαμε όταν μιλάμε για το Brexit. Μάλλον θα χάσουμε 14 ε, δισεκατομμύρια γιατί το Ηνωμένο Βασίλειο είναι καθαρός ε, συνεισφορέας αλλά άμα συναυθούν συμφωνίες όπως με την ε, Νορβηγία και την Ελβετία θα δημιουργηθούν οι πόροι. Και τώρα κοιτάμε τον ευρωπαϊκό προπολογισμό και αναρωτιόμαστε ποιοι θα είναι αυτοί οι πόροι γιατί δεν εμφανίζονται. Γιατί θα απευθείας σε χώρες που αποφελούνται από την πολιτική ε, συνοχή. Εσείς στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο θα έπρεπε να καταγγείλετε αυτές τις πρακτικές. Αν ε, αύριο μεθαύριο το Ηνωμένο Βασίλειο καταβάλει 4, 5, 6 δισεκατομμύρια στα πλαίσια συμφωνίας όπως αυτή που έχει συναυθεί με τη Νορβηγία και την Ελβετία, αυτό σημαίνει ότι δεν θα εμφανίζονται αυτά τα ποσά στο προπολογισμό. Με εκπλήσει το ότι δεν κάνετε καμία αναφορά σε αυτό. Πώς μπορούμε να έχουμε έναν προπολογισμό δεν λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές δαπάνες, τα πραγματικά έσοδα. Διαθέτουμε 3 δισεκατομμύρια για το μηχανισμό για την Τουρκία που θα έπρεπε να, νομίζετε, θα έπρεπε να ονομάζεται μηχανισμό στήριξη για τους ε, Σύρους πρόσφυγες και στην πράξη φαίνονται μόνο 2 ε, δισεκατομμύρια. Στην ε, έκθεσή σας καλό θα ήταν να ε, κάνετε κάποιες παρατηρήσεις σχετικά με αυτές τις ιδιωτηριότητες προκειμένου ο προϋπολογισμός να είναι πιο ευαγανάγνωστος, πιο ξεκάθαρος σχετικά με τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μιλήσατε και για την προστιθέμενη αξία. Μπορούμε να ξεφύγουμε από τον ορισμό των κοινών ευρωπαϊκών αγαθών. Γιατί βλέπουμε με την ε, παγκοσμιοποίηση ότι υπάρχουν ε, κάποια κοινά αγαθά. Σε κάποιες περιπτώσεις η προστιθέμενη αξία δεν θα είναι να μεταφερθεί η στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κάποια κονδύλια να περάσουν από, τα εθνικά, από τους εθνικούς προϋπολογισμούς στο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό θα αποδεικνύει ποια είναι η προστιθέμενη αξία. Αν δεν είναι αποτελεσματικές οι δαπάνε σε ορισμένους τομείς σε εθνικό επίπεδο, ενώ αν η διαχείριση γινόταν σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα ήταν πολύ πιο εύκολο να αποδειχτεί η προστιθέμενη αξία της ευρωπαϊκής ε, ε, αξίας. Πρέπει να οριστεί αυτή η προστιθέμενη αξία αξία. Υπάρχει προσθέμενη αξία, για παράδειγμα, στα ταμεία συνοχή, αφού βασίζονται στην αλληλεγγύη, προκειμένου να αναπτυχθούν κάποιες ε, περιφέρειες. Ε, για τα υπόλοιπα όμως ε, είναι θέμα κοινή διαχείριση, διαχείριση από κοινού. Όλα όσα υπόθηκαν ήταν πολύ ενδιαφέροντα είπατε ότι καλό θα ήταν να υπάρχει ε, συμπληρωματικό ε, οικονομικό σχέδιο ε, που να συμπληρώνει το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Φυσικά υπάρχει, χρειάζεται προβλεψιμότητα για τις επενδύσεις. Δεν θα είχε ενδιαφέρον να υπάρχει κάθε χρόνο να γίνονται συζητήσεις για το ποιες θα μπορούσαν να είναι οι απρόβλεπτες καταστάσεις, οι έκτακτες ανάγκες. Καλό θα ήταν να ξανασυναντηθούμε τις επόμενες εβδομάδες προκειμένου να συζητήσουμε τι θα μπορεί να είναι ακριβώς ε, ο προϋπολογισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης, να, να έχουμε ένα πιο κριτικό ε, βλέμμα. Είναι πάντως επίγον το δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανακτήσει το ρόλο που του αναλογεί και να τηρεί κάποιες αρχές, τίσια βάση ε, ε, και διαφάνεια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να ε, προσθέσει κάτι σχετικά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα Θα ήθελα να ευχαριστήσω την, ε, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο για αυτή την ε, παρουσίαση, μιας και αυτή τη στιγμή προετοιμάζουμε την πρόταση που θα υποβάλουμε τον Μάιο. Υπάρχουν κάποιοι τομείς στους οποίους υπάρχει κοινή προσέγγιση με την ε, Επιτροπή σε ό,τι αφορά το πολιτές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο, σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια, την απλοποίηση, ε, τη λογοδοσία είναι βασικές αρχές για την προετοιμασία του επόμενου πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου. Εγώ θα ήθελα να εστιάσω σε τρία βασικά ζητήματα που αναφέρθηκαν. Πρώτον, η προστιθέμενη αξία για την ε, Κομισιόν, όπως έχει επαναληφθεί, αυτή η έννοια είναι δύσκολο να οριστεί, πρέπει να αναλυθεί, να εξεταστεί βάσει πολλών στοιχείων ε, αποτελεσματικότητας, εξορθολογισμού, συνεργειών και εξυγχρονισμού των προγραμμάτων θα μπορούσε να είναι δύσκολο κατά τη γνώμη μας, θα ήταν δύσκολο να συναυθεί συμφωνία, να συμφωνήσουμε για ένα κοινό ορισμό, καλύτερο θα ήταν να έχουμε μια κοινή αντίληψη της έννοιας της προστιθέμενης αξίας, χωρίς όμως η προστιθέμενη αξία να είναι ένας ε, μαθηματικός τύπος. Ναι, αυτό είναι η προστιθέμενη αξία. Μπορείς να υλοποιείς αυτό το πρόγραμμα, αλλά όχι το άλλο. Το δεύτερο που θα ήθελα να πω είναι οι μακροπρόθεσμες προβλέψεις εσόδων και εξόδων. Η διασφάλιση των πληρωμών και ο έλεγχός τους είναι κοινή στόχη. Θα θέλαμε στην πρότασή μας σχετικά με το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο να δώσουμε ε, όσα περισσότερα στοιχεία γίνεται από αυτά που έχει προτείνει το ελεγκτικό συνέδριο. Υπάρχει ένα νέο άρθρο, το άρθρο 247, που προβλέπει μια νέα ενημέρωση σχετικά με τις μελλοντικές προβλέψεις εσόδων και εξόδων. Θα λάβουμε υπόψη μας ε, ε, τους κινδύνους που απορρέουν από τις εγγυήσεις και τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Θα ήθελα όμως να τονίσω πάντως ότι αυτή τη στιγμή όλα οι λεπτομέρειες ε, συμπεριλαμβάνονται στην, ε, στην έκθεση της Επιτροπής. Και το τελευταίο που θα ήθελα να πω είναι το πλαίσιο απόδοσης. Συμφωνούμε με το ηλεκτρικό συνέδριο ότι πρέπει να απλοποιήσουμε αυτό το πλαίσιο που χρησιμοποιούμε. Είναι σημαντικό να εντοπίσουμε τις πραγματικές προτεραιότητες προκειμένου να επιτευχθούν οι στόφοι και να εντοπίσουμε τους βασικούς δείκτες που θα επιτρέψουν την Κομισιόν να εξηγήσει πώς ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμβάλλει στην ε, ε, ανταπόκριση σε αυτές τις προτεραιότητες. Είναι δύσκολο το θέμα φυσικά, ε, μιας και έχουμε 700 δείκτες. Αρκεί να σας το πω αυτό για να καταλάβετε. Το, το θέμα δεν είναι καθόλου εύκολο. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά ήθελα να σας πω κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Κύριε Γκρέγκορ. Μπορούμε να τελειώσουμε. Στις 12.30 δεν γίνεται. Έχουμε πρόβλημα με τους διερμηνείς όμως. Μπορείτε να είσαστε συντομότατος, ούτω ώστε να μπορέσουμε να σας ξαναφέρουμε εδώ. Γιατί δεν μπορούμε να μείνουμε σε αυτήν την κατάσταση. Θα πρέπει κάπου να καταλήξουμε σε κάποιες συστάσεις. Διεξοδικές χωρίς να υποτιμούμε την ανάγκη ε, και κριτικής αλλά και σωστής διάγνωσης. Uh, uh, Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Θα προσπαθήσω να εστιάσω σε οριζόντια θέματα τα οποία αναφέρθηκαν αρκετές φορές. Φυσικά μπορούμε να ξανάρθουμε στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού και στην Επιτροπή Προπολογισμών όποτε θέλετε ή και στις δυο μαζί και θα προσπαθήσα, προσπαθήσαμε να χωρίσουμε τα ενημερωτικά έγγραφα σε δύο για να ακούσουμε και ερωτήσεις και να απαντήσουμε. Στη δεύτερη φάση έχουμε πλέον ευκαιρίες για ερωτήσεις και απαντήσεις. Λοιπόν, για το πλαίσιο επιδόσεων και την προσθέμενη αξία. Είναι ένα τομέα όπου είναι εύκολο σχεδόν κανεί να, κάνει, να δίνει συστάσει, αλλά σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του στι τομεακέ πολιτικέ, γιατί και το πράγμα δυσκολεύει. Δεν λέμε ότι ο μη σεβασμός ή ο χαμηλότερο σεβασμός της, ε, της προστιθέμενης αξίας αυτό σημαίνει ντε και καλά περικοπές στον προϋπολογισμό. Δεν λέμε κάτι τέτοιο, έτσι. Ο ενωσιακός προϋπολογισμός θα πρέπει να παραμείνει ένας αναδιανεμητικός προϋπολογισμός στο μέλλον, σε κάποιο βαθμό. Αλλά παράλληλα οι πολιτικές να ε, εστιάσουν περισσότερο σε δείκτες και σε αποτελέσματα. Συμφωνώ με αυτούς που λένε ότι είναι δύσκολο να ορίσουμε την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Προς το παρόν, λοιπόν, χρησιμοποιούμε τον ορισμό της Κομισιόν, που παρουσιάστηκε επίσης και υπάρχει και στο έγγραφο προβληματισμού. Ε, αυτό σημαίνει ότι μερικές φορές μπορεί να έχουμε διαφοροποιημένη συγχρηματοδότηση και να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να συνεισφέρουν περισσότερο σε διαδικασίες και πολιτικές που έχουν λιγότερη προσθέμενη αξία. Να ένας τρόπος να το κάνουμε, ας πούμε. Για την ευελιξία και το οικονομικό σχέδιο, είναι σημαντικό όλες οι προφορίες που θα έχουμε για τους πόρους εκτός του προϋπολογισμού να είναι διαθέσιμες στην διαδικασία προϋπολογισμού. Μου αρέσει η παράφραση 73 της θέσης του Κοινοβουλίου. Για τη δική μας ε, εντολή θα ήθελα να λάβουμε στήριξη από το Κοινοβούλιο, γιατί είναι πολύ σημαντική αυτή η στήριξή σας και να μπορέσουμε να ελέγχουμε όχι μόνο τα, τις δαπάνες του προπολογισμού, αλλά μαζί με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, όσο περισσότερα πράγματα ε, χρηματοδοτούμε ε, και εκτός προπολογισμού, τόσο πιο σημαντικό είναι ο συντονισμό. Παραδείγματο χάρη ε, ναυτιλιακέ μεταφορέ, όπου χρηματοδοτούσαμε και από τον προπολογισμό και εκτό προπολογισμού. Και συγχρηματοδοτούσαμε και η ΜΕΝ και η ΔΕ και δεν λειτουργούσε το πράγμα καθόλου. Για τι ευελιξίε και τι πληρωμέ, θέμα που αναφέρθηκε, συμφωνούμε με το Κοινοβούλιο ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν όρια στι μεταφορέ ε, πιστώσεων από χρόνο σε χρόνο σε χρόνο που δεν χρησιμοποιήθηκαν προς ε, τα επόμενα έτη που μπορεί να χρησιμοποιηθούν. Ελπίζω να αλλάξει αυτό. Για τους ίδιους πόρους είδα ότι η θέση μας ε, από το 1999 μέχρι το 2005 και από το 2005 μέχρι το 2012 είναι συγχρονισμένη με του Κοινοβουλίου. Προς την ίδια κατεύθυνση κινούμαστε. Στην τελευταία γνωμοδότηση του 2012 είχαμε παρατηρήσει ότι οι διπόροι που βασίζονται στο ΦΠΑ είναι περίπλοκοι και η σχέση μεταξύ του ποσοστού ε, ε, ε είναι πρόβλημα και επίσης θα πρέπει να μειώσουμε τις εισφορές από τους ρεωνιακούς δασμούς ε, ε, ιδίως για το κεφάλαιο 5 στο οποίο δουλεύω πολύ πρόσφατα είδαμε ειδικά λόγω του Brexit, ότι η διαχείριση των οικονομικών κινδύνων στους παραδοσιακούς ίδιους πόρους, του ΣΤΟΡ, ε, θα είναι αντικείμενο και των επομένων ελέγχων μας. Θα σταματήσω και θα, πω, θα σας πω τα υπόλοιπα σε άλλη <laughs> φορά, σε άλλη φάση. Να προσθέσουμε και μια άλλη αρχή, την αρνητική προσθέμενη αξία. Μερικές φορές η ανεπάρκεια της Ευρώπης κοστίζει χρήμα ειδικά σε ό,τι αφορά τη φορολογική απάτη, ε, τη, την απάτη του ΦΠΑ. Θα μπορούσατε να μιλήσατε λοιπόν και την αρνητική προσθεμένη αξία στην έκθεσή σας, όταν υπάρχει μια ανεπάρκεια της Ευρώπης. Για να τονίσουμε την ανάγκη για Ευρώπη. Bien, nous allons rester là, mes chers collègues. Θα σταματήσουμε εδώ. Ε, ξαναρχίζουμε στις 2.30, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι οι νέε ε, διατάξεις ε, που έχουμε και τα ωράρια. Μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στα πλαίσια ενό εργαστηρίου που αφορά την ε, δημοσιονομική ικανότητα της Ευρωζώνης.